Good afternoon, colleagues. We are starting the meeting of our committee. As we understand, the last working week Γεια σας, συνάδελφοι. Είναι η τελευταία συνεδρίαση πριν το καλοκαίρι και βλέπετε ότι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλος ε, ενθουσιασμός. Ε, προτείνω τις εξής αλλαγές στην ε, ημερήσια διάταξη. Σημείο 17, διαρθρωμένος διάλογος με τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, Επίτροπο για ζητήματα μετανάστευσης εσωτερικών υποθέσεων Δυστυχώ πρέπει να αναβληθεί καθώς είχε ανηλυμένε υποχρεώσεις. Σημείο 15. Ψηφοφορία για την απελευθέρωση των θεωρήσεων για το Κόσοβο. Εισηγητή ο κύριο Φαγιών. Δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Καθώς η αξιολόγηση από πλευράς κομισιών για κάποιους συγκριτικούς δέκτε δεν έχει ακόμα παραληφθεί από τον εισηγητή. Υπάρχουν ε, ενστάσεις για την ημερήσια διάταξη. Αν όχι, θεωρείτε ότι έχει εγκριθεί. Παρακαλώ να σημειώσετε ότι υπάρχει διερμηνία σε όλες τις γλώσσες, εκτός από δανέζικα, ιρλανδικά, κροατικά και λετονικά. Έγκριση των συστάσεων των συντονιστών. Πρέπει να γίνει, είναι το επόμενο θέμα. Βάση του άρθρου 205 μπορείτε να δείτε και στο σχετικό σημείωμα της συνεδρίασης της 21ης Ιουνίου 2018 ότι οι συντονιστές ε, έχουν προχωρήσει σε κάποιες συστάσεις. Υπάρχει σχετικό έγγραφο όπως είπα. Μπορείτε να το δείτε. Ε, ορισμός συγγητών, μεγάλος κατάλογος, και καγκάλα από το, από το ΕΛΚ, ορίστηκε η συγγήτρια για την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού ε, εγγράφου ταξιδιωτικού για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Η κυρία Χολμάιερ ορίστηκε εισηγήτρια για την πρόταση κανονισμού για το Εσωτερικό Ταμείο Ασφάλειας. Η Τάνια Φαγιόν από τους Σοσιαλιστές ορίστηκε εισηγήτρια για την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση στο πλαίσιο του Ολοκληρωμένου Ταμείου Διαχείρισης Συνόρων του σχετικού φακέλου. Η κυρία Νταλή, εισηγήτρια για την πρόταση κανονισμού για την ε, δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης. Επίσης, εισηγητής για το πρόγραμμα δικαιοσύνης, ο κ. Βαλέρο, για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την θέσπιση του προγράμματος δικαιωμάτων και αξιών. Η κυρία Φεράρα, από, τους, από το EFDD, ορίστηκε εισηγήτρια για την απόφαση του Συμβουλίου για την σύναψη από πλευράς Eurojust Συμφωνία συνεργασίας με την Ρουμανία. Τώρα, συντάκτης γνωμοδοτήσεων. Λένερς. Για το ΕΛΚ ορίστηκε συντάκτης για την πρόταση κανονισμού για την ψηφιακή Ευρώπη περίοδος 2017-2020. Λένερς επίσης. Εισηγητής για την πρόταση για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα Ταμείο Διαχείρισης Συνόρων και την ε, προμήθεια εξοπλισμού. Σοσιαλιστές, εισηγήτρια για το ζήτημα του, των ε, Ταμείων Συνοχής και Περιφερικής Ανάπτυξης, η κυρία Σωράγια Πόστ. Επίσης, ορίστηκε συντάκτρια γνωμοδότησης για την πρόταση κανονισμού για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Πλάς. Τερικάμπρας από τους Πράσινους ορίστηκε συντάκτης γνωμοδότησης για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του ενωσιακού προϋπολογισμού σε περιπτώσεις γενικευμένων ε, ελλείψεων όσον αφορά το κράτος δικαίου και την εφαρμογή του στα κράτη-μέλη. Βαλέρο. Γνωμοδότηση για την πρόταση κανονισμού σχετικά με τη δημιουργία του μηχανισμού υπερφρή προενταξιακής ε, διαδικασίας. Πρόταση κανονισμού, η ε, οδηγία, συγγνώμη, για την επαναχρησιμοποίηση των ε, πληροφοριών δημοσίου τομέα. Αναδιατύπωση. Ζήλστρα από το ΙΕΝΕΦ e ορίστηκε συντάκτης γνωμοδότησης σχετικά με την πρόταση κανονισμού για την θέσπιση κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Ταμείο, το Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το ε, Ταμείο για τη Θάλασσα και την Αλία, καθώς και τους δημοσιονομικούς κανόνες που διέπουν αυτά τα ταμεία, καθώς και το Ταμείο Μετανάστευσης Ασύλου, Διαχείρισης Συνόρων και Θεωρήσεων. εγκρίνει η Επιτροπή μας τις συστάσεις των συντονιστών αυτές. Δεν βλέπω να υπάρχουν αντιρρήσεις, επομένως θεωρώ ότι εγκρίνονται. Σημείο 3. Ε, κατεξοδότηση και εκτελεστικές πράξεις. Έγκριση του προγράμματος εργασίας Κομισιών για το 2018 και τη χρηματοδότηση των ε, δράσεων της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εσωτερική, στο, πλαίσιο του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλισης για την πρόληψη, την αντιμετώπιση και την ε, καταπολέμηση του, της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Λάβαμε εκτελεστική πράξη της Κομισιόν για, την, ε, για το πρόγραμμα εργασιών της Κομισιόν του 2018 και τη χρηματοδότηση αυτού στο πλαίσιο του, του, ε, του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλισης. Το, ο μηχανισμός για την ε, πρόληψη και τη διαχείριση κρίσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο βασικός κανονισμός είναι ο κανονισμός 514 του 2014 και η παραλαβή αυτή αυτής της ε, ε, πρότασης ε, κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της ΛΥΜΠΕ μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας και στις 19 Ιουνίου. Ορίστηκε προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Αν έχετε τέτοιε ενστάσει, παρακαλώ ενημερώστε την γραμματεία τη ΛΥΜΠΕ πριν από τι 10 Ιουλίου του 2018, δηλαδή αύριο έω τι 12 το μεσημέρι. Ο πρόεδρο έχει αποστείλει μαζί με τον πρόεδρο της ΕΚΟΝ κοινή επιστολή προς την Επίτροπο Γιούροβα για την διαβίβαση πριν από το καλοκαίρι πιθανής ε, κατεξοδότησης πράξης η οποία θα ορίζει χώρες που θα βρίσκονται στον κατάλογο επικινδύνων χωρών με βάση τον, την οδηγία για την, ε, ε, για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Ψηφοφορία ε, θα γίνει αύριο στις 9 και 4 ξεκινάει παρακαλώ φροντίστε να έχετε τις ηλεκτρονικές κάρτες ψηφοφορίας σας μαζί σας Λοιπόν, έχω και μια ανακοίνωση να σας κάνω. Μάλλον θέλω να δώσω το λόγο στους ε, διερμηνείς για να διαβάσουν το κείμενό τους. Can it be heard? Είναι η 35η μέρα διαφοράς με την διοίκηση και συνεχίζεται η απεργία των διερμηνέων. Οπότε σας πληροφορούμε ότι δεν πρέπει να υπάρξει υπέρβαση χρόνου. As I was signaled, it is done. Λοιπόν, αμοιβαία αναγνώριση ε, στις αποφάσεις δέσμευσης και δίμευσης. Σημείο 3, ημερήσια διάταξη, ενημέρωση για τις διαπραγματεύσει. Στις 20 Ιουνίου η Κορεπέρ συμφώνησε επί συμβαστικού κειμένου για τον κανονισμό αυτό χάρη στο σκληρό έργο της εισηγήτριάς μας, της κυρίας Γκρίσμπακ. Θα θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι πολύ ικανοποιημένη που σας, παρουσιάζω τη συμφωνία του τριμερούς διαλόγου για την, αναγνώριση, την αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων δέσμευσης και δίμευσης, που είναι ένα ευρωπαϊκό εργαλείο συνεργασίας. Πάρα πολύ χρήσιμο για να καταπολεμήσουμε τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος. από ό,τι θυμάμαι, 1% των εγκληματικών προσόδων ανακτώνται μέχρι στιγμής. Το υπόλοιπο 99 δεν ε, δημεύεται. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω όλους και όλους τους ηγητές για τη συνεργασία τους και τη δουλειά τους, ειδικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων, που ήταν πολύ πιο δύσκολες από ό,τι προβλεπόταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ φυσικά τις ε, ομάδες τριμερούς διαλόγου του Συμβουλίου και της Κομισιόν, παρά το γεγονός ότι είχαμε σημεία δύσκολα, παρόλα αυτά καταφέραμε να δουλέψουμε μέσα ένα πνεύμα συνεργασία με βάση τον κοινό μας στόχο που ήταν να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό εργαλείο. Αυτή η διαθεσμική διαπραγμάτευση ξεκίνησε τέλη Ιανουαρίου 2018 μετά την ψηφοφορία στην ε, Κοινοβουλευτική Επιτροπή και οργανώσαμε αμέσω ένα τριμερή διάλογο και υιοθετήσαμε μία προσωρινή συμφωνία τον Ιούνιο. Θα ήθελα να επανέλθω, αν μου επιτρέπετε, στους βασικούς στόχους που μας ε, οδηγούσαν καθ' όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Ε, το νήμα στις διαθεσμικές διαπραγματεύσεις ήταν να υπάρξει μία ε, ρήτρα, μία αναγνώριση με βάση τα θεμελιώδη δικαιώματα και αυτό το συμμερίζονταν γενικώ όλοι οι σκιώδεις εισηγητές. Ο βασικός μας στόχος αφορούσε την νομική μορφή του εργαλείου αυτού, του μέσου αυτού, Θέλαμε, όπως και η Κομισιόν, αυτή η νομοθεσία να είναι ένας κανονισμός. Δεν ήταν και τόσο απλό, γιατί αυτό δεν επιθυμούσε στην αρχή το Συμβούλιο και θέλαμε να, το, να επεκτείνουμε το πεδίο εφαρμογής και σε ποινικά θέματα. Το πετύχαμε τελικά. Δεύτερος στόχος ήταν ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Είπα και προηγουμένως, εκεί ξεκίνησαν δυσκολίες. Εδώ στην κοινοβουλευτική θέση είχαμε υιοθετήσει αυτή τη ρήτρα της μη αναγνώσης που βασίζεται στα θεμελιώδη δικαιώματα για την ε, δέσμευση και τη δίμευση. Στην ε, πρόταση της Κομισιόν και του Συμβουλίου όμως αυτή η ρήτρα δεν υπήρχε. Και το Συμβούλιο μάλιστα στην αρχή ήταν αντίθετο. Αφιερώσαμε τρεις συνεδριάσεις του τριμερούς διαλόγου και πολυάριθμες ενδιάμεσες συνεδριάσεις και καταφέραμε τελικά μία ρήτρα για τις αποφάσεις ε, δέσμευσης και ε, με μια ρητή αναφορά των θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και μια μνήα στη χάρτα. Ευχαριστώ ακόμα μια φορά του συναδέλφους για το πνεύμα συνεργασίας και συμβιβασμού για το θέμα αυτό και Ήδη από το πρώτο άρθρο βάζαμε και, βάλαμε και το σεβασμό της αρχής της αναλογικότητας και της αναγκαιότητας. Τρίτο σημείο. Δουλέψαμε για τις καλύτερες δυνατές δικονομικές εγγύησεις. Δηλαδή, ξαναείδαμε τον ορισμό των ενδιαφερομένων ατόμων από την απόφαση με την υποχρέωση ενημέρωσή του, ούτω ώστε το σύστημα ένδικων μέσων και προσφυγής να είναι ανοιχτό και αποτελεσματικό. Τέταρτο βασικό στόχο για την ομάδα μα ήταν η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα τη νομική πράξη για το θέμα των προθεσμιών. Πρέπει να σα πω ότι η θέση του Κοινοβουλή ήταν πολύ φιλόδοξη. Ε, προσθέσαμε πάρα πολλέ προθεσμίε. Δεν θέλω να μπω σε όλε τι λεπτομέρειε. Έχετε όλα τα στοιχεία στο έγγραφό σα. Δεν πετύχαμε όλα όσα επιθυμούσαμε για το σημείο αυτό, αλλά για τις διάφορες φάσεις της διαδικασίας καταφέραμε να βάλουμε το without delay, ούτως ώστε να επιτρέψουμε οι αρχές να μπορέσουν να εκτελέσουν πάρα αυτά τις αποφάσεις. Εν συνεχεία, και τέλος για τις προθεσμίες πάντα, ο κανονισμός ε, βάζει μία προθεσμία 45 ημερών, για την αναγνώριση και την εκτέλεση των αποφάσεων ε, δίμευσης. Θέλαμε πιο μικρή προθεσμία, το Συμβούλιο ήθελε 60, ο Συμβασμός μας έδωσε το 45 μέρες. Πρώτο τελευταίο στοιχείο, ο στόχος ήταν η καλή διαχείριση των ε, δεσμευμένων και δημευμένων ε, περιουσιακών στοιχείων και η επαναχρησιμοποίησή τους για κοινωνικούς σκοπούς. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο επ' αυτού έδινε μεγάλη σημασία στην ε, αναγνώριση του θύματος σε ό,τι αφορά τη διαχείριση των στοιχείων αυτών, των περιουσιακών αυτών στοιχείων και αυτό απεικονίζεται πολύ καλά στο τελικό κείμενο γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό τα θύματα να αποζημιώνονται φυσικά. Επίσης, πετύχαμε μετά από κάποιες συνεδριάσεις την ε, καλή επαναχρησιμοποίηση των ε, δημευθέντων αγαθών ε, για κοινωνικούς σκοπούς με ένα κεντρικό γραφείο διαχείρισης των περιουσιακών στοιχείων και ένα γραφείο για την αποζημίωση των θυμάτων, κυρίως των οικογενειών των αστυνομικών, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο στην προετοιμασία που κάναμε μαζί με τους συναδέλφους, δηλαδή πριν ξεκινήσουμε τους τριμερείς διαλόγους. Εν συνεχεία, η θέση σε ισχύ Απογοητευτήκαμε λιγάκι γιατί θα θέλαμε πιο μικρή προθεσμία. Τελικά όμως μετά από 24 μήνες θα εφαρμοστεί. Γιατί κατέτοιμα του Συμβουλίου θα πρέπει να αφήσουμε χρόνο στα κράτη-μέλη για να προσαρμόσουν την νομοθεσία του. Δεν είναι καταπληκτική προθεσμία, αλλά καλύτερα να εφαρμόσουμε σωστά αυτό το εργαλείο παρά να έχουμε μία νομοθεσία η οποία θα εφαρμόζεται μερικώ, άσχημα ή καθόλου στη χειρότερη περίπτωση. Καταληκτικά ευχαριστώ τους συναδέλφους για την ε, υποστήριξη, για τη δουλειά τους, για το πνεύμα επικοδομητικής συνεργασίας. Νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας ένα κανονισμό, το οποίο, οποίος είναι πάρα πολύ βάσιμος, μπορεί να είναι γρήγορος, αποτελεσματικός και πιο δίκαιος, ελπίζω, με καλύτερες εγγύσεις ό,τι αφορά τα βασικά δικαιώματα Αυτά είναι κάποια βασικά έτσι, στοιχεία, εντάχει σας τα λέω, για τους στόχους που προωθήσαμε μαζί με το Συμβούλιο και πλαισιωμένοι φυσικά από την ε, Κομισιόν. Ευχαριστώ κυρία Γκρίσμπεκ για το έργο σας, για αυτήν την πολύ σημαντική έκθεση. Κύριε Μακοβέη, βλέπω ότι θέλει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, κάποια λίγα λόγια θέλω να πω. Πρόκειται για κανονισμό που αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικονοτήτων για την ε, καταπολέμηση της τρομοκρατίας, του οργανωμένου κλίματος και της ε, περιστολής των δυνατοτήτων χρηματοδότησης αυτών των δραστηριοτήτων. Βεβαίως, ε, ευχής έργων θα ήταν να είχαμε ένα πιο ισχυρό και πιο ταχαίως εφαρμοζόμενο εργαλείο όσον αφορά τη δίμευση περισσοκών στοιχείων και τη δέσμευση. Εν πάση περιπτώσει, έχουμε πλέον κάποιους νέους κανόνες για τη δίμευση και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και στην ε, πρόταση της Κομισιόν το bona μέρος ε, αντικαταστήθηκε από, αντικαταστάθηκε από τον όρο ε, πληττόμενο μέρος. Θέλω να πω κάτι σε σχέση με αυτό. Αναφέρεται πλέον στο κείμενο ότι η δίμευση από τρίτους είναι δυνατή αν πρόκειται για δωρεά, αν η τιμή πώληση από τον καταδικαστέντε ε, ε, αποκλίνει ε, σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ε, αξία της αγοράς ή αν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη ένδειξη ότι η μεταβίβαση περιουσίας έχει γίνει για να αποφευχθεί η δίμευση. Τίποτα από όλα αυτά όμως δεν εξασφαλίζεται μέσω των διατάξεων της οδηγίας και δυστυχώς εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου γι' αυτό. Υπάρχουν επίσης χρονικά όρια για την αναγνώριση ε, της δίμευσης και της δέσμευσης που αυξήθηκαν από 30 στις 40 ημέρες σε σχέση με την πρόταση την αρχική της Κομισιόν. Πρόκειται λοιπόν για μια καθυστέρηση που θα αφορά την ίδια την αναγνώριση και την εφαρμογή, την υλοποίηση της απόφασης δίμευσης ή ε, δέσμευσης. Δηλαδή πρώτα δεσμεύεις κάτι βεβαίως και μετά το δημεύεις. Εγώ θα έλεγα ότι είναι πραγματικά ανάγκη η διαδικασία αυτή να ολοκληρώνεται πολύ πιο γρήγορα, διότι υπάρχει ο κίνδυνος να μην βρει τίποτα μετά στο τέλος από τον ε, καταδικαστέντα. Να μην βρει κανένα περιουσιακό του στοιχείο για να δημεύσει ή να δεσμεύσει. Εν πάση περιπτώσει αυτά ήθελα να πω και να επαναλάβω για άλλη μια φορά ότι πραγματικά θα προτιμούσα να είχαμε καταλήξει σε ένα πολύ ισχυρότερο εργαλείο. Ευχαριστούμε κυρία ε, Μακοβέη. Κυρία Γκρίσμπεκ, θέλετε να σχολιάσετε, να απαντήσετε. Έχετε ένα λεπτό στη διάθεσή σας. Ναι, καταλαβαίνω τις παρατηρήσεις της συναδέλφου. Και εγώ θα προτιμούσα κάτι τέτοιο. Ήθελα να πάμε πιο πέρα. Και για άλλα σημεία, πέρα από αυτό που ανέφερε η κυρία Μακουβέη. Αλλά δουλέψαμε πάρα πολύ γρήγορα, με για να βρούμε μια ισορροπία. Καταλαβαίνω πολύ καλά τι θα επιθυμούσε η κυρία Μακοβέη. Ήταν δύσκολη όμως η υιοθέτηση αυτής της ισορροπίας. Θα ήταν ενδιαφέρον να τα είχα όλα αυτά τα στοιχεία νωρίτερα, ούτω ώστε να λάβω υπόψη μου τα, τις επιθυμίες της για να είμαστε και πιο δυνατοί στη διαπραγμάτευση. Ε, Εκτός μικροφώνου. Δεν είναι αγώνα αυτό. Είπα ότι λυπάμαι απλώ. Έχουμε ήδη ε, μία οδηγία για την ε, δέσμευση και τη δίμευση που δεν ε, εφαρμόζεται σωστά ή λαθο λάθος από πολλά κράτη-μέλη. Αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα. επιση αυτή στιγμή λαμβάνεται δικαστική απόφαση για να καταδικαστική εναντίον κάποιου για δέσμευση ή δίμευση, αυτό θα πρέπει να γίνει γρήγορα, να εφαρμοστεί γρήγορα. Γιατί το πρόβλημα δεν είναι ότι θα πάει αυτό ε, το να πάει στη φυλακή. Το θέμα είναι πώ θα ανακτήσουμε τα περιουσιακά του στοιχεία και πώ θα ξαναμπούν τα χρήματα στον προπολογισμό. Και δεδομένου ότι μιλάμε για δισεκατομμύρια ευρώ, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ευχαριστώ, κυρία Μακοβέη. Σας ενδιαφέρει πολύ αυτό το θέμα. Ε, ασχοληθήκαμε και στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία με αυτό. Του, του, αύριο ψηφίζουμε. Και Πιστεύω και η συγγήτρια ήθελε να, πάει, να πάμε πιο μακριά, αλλά πάντα στη ζωή χρειάζεται να πετύχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στο τι μπορούμε και το τι θα θέλαμε να πετύχουμε. Αύριο θα γίνει ψηφοφορία του κειμένου. Στην, ε, στις ψηφοφορίες θα ξεκινήσουν σε 9 και 50 ακριβώς. Πάμε στο σημείο 4, που είναι μια ανταλλαγή απόψεων με την κυρία Κάθριν Ντεμπόλ, εκτελεστική διευθύντρια της Europol. Καλώς ήρθατε. Με μεγάλη χαρά σας ε, υποδεχόμαστε στην Επιτροπή μας. Κυρία Ντεμπόλ, διοριστήκατε ως νέα εκτελεστική διευθύντρια της Europol 1η Μαΐου και με μεγάλη χαρά σας υποδεχόμαστε εδώ στην Επιτροπή Ξέρω ότι σας απασχολούν, ε, ή μάλλον και εμάς μας απασχολούν τα ίδια θέματα της αρμοδιότητάς σας. Ε, θα σας δώσω, κυρία Ντεμπόλ, το λόγο για 10 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι, είναι μεγάλη μου τιμή να βρίσκομαι εδώ ενώπιον σα, ενώπιον τη Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, με την νέα ιδιότητά μου ω εκτελεστική διαθετήρια τη Europol. 70 μέρε ε, κλείνουν από τότε που ανέλαβα τα ενία τη Europol. Χαίρομαι που έχω τη δυνατότητα να μοιραστώ μαζί σας με την Επιτροπή σας που είναι από τα πιο σημαντικά ενδιαφέροντα μέρη για μας ε, τις πρώτες μου εμπειρίες από την Europol. Από την πρώτη στιγμή εργάστηκα προς την επίτευξη των ε, στόχων που σας ανακοίνωσα στις 29 Ιανουαρίου στην ακρόαση εδώ στη Λίμπε για τον διορισμό μου. Και σας διαβεβαιώ ότι θα συνεχίσω να εργάζομαι για τους ίδιους στόχους στι επόμενες εβδομάδες και μήνες. Μία από τις πρώτες μου προτεραιότητες είναι να κατανοήσω τις ανάγκες, προσδοκίες και ανησυχίες των ε, βασικών ε, ενδιαφέρμενων μερών για την Europol, ε, τις αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη. Τι τελευταίε 70 μέρε, λοιπόν, έχω συναντηθεί με διοικητέ αστυνομία και επικεφαλής άλλων αρχών επιβολή του νόμου σε πολλά κράτη-μέλη. Ως ε, διοικήτρια της Europol θέλω να γνωρίζω ακριβώς ε, ποιες είναι οι προσδοκίες αυτών των εθνικών αρχών από την Europol. Πιο ειδικά θα ήθελα να ανταποκριθώ με πιο αποτελεσματικό τρόπο ε, στις επιχειρησιακές τους ανάγκες και στις στρατηγικές τους ανάγκες για την καλύτερη αντιμετώπιση μελλοντικών απειλών. Κατόπιν συζητήσεων ε, με την πλειονότητα των κρατών μελών, επιβεβαιώνω ότι οι εθνικέ αρχέ δηλώνουν την ικανοποίησή του ό,τι αφορά τη στήριξη που λαμβάνουν από την Europol. Υπάρχει θετική ανατροφοδότηση που αφορά κατά βάση την ε, επί 24 ώρου βάση διαθεσιμότητα τη επιχειρηματική μα υποστήριξη, ε, την τεχνογνωσία και πραγματομοσύνη της Europol σε εξειδικευμένα πεδία, ε, για παράδειγμα έγκλημα στον κυβερνοχώρο και, και τρομοκρατία και η στήριξη επιτόπου τους Europol κατά τη διάρκεια των ερευνών. Όμως ε, οι διοικητές ε, της αστυνομία μου είπαν ότι υπάρχουν και τομείς όπου θα μπορούσε να αυξήσει τον αντίκτυπό της η Europol και εμείς θέλουμε να βελτιώσουμε περαιτέρω αυτή τη συνεργασία. Οι επικεφαλείς των Εθνικών Αρχών Επιβολή του Νόμου μου ζήτησαν να βελτιώσουμε την αναλυτική μα ικανότητα, να δίνουμε ε, πιο τεχνική υποστήριξη και υποστήριξη προγνωμοσύνη. Οι δραστηριότητε impact, που είναι δηλαδή οι προτεραιότητε προτεραιότητές μα ω προ το έγκλημα να διασυνδέονται καταλήλω με τι εθνικέ προσπάθειε και να διευκολύνουμε την επικοινωνία μεταξύ ε, των αρχών επιβολή του νόμου στην Ευρώπη. Η διάσκεψη των διοικητών τη αστυνομία ε, το Σεπτέμβριο θα είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ε, συζητήσουμε πώς έχει κατάσταση σήμερα και ποια βήματα πρέπει να λάβουμε στο μέλλον. Μία ακόμα σημαντική πτυχή του έργου μου κατά τις πρώτες εβδομάδες της θητείας μου είναι συνεργασία με, τις, με τους άλλους οργανισμούς ε, δικαιοσύνης και εσωτερικών. Είναι ένας τομέας ο οποίος έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια και εγώ θέλω να συνεχιστεί αυτή η τάση περαιτέρω. Θέλω λοιπόν να διασφαλίσω την συμπληρωματικότητα αλλά και την ευελιξία, προκειμένου η συνεργασία μεταξύ των ε, ε οργανισμών και το σχετικό πλαίσιο να είναι ε, πιο αποτελεσματικό. Ήδη έχω συναντηθεί με ε, οργανισμούς δικαιοσύνης και ιστορικών υποθέσεων, όπως με τον πρόεδρο της Eurojust, ε, τους διοικητικούς, εκτελεστικούς διοικητές της ΕΠΟΛ, του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, της Λίζα και του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Ισότητας των Φύλων και της Υπηρεσίας Εξωτερικές Δράσεις. Επίσης, συναντήθηκα και με τον ε, εκτελεστικό διευθυντή της Frontex και ένα απτό παράδειγμα που έχω να σας δώσω είναι ότι για πρώτη φορά θα γίνει μια κοινή συνάντηση του Διοικητικού Συμβουλίου Frontex και Europol τον Οκτώβριο για να συζητήσουμε τα κοινά μας ζητήματα. Με όλους τους οργανισμούς έχουμε συζητήσει πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τη συνεργασία από επιχειρησιακής και στατικικής άποψης. Και θεωρώ ότι υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των οργανισμών και ισχυρή βούληση επίσης. Η Europol θα προεδρεύσει του δικτύου των οργανισμών ΔΕΗ το 2019. Αυτή η σύνθεση και αυτό το βήμα ε, αποτελεί ακόμα μία ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συνεργασία και να εντοπίσουμε δυνατότητες συνεργειών μεταξύ των οργανισμών. Είμαι αρχάρι βέβαια και εγώ εδώ, οπότε μου παίρνει και εμένα λίγο χρόνο στη Europol να μάθω περισσότερα για την δομή, τις διαδικασίες ε, που ακολουθούνται. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να καταλάβω τον ρόλο ε, και τα καθήκοντα των συναδέλφων μου στο πλαίσιο του οργανισμού μας. Γι' αυτό και ξεκίνησα μία σειρά άτυπων συναντήσεων με τους ε, συναδέλφους μου για να μάθω περισσότερα για το έργο τους ε, στο σύνηθες ε, περιβάλλον, εργασιακό τους περιβάλλον. Εδώ έχω αντίστοιχη εμπειρία, όπως και με τους οι εμπειρίες μου μάλλον ήταν ίδιε ίδιες, και με τι συναντήσει μου με τους διοικητέ ε, των ε, Εθνικών Αρχών του Νόμου, ότι είναι ένας ε, οργανισμός που λειτουργεί καλά, με έμπειρο και προσιλωμένο προσωπικό. Και πολλοί είπαν ότι θέλουν να συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια. Πολλά μέλη του προσωπικού μα έχουν ε, εξειδικευμένη προγνωμοσύνη, για παράδειγμα από αποκριτογράφηση ή εξάρθρωση ε, εργαστηρίων ναρκωτικών ουσιών. Για παράδειγμα, η Europol πρόσφατα βοήθησε και υποστήριξε τις ισπανικέ αρχές στην εξάρθρωση ενός από τα, μεγαλύτερα δίκτυα ε, ναρκωτικών στην Ισπανία. Θέλουμε να ενισχύσουμε παράλληλα την ε, ε, καταπολέμηση της ε, διακίνησης ανθρώπων και να βοηθήσουμε τις εθνικές αρχές για την καταπολέμηση των δευτερογενών μετακινήσεων στην Ευρώπη. Αυτά τα βασικά στοιχεία θα τα υπερθυμίσουμε και στο άτυπο Συμβούλιο ΔΕΗ στο Ινσμπρουκ αυτή την εβδομάδα. Στο πλαίσιο της μετανάστευσης, η Europol δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην καταπολέμηση ενό από τα βασικά ζητήματα σήμερα που είναι η διακίνηση και μετάλλευση ε, μεταναστών σε δύσκολες και επικίνδυνες καταστάσεις. Και αυτό αφορά και παιδιά. Αυτή η εγκληματική δραστηριότητα και αυτή η αγορά, αν θέλετε, είναι από τις πιο επικερδείς και συνδέεται άρρηκτα και με άλλες μορφές ε, εγκλήματος όπως η διακίνηση ναρκωτικών και ούτω καθεξής. Ένα από τα βασικά ε, μελήματα και καθήκοντα της Europol είναι να παράσχει ε, υποστήριξη στις διοικητικές έρευνες, στις αστυνομικές έρευνες που γίνονται μάλλον από τις εθνικές αρχές. Και έχουμε ανταποκριθεί σε μία σειρά υψηλού επίπεδου έρευνες όπως για παράδειγμα και στην περίπτωση, στην υπόθεση της ε, δολοφονίας ε, δημοσιογράφων και στη Μάλτα και στη Σλοβακία. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει λάβει ισχυρή θέση και ζήτησε μεγαλύτερο ρόλο της Europol σε αυτές τις έρευνες και λίγο μετά από την έναρξη των εθνικών ερευνών και η Μάλτα και η Σλοβακία ζήτησαν την συνδρομή της Europol. Οι δραστηριότητες υποστήριξής μας λοιπόν συνεχίζουν, η συνεργασία και με, ε, με τις εθνικές αστυνομικές αρχές και των δύο χωρών συνεχίζεται και έχει αποτελέσματα. Θα εξακολουθήσουμε να υποστηρίζουμε τις αρχές της Μάλτας και της Σλοβακίας ε, με κάθε δυνατό τρόπο. Στρέφουμε τώρα στις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Europol. Θεωρώ ότι μία από τις βασικές προκλήσεις για την Europol αυτή τη στιγμή είναι το πρόβλημα που υπάρχει με ε, τους πόρους ενώ αντιμετωπίζουμε νέες επιχειρησιακές προκλήσεις και αυξανόμενο όγκο δεδομένων, η Europol χρειάζεται και αυξημένους πόρους για να διατηρήσει ε, την, ε, τις τεχνολογίες εχμής που έχει σε πληροφορικά συστήματα και αναλυτική ικανότητα. Παράλληλα, ε, αυτό θα πρέπει να έχει αντίκρισμα και στα επίπεδα θέσεων στο προσωπικό, ανθρωπίνου δυναμικού. Το Φεβρουάριο το Διοικητικό Συμβούλιο της Europol υιοθέτησε ένα προσχέδιο προπολογισμού που προέβλεπε τα απαιτούμενα επίπεδα επενδύσεων. Δυστυχώς, η σημερινή πρόταση για τη Europol στο πλαίσιο του προσχεδίου του Ευρωπαϊκού Προπολογισμού για το 2019 ε, δεν στέκεται στο ύψος των αναγκών της Europol και μάλιστα επιβάλλει και ουσιαστική μείωση σε σχέση με τον προπολογισμό του 2018. Στις ε, συζητήσεις μου με τους διοικητές ε, των Εθνικών Αστυνομικών Αρχών και άλλων αρχών, πολλές φορές άκουσα ότι η Europol είναι μία από τις, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς ε, ε, οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εγώ αυτή την εμπειρία έχω αποκομίσει. Και υπάρχει επίσης και συνένεση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να επενδύσει στα εργαλεία ασφαλείας που διαθέτει. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και η Europol. Όμω έχουμε ε, νέο εκτελεστικό διευθυντή τη Europol και εξ ονόματο Europol πρέπει να σας ε, πω ότι με προβληματίζει ιδιαίτερα αυτό το κενό μεταξύ, το χάσμα μεταξύ τη ε, αρχική πρόταση του Europol, όπω υιοθετήθηκε από τα κράτη-μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο, και της τρέχουσας πρότασης για το 2019. Το κενό αυτό αντιστοιχεί σε 21 εκατομμύρια ευρώ και 38 θέσει εργασία. Και ε, αυτή η τάση επιβεβαιώνεται και στις προτάσεις για το πολιτε δημοσιονομικο δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 που δεν προβλέπουν ουσιαστική αύξηση των πόρων για την Europol. Εάν δεν ε, ε, υπάρξει επανόρθωση αυτού του κενού ε, και δεν παρασχεθούν οι απαραίτητοι πόροι, τότε και οι συνεχιζόμενες και οι προγραμματισμένες μας πρωτοβουλίες σε διάφορους τομείς θα επηρεαστούν αρνητικά. Αυτό σίγουρα θα επηρεάσει αρνητικά και τις επιχειρησιακές ικανότητες της Europol. Έχουμε συμφωνήσει να έχουμε αξιωματούχου στην Ιταλία και στην Ελλάδα για τους ελέγχους ασφαλείας και αξιωματικού συνδέσμου στα Δυτικά Βαλκάνια. Συμφωνήσαμε όλοι ότι η αποκρυπτογράφηση και η στήριξη των κρατών μελών σε αυτόν τον τομέα είναι ε, απαραίτητης και ω διοικήτρια της Europol ε, σας καλώ ε, να υιοθετήσετε τον κατάλληλο προπολογισμό για, για την κάλυψη των αναγκών αναλάβαμε 20.000 περισσότερες επιχειρήσεις από το 2016 και θεωρούμε ότι αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί περαιτέρω. Χρειαζόμαστε λοιπόν τους αντίστοιχους πόρους για να υποστηρίζουμε τα κράτη-μέλη στις έρευνές τους για την τρομοκρατία και την ε, νομοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Χρειαζόμαστε τα πληροφορικά μας ε, συστήματα για να σας υποστηρίξουμε και με την αυξανόμενη ζήτηση για τις υπηρεσίες και με αυτό το αυξανόμενο κενό στη χρηματοδότηση, αυτό μας προβληματίζει ιδιαίτερα. Εσείς στο Κοινοβούλιο έχετε συμβάλει ιδιαίτερα ε, στην αύξηση και στην ανάπτυξη της Europol από τότε που έγινε οργανισμός ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2010 έχετε προτείνει επιπρόσθετους πόρους και θέσεις προσωπικού για τη Europol για να αντιμετωπίζει ε, τις εξελισσόμενες προκλήσεις. Ε, πραγματικά ευχαριστώ την ευγνωμοσύνη μου και προς την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών που έχει διδραματίσει θεμελιώδη ρόλο στην ανάπτυξη του οργανισμού μας τα τελευταία χρόνια. Χαιρετίζω ε, και την έκθεση της ε, ειδική Επιτροπής για την Τρομοκρατία. Χαιρετίζω την απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την εντολή να διαπραγματευτεί συμφωνίες επιχειρησιακής συνεργασίας με τρίτες χώρες. Κυρίε και κύριοι, δεσμεύομαι να συνεχίσω να σας ε, παρέχω όσο γίνεται περισσότερη στήριξη με την παροχή πληροφοριών στους τομείς ειδίκευση και αρμοδιότητά μου. Είμαι βέβαιη ότι πολλοί από εσά θα έχετε ερωτήματα που θα με επιτρέψουν να επισέλθω σε περισσότερε λεπτομέρειε. Κλείνοντα, θα σταθώ ε, στι προτεραιότητέ μου. Πρέπει να κατανοήσουμε τις προσδοκίες ε, των εθνικών αρχών και να βρούμε μια ισορροπία με τις προσδοκίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να βρούμε την καλύτερη δυνατή επιχειρησιακή στήριξη, αναλυτική και ε, τεχνολογική ικανότητα βασικό μας μέλημα. Πρέπει να διασφαλίσουμε ε, τους απαραίτητους πόρους για την ανάπτυξή μας κατά τη διάρκεια της ε, θητείας μου και να διασφαλίσουμε και την ε, διαφανή συνεργασία και ανοιχτό πνεύμα συζήτησης με όλα τα διεθνώνα μέρη. Ε, να υπογραμμίσω και πάλι τη σημασία που αποδίδω στη σχέση μεταξύ Europol και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Κοινοβουλίου και ότι είμαι πάντα στη διάθεσή σας. Σας ευχαριστώ ε, για την προσοχή σας και με τα χαρά να απαντήσω στις τυχόν ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πολ. Ήσασταν σαφέστατοι, ιδίω όσον αφορά τα δημοσιονομικά ζητήματα και τα προβλήματα προπολογισμού που αντιμετωπίζει η Ευρωπόλ. Ο κύριο Διζντεμέρα έχει το λόγο από τον μακρύ κατάλογο μιλητών που έχουμε καταρτήσει. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ την ε, Γενική Διευθύντρια της Europol και την καλωσορίζω. Εκτιμούμε πολύ που μόλις 70 μέρες αυτή στιγμή ανέλαβε τα καθήκοντά της, έρχεται εδώ στην Επιτροπή μας. Η παρέμβασή της συνοψίζεται σε τρία λόγια. Στόχοι, προκλήσεις και προτεραιότητες. Δεν θα μιλήσω για τους στόχους γιατί τους ξέρουμε και μας τους ε, ανέφερε και στους προηγούμενους, ε, στην προηγούμενη εμφάνισή της και συμφωνούμε. Θα ήθελα να κάνω απλώς λίγα σχόλια λοιπόν σε ό,τι αφορά τις προκλήσεις και τα ένδικα μέσα. Η, συγγνώμη, και τους πόρους. Η Europol χρειάζεται και τις 38 θέσεις εργασίας και τα 21 εκατομμύρια. Και τα χρειάζεται Χρειάζεται αυτούς τους πόρους. Γιατί? Ξέρετε ότι η πληροφορική είναι η ραχοκοκαλιά της Europol. Και η πληροφορική μπορεί να επιδεινωθεί. Μπορεί διάφορα σχέδια, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν, να μην ολοκληρωθούν λόγω έλλειψης ε, πόρων, κονδυλίων. Αυτό είναι το πρώτο που θα ήθελα να πω. Δεύτερον, μας φαίνεται πολύ έξυπνη πορεία, η πορεία σας, κυρία μου. Το γεγονός δηλαδή ότι συναντηθήκατε με 20 αστυνομικούς διευθυντές αυθυντές, και σχεδόν με όλα τα θεσμικά όργανα, οργανισμούς και υπηρεσίες της Ένωσης που ασχολούνται με την ασφάλεια. Το να δώσετε ε, στήριξη, το να επενδύσουμε στην τεχνολογία και το να έχετε καλή σχέση με το Κοινοβούλιο στα πλαίσια της ε, διαφάνειας ε, μας φαίνεται εκ των ονουκάνευ. Ξέρετε πολύ καλά ότι το Σεπτέμβριο θα κάνουμε τρίτη συνεδρίαση της ομάδας κοινοβουλευτικού ελέγχου και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας για το θέμα αυτού του ελέγχου του προϋπολογισμού. Και επίσης, τελευταία σχόλια, την περασμένη εβδομάδα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη σύστασή του για τη διαπραγμάτευση χωριστών α, συμφωνιών με την Ιορδανία, Τουρκία, Ισραήλ, Τουρκία, ε, Λίβανο, ε, Αίγυπτο και Αλγερία. Χωριστέ συμφωνίε με αυτέ τι τρίτε χώρε. Είναι 8 χώρε. Μπορείτε να μα μιλήσετε λιγάκι για αυτή την προστιθέμενη αξία ε, που θα έχουν αυτές οι χωριστές διμερείς συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αυτές τις 8 τρίτες χώρες για την ασφάλεια των Ευρωπαίων πολιτών. Κυρία Γκόμες, ευχαριστώ κυρία Διευθύντρια. Χαίρομαι που είστε μαζί μας και συμμερίζομαι και εγώ τις ανησυχίες που εκφράσατε ότι μειώνεται ο προϋπολογισμός της Ευρωπόλ την ίδια στιγμή που τα καθήκοντα και οι, οι ικανότητες ε, που χρειάζεται για, την εκπλήρωση αυτών των ε, καθηκόντων αυξάνονται. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μας προειδοποιήσατε γι' αυτό και αυτό βεβαίως ε, μας ε, γεμίζει με ευθύνε όσον αφορά τις διαπραγματεύσει στις οποίες θα προσέλθουμε με το Συμβούλιο και την Κομισιόν. Από τις επαφές που είχα με αρχές επιβολής του νόμου στα κράτη-μέλη ε, έχω σχηματίσει την άποψη ότι ε, ε, είναι ευρύτατα παραδεκτή η σημασία που έχει η Ευρωπόλ και είναι πραγματικά πολυάριθμοι οι τομείς στους οποίους η Ευρωπόλ μπορεί να συμβάλλει σημαντικότατα όσον αφορά την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματο ή την ε, τρομοκρατία, για παράδειγμα. Και εδώ πολλέ φορέ τα κράτη-μέλη δεν κατανοούν τι ακριβώ διακυβεύεται. Μιλώ για ε, μια ε, ευρωπαϊκή FIU. Είναι και έτοιμα δικό μας, μιας χρηματοοικονομικής μονάδας δηλαδή, που θα, που θα πρέπει να δημιουργηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι αίτημα το οποίο έχουμε υποβάλει πολλέ φορέ στι διαπραγματεύσει μα με τα άλλα θεσμικά όργανα. Και είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε αυτό. Διότι αν οι κυβερνήσει του Συμβουλίου πραγματικά εννοούν τι εξαγγελίε του όσον αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία, πρέπει ταυτόχρονα να καταπολεμηθεί και το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Ε, και αυτό είναι απαραίτητο να γίνει και σε ενωσιακό επίπεδο. Άτυπα πολλά γίνονται, αλλά πρέπει να πάρουν επίσημη μορφή ε, αυτές οι συνεργασίες. Και το ερώτημά μου προς εσάς είναι, ε, έχει σημειωθεί πρόοδος, ποιες είναι οι προκλήσεις που ε, διαπιστώνετε εσείς όταν ε, ιδίω γνωρίζουμε ότι κάποια κράτη-μέλη πλέον λειτουργούν ως κόμβοι για τα κρυπτονομίσματα, που ξέρουμε πολύ καλά πόσο τελικά έχουν αξιοποιηθεί από το οργανωμένο έγκλημα και την, ε, και την τρομοκρατία, τα κρυπτονομίσματα αυτά. Εγώ δεν θα σας απευθύνω ερωτήματα όσον αφορά τις έρευνες που γίνονται στην Μάλτα και στη Σλοβακία και που αφορούν την δολοφονία δημοσιογράφων όπου οι αρχές ζήτησαν οι ίδιες τη σύνδρομη της Ευρωπόλ. Αλλά Εξ όσων γνωρίζουμε, τουλάχιστον από την υπόθεση της Μάλτας, υπάρχουν και ορισμένα όρια στην ε, συνεργασία αυτή. Όρια που πηγάζουν από την ίδια την εντολή της Ευρωπόλ ε, ε, και από το γεγονός βεβαίως ότι δεν μπορεί η Ευρωπόλ να υπερβεί τα όσα της έχουν ζητήσει οι ίδιες αρχές που έχουν ζητήσει τη βοήθειά της. Όταν λοιπόν έχουμε αρχέ οι οποίε δεν θέλουν να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, ε, τότε προφανώ και η Ευρωπόλα αντιμετωπίζει ένα περιορισμό στη δράση τη. Και αυτό έχει σχέση και με την εντολή τη Ευρωπόλη και το πλαίσιο δράση τη. Τι μπορείτε να μα πείτε ω προ αυτά, Ποια είναι η δική σα θεώρηση. Ξέρω ότι ε, έχετε αναλάβει τα καθήκοντά σας πριν από λίγες σχετικά μέρες, όμως φαντάζομαι ότι είχατε την ευκαιρία μέχρι στιγμή να σχηματίσετε μια εικόνα και θα θέλαμε να μα την παρουσιάσετε. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρο. Παρακαλώ, συνάδελφοι, σεβαστείτε το όριο των δύο λεπτών. Ο λόγο στην κυρία Μακοβέη. Δύο λεπτά θα μιλήσω. Καταρχάς θα ήθελα να σας συγχαρώ για την εκλογή σας. Είναι και η πρώτη φορά που σας συναντώ προσωπικά. Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στο έργο σας και καλή τύχη. Κατά τη γνώμη μου, η Ευρωπόλ μπορεί να αποτελέσει στο μέλλον την Ευρωπαϊκή Ιντερπόλ. Ήδη Πρόκειται για το σημαντικότερο οργανισμό που έχουμε στη διάθεσή μα για την καταπολέμηση του διασυνοριακού, του σοβαρού, του οργανωμένου εγκλήματο τη τρομοκρατία. Ε, και πρόκειται για, μια, για ένα τεράστιο και πολύπλοκο έργο βεβαίω το να εντοπίζει και να αντιμετωπίζει κανεί όλε αυτέ τι εγκληματικέ δραστηριότητε. Όσον αφορά τα, τα πρακτικά σημεία, νομίζω ότι το σημαντικότερο που, θέμα που θέσατε είναι βεβαίω ο προπολογισμό σα. Και είπε και η συνάδελφό μου, η Άννα Γκόμε, ότι είναι πραγματικά δύσκολο να καταλάβουμε για ποιο λόγο μειώθηκε ο προπολογισμό για το 2019 κατά 8 εκατομμύρια σε σχέση με τον προπολογισμό του 2018. Όταν γνωρίζουμε όλοι ότι τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις βεβαίως καθώς και το έργο της Ευρωπόλ αυξάνεται σταθερά. Μιλάμε για καταπολέμηση κυβερνοεγκλήματος, ε, την ε, αποτροπή και την καταπολέμηση τρομοκρατικών επιθέσεων, ε, απειλών, διασυνοριακών, περιπτώσεων απάτης. Όλα αυτά εμπίπτουν στις δραστηριότητες Ευρωπόλ. Έχω λοιπόν να σας δώσω κάποια ερωτήματα. Όσον αφορά αυτήν την προτινόμενη μείωση κατά 8 εκατομμύρια του προπολογισμού σας, ποιες δραστηριότητες θα εγκαταλείψετε, θα αναγκαστείτε δηλαδή να εγκαταλείψετε, αφού θα σας λείπουν αυτά τα 8 εκατομμύρια. Είχατε ήδη κάποιες προγραμματισμένες δράσεις για το 2019 τις οποίες θα αναγκαστείτε να περικόψετε να ματαιώσετε για το 2019 λόγω της περιστολής του προπολογισμού. Τρίτον, ποιες είναι οι ανάγκες σας, οι χρηματοδοτικές, οι προτεραιότητες σας που αντιστοιχούν σε, σε αυτές τις προτεραιότητες, οι δημοσιονομικές σας οι ανάγκες λοιπόν. Θέλω δηλαδή να, ρωτώ, να ρωτήσω ποια είναι τα κονδύλια που είναι απαραίτητα προκειμένου η, η Ευρωπόλη να μπορεί να ανταποκριθεί στις προτεραιότητες που έχει η ίδια θέση. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Μακοβέη. Η κυρία Ιντβελτ. Ευχαριστώ. Uh, κυρία Βόλα, καλώ ήρθατε και πάλι στη Λίμπε. Δεύτερη φορά έρχεστε εδώ όντω. Ορισμένα συγκεκριμένα ερωτήματα μετά και από την παρέμβαση τη κυρία Γκόμες. Ε, για τις ε, έρευνες εξυχνίας των δολοφονιών στη Μάλτα και στην Σλοβακία. Μιλήσατε για αγαστή συνεργασία και ότι οι τοπικές αρχές δηλώνουν την ικανοποίησή τους από τη συνδρομή σας. Όμως, ε, δεν είναι ιδιαίτερα μετριοπαθές όλο αυτό, γιατί είναι πολύ ανησυχητικά τα σημάδια. Πρώτον, έχουν περάσει τόσοι μήνες και ούτε καν υπάρχει ένα, μια πρώτη ένδειξη διαλεύκανσης ε, των δολοφονιών αυτών προς την κοινή γνώμη. Όσοι λοιπόν έχουν διαπράξει τις δολοφονίες ή ε, ζήτησαν, ε, διέταξαν αυτές τις δολοφονίες, ακόμα είναι ελεύθεροι. Τι έχει γίνει λοιπόν ουσιαστικά. Έτσι κι αλλιώ ε, αμφισβητείται πλέον ε, η ανεξαρτησία των αστυνομικών αρχών στη Μάλτα. Μετά υπάρχει το ζήτημα του τηλεφώνου ενός, ε, της δήμευσης ενός τηλεφώνου ενός δημοσιο, τσέχου δημοσιογράφου Σλοβακία. Θα ήθελα, αν έχετε περισσότερες πληροφορίες, να τη μοιραστείτε μαζί μας. Είπατε ότι παρέχετε κάθε δυνατή συνδρομή προς τη Μάλτα και τη Σλοβακία. Τι είδους περιορισμούς όμως ε, βλέπετε και πού θα θέλατε περισσότερες ε, αρμοδιότητες. Και το δεύτερο ερώτημα. Υπάρχει πίεση ως προς το κράτος δικαίου σε μια σειρά κράτη-μέλη. Ε, η δικαιοσύνη, της οποίας η ανεξαρτησία πλέον πλήττεται. Κάποιες φορές ακόμα και οι ίδιες αρχές εμπλέκονται στην νομοποίηση εσόδων παράνομες δραστηριότητε ή στη διαφθορά, εποπτικές αρχές. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη στο καθημερινό σας έργο στην ανταλλαγή πληροφοριών. Για παράδειγμα, ε, στην ε, μονάδα αυτή χρηματοοικονομικών πληροφοριών, γιατί ξέρετε ότι κάποιες από τις πληροφορίες που ε, μπαίνουν στο σύστημα μπορεί να μην είναι αξιόπιστες. Πώς το χειρίζετε αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ, Στοχόφσκι. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Διευθύντρια για την παρουσία της εδώ. Δύο λεπτά έχω στη διάθεσή μου, επομένω ε, τρία ερωτήματα να σα θέσω εν συντομία. Πρώτον, πριν από δύο χρόνια, ο προκάτοχό σα είχε πει στην Επιτροπή μα ότι θα καταπολεμήσει συγκεκριμένε ε, μορφές απάτης ε, που διαπράττονται ευρέως ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ στο Βέλγιο υπάρχει βέβαια ένας νόμος που το επιλύει και το καλύπτει, αλλά ε, πρόκειται για μία μορφή απάτης ε, που, που ουσιαστικά παράγει κέρδη 13 δις ευρώ. Δεν έχει γίνει όμως κάτι στην πράξη σε ό,τι αφορά τα οχήματα και τα πειραγμένα κοντέρ. Δεύτερον, ε, εγώ είμαι σκιώδης συζητητής ε, στην Επιτροπή ε, Προπολογισμών. Πάντα λοιπόν προσπαθώ να αυξήσω τον προπολογισμό της Europol και τις θέσεις του προσωπικού για τους οξαματούχους που εργάζονται σε χώρες σε κατάσταση κρίσης, όπως στη Λιβύη, για παράδειγμα, που προσπαθούν να καταπολεμήσουν την ε, διακίνηση ανθρώπων. Επομένω, να ρωτήσω, υπάρχει βελτίωση ό,τι αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών και Europol, γιατί ξέρω το 2016 ορισμένα κράτη-μέλη δεν έδιναν στοιχεία ή έδιναν ελάχιστα Υπάρχει βελτίωση προ αυτό. Ευχαριστώ. Very much and the last... Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντεμπχέ, τελευταίος ομιλητής. Ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Σας ξαναβλέπουμε λοιπόν δύο μήνες περίπου μετά από τον διορισμό σας. Άκουσα με μεγάλη προσοχή την παρέμβασή σας ε, και έχω να πω τα εξή. Η φιλοσοφία που ε, ε, υπερασπίζεστε για τον ρόλο της Europol είναι πραγματικά πολύ σωστή. Μιλήσατε ότι η Europol πρέπει να είναι κέντρο ανταλλαγής πληροφοριών, ανάλυσης ένα κέντρο υποστήριξης και συνδρομής ε, για συγκεκριμένες πρωτοβουλίες και για το συντονισμό. Θεωρώ ότι είναι η σωστή φιλοσοφία που δεν ε, ε, υπησέρχεται στις αρμοδιότητες των, άλλων, των κρατών μάλλον, απλώς συμπληρώνει και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της δράσης τους. Η έκκληση που απευθύνατε για την αύξηση των χρηματοδοτικών μέσων με βρίσκει απολύτω σύμφωνο. Και εγώ συμμετέχω στην Επιτροπή Προπολογισμών. Ήδη πήρε το λόγο ο συνάδελφο από το ΕΛΚ και νομίζω ότι ε, εάν ενώσουμε τι δυνάμει μα, η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ και η Επιτροπή Προπολογισμών, θα ε, πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Γιατί δεν ήταν σωστή αντιμετώπιση ε, που σας επιφύλαξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως προς αυτό. Δύο ερωτήματα τώρα που προκύπτουν από το έργο που κάνουμε στην Ειδική Επιτροπή για Τρομοκρατία. Δημοκρατία. Κατά τη διάρκεια συναντήσεων που είχαμε με τις αστυνομικές αρχές στα κράτη-μέλη, μίλησαν για τους κινδύνους που ενέχει η κρυπτογράφηση των δεδομένων αυτή τη στιγμή. Αυτό έχει να κάνει ε, με τι δυνατότητε που υπάρχουν για την αποκρυπτογράφηση. Τι κάνετε σε αυτόν τον τομέα και αν υπάρχει συνεργασία με τα κρατημέλη. Δεύτερον, ένα από τα μεγάλα δράματα που αποστροποιεί και ένα τμήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι τα όσα ε, συμβαίνουν στην Μεσόγειο και ε, την ε, διακίνηση σε αυτόν τον τομέα λοιπόν που έχει επιπτώσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ενεργό ρόλο να δυναματίσει η Europol. Τι κάνατε ακριβώς ε, λοιπόν για να καταπολεμήσετε την διακίνηση ανθρώπων, να καταπολεμήσετε και τους διακινητές και ποια είναι η κατανομή ε, του άχθου σε σχέση και με την Frontex. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Ντεμπόλα, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Να ξεκινήσω απαντώντας τον κύριο Δίας Δεμέρα. Σας ευχαριστώ που υποστηρίζετε τις προτεραιότητες και τους στόχους της Europol. Έχουμε προβλήματα πληροφορικής, όντως. Τα τελευταία χρόνια, λόγω των τρομοκρατικών επιθέσεων και, των, και της διακίνησης λαθρομεταναστών, ενισχύσαμε το Κέντρο Αντιτρομοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το Κέντρο ε, Καταπολέμησης της Λαθρομετανάστευσης. Ε, αλλά επειδή έχουμε περιορισμένο προϋπολογισμό, χρειάστηκε να υποβαθμίσουμε σε προτεραιότητα την πληροφορική μας και το τμήμα πληροφορικής. Όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για την τεχνική υποστήριξη και γιατί η Europol είναι ένα κέντρο ενημέρωσης και θα πρέπει να λαμβάνει πληροφορίες, να μοιράζεται και να επεξεργάζεται τις πληροφορίες και επομένως θα πρέπει να είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο στον τομέα της πληροφορικής. Τι χρειαζόμαστε, επομένως χρειαζόμαστε πόρους για να αναπτύσσουμε συστήματα πληροφορική για να μπορούμε να βοηθάμε όπως πρέπει τα κράτη-μέλη. Η τεχνολογία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για μας. Η συνεργασία με τον ε, γενικό επόπτη αυτό προστασία δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είχαμε την πρώτη συνάντηση με τον επόπτη της Βουλγαρίας όταν ήμουν παρατηρήτρια και εν συνεχεία ε, ήρθε στην ε, ο Γενικός Επόπτης Προστασίας Δεδομένων ήρθε στο, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου μας ως παρατηρητής. Ε, νομίζω υπάρχει, έχει νόημα να υπάρχει και μια πολιτική παρακολούθηση του, της Europol και να έχουμε στενότερες σχέσεις με, τις εθνικές, με τα εθνικά και ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και οι συμβουλές σας ε, τις θεωρώ κατευθυντρίες γραμμές για το μέλλον της Europol. Είμαι έτοιμη να απαντήσω και σε ερωτήσεις ε, και για θέματα προστασίας δεδομένων. Ε, ελπίζω το Σεπτέμβριο να συζητήσουμε τέτοια θέματα οι συμφωνίε οι επιχειρησιακέ συμφωνίες με τρίτε χώρε είναι πάρα πολύ σημαντικέ ε, για την Europol, γιατί δεν έχουμε επιχειρησιακέ συμφωνίε με τρίτε χώρε τώρα και υπάρχει σαφή σχέση ανάμεσα στην ε, εξωτερική διάσταση τη ασφάλεια και την εσωτερική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επομένω πρέπει να συνεργαζόμαστε με τρίτε χώρε. και είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο να καθοδηγεί την Κομισιόν και να συμφωνεί με τις εξέλιξεις στον τομέα αυτό, γιατί θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι μπορούμε να προβλέψουμε και ότι έχουμε στη διάθεσή μας τις ε, πιο ακριβείς πληροφορίες, ούτω ώστε να δώσουμε απαντήσεις ε, στις απειλές που αφορούν την ασφάλεια στην Ένωση. Κυρία Η Ευρωπαϊκή Μονάδα Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών. Το θέμα της Μάλτας επίσης και της ε, Σλοβακίας τα κέντρα, για τα κρυπτονομίσματα ε, με την Ιρλανδία. Σε αυτό το τομέα, όχι μόνο η Ιρλανδία, πολλά άλλα κρατημέλη ζητούν ε, την ε, ενίσχυση της Europol για να τις βοηθήσουμε στις έρευνες για κατάρτιση, για να εντοπίσουμε τις απειλές και, για, και ζητούν, ας πούμε, κατάρτιση για αστυνομικούς ε, και για εισαγγελεί. γιατί ε, έχουμε πρόβλημα με πλαστή χρήση, προβληματική χρήση των ε, κρυπτονομισμάτων. Ε, υπάρχει μια ετοιμότητα στα κράτη-μέλη και γι' αυτό ακριβώ έκανα μια συζήτηση με το Γενικό Διευθυντή τη ΣΥΠΟΛ για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί για το θέμα τη κατάρτιση. Γιατί εάν πρέπει να προβλέψουμε κατάρτιση σε επίπεδο Europol, αυτό σημαίνει ότι υποστηρίζουμε λιγότερο τι έρευνε, τι επιχειρησιακέ έρευνε. Ε, Το κέντρο ε, ευρωεγκλήματος, του ευρωεγκλήματος, έχει μεγάλη πραγματογνωμοσύνη για τα κρυπτονομίσματα, έχουμε πραγματογνώμονες, ε, τους, ε, έχουν πολύ φόρτο εργασία, προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε, καταρτίζουμε αξιωματούχους ε, στα κράτη-μέλη αυτή τη στιγμή, μαζί και μαζί με τα κράτη-μέλη έχουμε δεσμευτεί, ειδικά κάποια κράτη-μέλη που έχουν ε, ειδικού να δουλέψουμε σε δίκτυο ε, ούτως ώστε να ανταλλάξουμε αυτή την, ε, επιμεριστούμε αυτή την ε, πραγματογνωμοσύνη και να υποστηρίξουμε τις έρευνες στα κράτη-μέλη για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα των κρυπτονομισμάτων. Πρέπει να γίνει πρόοδος. Για τη Μάλτα και τη Σλοβακία. Θα απαντήσω αργότερα σε αυτές τις ερωτήσεις. Για την ε, μονάδα χρηματοπιστωτικών πληροφοριών. Υπάρχει στενή συνεργασία, στενή συνεργασία με τις διοκτικές αρχές και με τις εθνικές ομάδες. Έχουμε επιχειριακές ε, έρευνες, έχουμε πραγματογνωμοσύνη και έχουμε και μια διάσκεψη σε επίπεδο Europol, ή διασκέψεις μάλλον, για το θέμα αυτό. Παρ' όλα αυτά πρέπει να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος και το ξέρουμε αυτό. Πρέπει να δημιουργηθεί μια συνείδηση είναι το, πιο, το, πιο, το δεύτερο πιο σημαντικό πράγμα σε μία έρευνα αυτό. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε τα απαραίτητα βήματα για να σημειωθεί αυτή η πρόοδος. Κύριε Μακοβέη, σας ευχαριστώ για τα συγχαρητήριά σας για τον προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός που προτείνεται έχει κενά, είναι ανεπαρκής. Ο προτινόμενο προπολογισμό επηρεάζει τι ε, συνεχιζόμενε δραστηριότητε. Η ανάπτυξη, ε, παραδείγματο χάρη εξωματικών προσκεκλημένων στα hotspot, ε, διατήρηση πλατφορμών για αποκρυπτογράφηση που θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσω τροποποιητικού προπολογισμού το 2018. Ε, ε, το 2018 λάβαμε 500 εκατομμύρια για τις πλατφόρμες αυτές αποκρυπτογράφησης, αλλά αυτό δεν προβλέπεται για τον προϋπολογισμό του 19 αυτά τα λεφτά. Επομένως δεν θα μπορέσουμε να συντηρήσουμε αυτές τις ε, πλατφόρμες αποκρυπτογράφησης. Επίσης, 26 επιπλέον ε, ε, άτομα που προσλάβαμε το 18, ε, συν 5 νέους συμβασιούχους και το κόστος του πολιετούς ε, χάρτη, οδικού χάρτη της Europol. Ε, έχουμε αιτήματα σε πολλούς τομείς. Θέλουμε περισσότερη Europol, ε, όχι λιγότερη, το λένε πολλοί, για να, για να υποστηρίξουμε τα κράτη-μέλη στις ερευνές τους. Το ζητάνε αυτό. Το να, δια, το να διαλύουμε δίκτυα λαθρεμπόρων, ας πούμε μας ζητάνε την υποστήριξη σε όλες τις χώρες γι' αυτό. Ε, θα πρέπει να εξυπηρετούμε όλο και περισσότερες διοκτικές αρχές και αρχές επιβολής του νόμου. Όταν πηγαίνω στα διάφορα κράτη-μέλη, ακόμα και τα τελωνία ζητούν περισσότερη συνεργασία με την Europol και θέλουν μεγαλύτερη εμπλοκή ε, τα κράτη-μέλη στον τρόπο λειτουργίας της Europol. Ε, θέλουν να στείλουν και αξιωματούχους συνδέσμου και να ανταλλάξουμε περισσότερε πληροφορίε με την Europol. Έχουμε όλο και περισσότερε επιχειρήσει. Και προβλέπουμε, ε, είδαμε αύξηση το τελευταίο χρόνο. Και θα πρέπει να δούμε ποιε είναι οι προτεραιότητέ μα και πού θα βοηθήσουμε τι έρευνε των κρατών μελών. Ε, σε πολύ περίπλοκες και πολύ ευαίσθητες ε, έρευνες έχουμε μειώσει την ε, συμμετοχή μας ή μάλλον την έχουμε αυξήσει ε, όπω στη Μάλτα και στη Σλοβακία και θα έχουμε όλο και περισσότερε αιτήσει τέτοιε ε, στο μέλλον. Θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη αναλυτική στήριξη ε, και ποιοτική ανατολική στήριξη, γιατί τα κράτη-μέλη ε, δεν μπορούν να επενδύσουν και τη χρειάζονται παρόλα αυτά τη στήριξη, ούτω ώστε για να, για να μπορούν ας πούμε, για τι έρευνέ του να έχουν την εικόνα της Ευρώπης. Επίσης, η διαλειτουργικότητα. Χρειάζεται περισσότερου πόρου. και θέλουμε να αναπτύξουμε νέες υπηρεσίες όπως ε, κλιματολογικά εργαλεία, τα οποία είναι πάρα πολύ ας πούμε, ακριβά για τα κράτη-μέλη. Ε, οι συγκεκριμένε επιπτώσει για το 2019 αν το σχέδιο προϋπολογισμού που υιοθετήθηκε από το ε, Διοικητικό Συμβούλιο το Φεβρουάριο φέτος ε, δεν διατεθεί, τότε θα υπάρχει πρόβλημα για την ε, πρόβλημα ε, στα hot spot τα μεταναστευτικά. Θα υπάρχει πρόβλημα για να αναπτύξουμε νέε στατιστικές, νέα εργαλεία για να καταπολεμήσουμε την ε, εγκληματικότητα στα κρυπτονομίσματα. Έχουμε μια μικρή νομική ομάδα που ασχολείται με αυτά, αλλά βλέπουμε ότι τα αιτήματα είναι τεράστια. Η ανάπτυξη συστημάτων που επιτρέπουν άμεση πρόσβαση σε ορισμένα δεδομένα τη Europol για χιλιάδε ερευνητέ. και εγκληματική ανάλυση, ανάλυση μάλλον εγκλημάτων στα κράτη-μέλη. Επίση, θα πρέπει να καινοτομήσουμε και να έχουμε ε, διελειτουργικέ τεχνικέ λύσει για την επεξεργασία ε, των πληροφοριών που αφορούν ε, τι μετακινήσει, τα ταξίδια, για να έχουμε καλύτερο έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διασταύρωση τώρα γίνεται αυτόματα πρέπει να γίνεται αυτόματα, ούτω ώστε να είναι εύκολη και να μην ξοδεύουμε λεφτά για τα, τη διασταύρωση δεδομένων που μπορεί να γίνει με αυτοματοποιημένα εργαλεία. Η υποστήριξη των κρατών μελών για να ε, κατεβάσουν το παράνομο τρομοκρατικό περιεχόμενο ε, δίκτυο Atlas ε, που είναι ένα δίκτυο ειδικών υπηρεσιών ε, σε διάφορα κράτη-μέλη ε, και η Europol ζήτησε να αναλάβει στον ιστικό ρόλο αυτού του δικτύου. Μπορούμε να το κάνουμε, αλλά φυσικά και αυτό χρειάζεται πόρους. Επίσης, θα πρέπει να βελτιώσουμε, όπως είπα ήδη, την καταπολέμηση του ξεπλήματος του χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, προωθώντας την ε, συνεργασία μεταξύ των ε, χρηματοπιστωτικών μονάδων πληροφοριών και των διοκτικών αρχών, αλλά μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και η το να παίξουμε το ρόλο ενός κέντρου για την έρευνα και την ανάπτυξη σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε συνεχώς καινοτόμοι και πρέπει να δούμε τι υπάρχει στην αγορά, ε, τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε εμείς, τι χρησιμοποιούν οι εγκληματίες και πώς οι αρχές πρέπει να ανταποκριθούν. Γιατί δεν μπορεί να το κάνει κάθε χώρα από μόνη της. Αν το κάνει από μόνη της, είναι σχεδόν αδύνατο να τα καταφέρει. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Ντεμπόλ. Νομίζω ότι ήταν πολύ ολοκληρωμένε, εξαντλητικέ θα έλεγα οι απαντήσει ε, σας σε όλες τις ερωτήσεις που ακούστηκαν. Διαφωνεί κάποιο. Α, μάλιστα, είχατε κάνει απλώς ένα διαλυματάκι, συγγνώμη. Ε, συνεχίζει η κυρία Ντεμπόλ. Οι επιδόσεις της Ευρωπόλ, λοιπόν, στον τομέα των διερευνήσεων εγκληματικών υποθέσεων στα κράτη-μέλη περιορίζεται βεβαίω από τον κανονισμό που διέπει τη λειτουργία μας. Συζήτησα αυτό το θέμα με τον αστυνομικό διευθυντή της Μάλτας και τον αστυνομικό διευθυντή της ε, Σλοβακίας. Στην αρχή της παροχή της στήριξή μας δεν ήταν εύκολο το προσωπικό τη Ευρωπόλη να γίνει δεκτό. Έγινε όμω αυτή η συζήτηση. Καταφέραμε και ορίσαμε αρμόδιο στην δική μας ε, υπηρεσία που έρχεται σε επαφή με τις τοπικές και εθνικές αρχές και βλέπω πλέον ότι η Ευρωπόλ έχει γίνει αποδεκτή από τις εθνικές αρχές επιβολής του νόμου ως τμήμα της διερεύνησης, των ομάδων διερεύνησης. Επίσης, ε, άνθρωποι που δουλεύουν για την Ευρωπόλ μπορούν πλέον να καταθέσουν, να καταθέσουν στο δικαστήριο. Εμείς δυστυχώ, ω Ευρωπόλ δεν βεβαίως ε, διαθέτουμε ε, μέτρα καταναγκασμού. Αποτελούμε απλώς τμήμα της ομάδας διερεύνησης και βεβαίως υπαγόμαστε στη δικαστική και αστυνομική δύναμη την οποία συνδράμουμε. Θα υπάρξει βεβαίως και μια σχετική συνάντηση τον Ιούλιο. Ε, όπως ε, ξέρετε, οι υπάλληλοι της Ευρωπόλ θα σας δώσουν περισσότερες πληροφορίες, αλλά μπορώ να σας απαντήσω από τώρα ότι ε, τηλέφωνα και τηλεφωνικές συνδιαλέξεις δεν έχουμε ερευνήσει στη Σλοβακία. Για τα τρία πολύ συγκεκριμένα ερωτήματα που μας θέσατε κύριε, επειδή έχω μόνο δύο λεπτά στη διάθεσή μου, θα πρότεινα να σας αποστείλω μια πιο ολοκληρωμένη απάντηση, αλλά γραπτός, όχι τώρα. Και κύριε Ντεπρέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το ερώτημα καταρχάς. Θα σας απαντήσω και εσάς, αν δεν έχετε αντίρρηση, ε, γραπτή απάντηση στο ερώτημά σας. Έχετε το λόγο, λέει ο Πρόεδρος, κυρία Η κυρία Ιντβελτ. Επειδή έκανα και ένα δεύτερο ερώτημα σχετικά με την ε, κοινοποίηση πληροφοριών στο πλαίσιο προβλημάτων που υπάρχουν στην εφαρμογή του κράτους δικαίου σε διάφορα κράτη-μέλη και νομίζω ότι είναι σαφές σε ποια αναφέρομαι. Μπορείτε να απαντήσετε σε αυτό το ερώτημά μου ε, επίσης γραπτός. Κυρία Ντεμπόλα απαντά ότι ναι, μπορεί. Πρόεδρος, νομίζω ότι καλύψαμε όλα τα θέματα και όλα όσα δεν απαντήθηκαν, εν πάση περιπτώσει, θα απαντηθούν γραπτός. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη για την ε, παρεξήγηση πριν από δύο λεπτά. Νόμιζα ότι είχε ολοκληρώσει τις απαντήσεις της ε, κυρία Ντεμπόλ. Εγώ φταίω. Πάντως, βλέπετε και από τις ερωτήσεις που σας έθεσαν οι συνάδελφοι ότι είναι πολύ ισχυρή η στήριξη που παρέχουν τα μέλη της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ προς εσάς, ιδίως ως προς την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων για τη λειτουργία σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε επιτυχία στο έργο σας. Σας ευχόμαστε. Now we can move to... Ωραία. Μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 5 της ημέρης σας διάταξης. Πλήρης εφαρμογή των διατάξεων του κεκτημένου Σέγγεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία κατάργηση ελέγχων στα εσωτερικά χερσαία, θαλάσσια και εναέρια σύνορα. Στη βάση αιτήματο των σοσιαλιστών τον Απρίλιο, οι συντονιστέ τη ΛΥΜΠΕ αποφάσισαν να συνταχθεί ε, γνωμοδότηση έκθεση ίδια πρωτοβουλία όσον αφορά την εφαρμογή του κεκτημένου Σέγγεν στη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Ως εισηγητή, υπενθυμίζω ότι έχουν περάσει 7 χρόνια από τότε που οι δύο αυτές χώρες έχουν εκπληρώσει όλα τα κριτήρια για να ενταχθούν πλήρως στον χώρο Σέγγεν, όμως η πολιτική απόφαση μπλοκάρεται στο Συμβούλιο έκτοτε. Η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν όλες τις υποχρεώσεις κράτους μέλους του χώρου Σέγγεν, όμως οι πολίτες των δύο αυτών χωρών εξακολουθούν να μην ε, απολαμβάνουν ε, ελεύθερη κυκλοφορία από και προς τις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι δύο χώρες αυτές είναι σαφές ότι ε, συμβάλλουν τα μάλα στην εσωτερική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς γιατί βρίσκονται στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης Παρ' αυτά όμως δεν έχουν γίνει δεκτές στον χώρο Σέγγεν ως πλήρη μέλη για πολιτικούς λόγους. Έχει συζητηθεί το θέμα αυτό πολλά και εδώ στην Επιτροπή μας στην Ολομέλεια καθώς και στο πλαίσιο της σχετικής απόφασης που εγκρίθηκε το Μάιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε πολλές περιπτώσεις λοιπόν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει θέσει την ξεκάθαρη ε, στάση του και στο πλαίσιο αυτό λοιπόν εντάσσεται και αυτή η έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας με την οποία καλείται το Συμβούλιο να λάβει επιτέλους την απόφαση προκειμένου μέσω ε, ενιαίας εκτελεστικής πράξης, νομοθετικής πράξης να εντάξει τις δύο αυτές χώρες. Θέλω να σας πω δύο λόγια για το υπόβαθρο. Το 2010 λοιπόν το Συμβούλιο πρότεινε ε, ε, την πλήρη προσχώρηση των ε, δύο αυτών χωρών στο χώρο Σέγγιν. Δεν υπήρξε συμφωνία τότε. Η Πολωνική Προεδρία τότε ε, πρότεινε μια συμβαστική πρόταση για τα ενιαέρια και τα θαλάσσια σύνορα, αναβάλλοντας όμως τα χερσαία σύνορα. Αλλά ακόμη και αυτή η απόφαση δεν έχει ληφθεί εδώ και 7 χρόνια, από το 2011, κάτι τελείως απαράδεκτο. Αν λάβει κανείς υπόψη του τις αξίες και τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεπίπεδη λοιπόν αυτή η διτή στάση που εμφανίζεται απέναντι στην ε, ε, Βουλγαρία και τη Ρωμανία ενέχει και ε, προϋποθέσεις και κινδύνους ακριβώς γιατί προβλέπονται επιπλέον κριτήρια για δύο κράτη-μέλη κατά ε, παράβαση των όσων ισχύουν για τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και με αυτόν τον τρόπο επίσης δημιουργούνται και ελλείψεις και χάσματα όσον αφορά την ενημέρωση και τη διακίνηση πληροφοριών, την ανταλλαγή πληροφοριών που ε, διακινούνται μεταξύ κρατών μελών που συμμετέχουν και κρατών μελών που δεν συμμετέχουν στον χώρο Σέγγεν. Γι' αυτό λοιπόν και καλούμε ε, να, ε, να, υπάρξει επιμονή ε, και επιβεβαίωση της απόφασης για την προσχώρηση των δύο αυτών χωρών στο χώρο Σέγγεν που είναι εξαιρετικά σημαντικές για ολόκληρο το χώρο Σέγγεν. Και όπως γνωρίζετε στον στην πρόσφατη έκθεση αξιολόγηση για τη λειτουργία του χώρου Σέγγεν που δημοσιεύθηκε, ε, λαμβάνονται και ε, τονίζονται μάλλον διάφορα, διάφορες ελλείψεις και προβλήματα που υπάρχουν προς τον, ε, λειτουργία, τη λειτουργία αυτού του χώρου. Ε, γι' αυτό και λοιπόν συντάξαμε αυτή την έκθεση. Προθεσμία για την, κατα... για την κατάθεση τροπολογιών είναι η 23η Ιουλίου. Σας παρακαλώ να τι υποβάλλετε. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στου σκιώδει ηγητέ. μα. ξεκινώντας από τον κύριο Κοέλιο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως ε, με όλα όσα είπατε. Το Κοινοβούλιο όχι επειδή το Κοινοβούλιο λοιπόν ε, στήριξε αυτή τη θέση εδώ και πολλά χρόνια όπως είπατε, αλλά επειδή έχουμε δίκιο. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για να δώσουμε το καθεστώς του πλήρους μέλους ε, της ζώνης Ένγεν ε, σε αυτές τις δύο χώρες. Το πρώτο βήμα είναι η τήρηση των κανόνων. Θεσπίσαμε λοιπόν κανόνες που λένε ότι κάθε κράτος μέλος που πληρεί τις ε, προϋποθέσεις θα πρέπει ε, να συμπεριλαμβάνεται στη ζώνη Σένγκεν. Και όχι μόνο ως προς το Κοινοβούλιο, αλλά και ως προς τα κρατημέλη, τεχνικές δηλαδή ομάδες. Από όλα τα κρατημέλη ε, είχαν διαπιστώσει και συμφωνήσει ότι και οι δύο αυτές χώρες πληρούν ε, τις περιποθέσεις. Αν θέλουμε λοιπόν να ακολουθήσουμε τους ε, κανόνες και να επιβάλλουμε κυρώσεις στις ε, χώρες που δεν ακολουθούν τους κανόνες, τότε θα πρέπει να προβλέπεται και η πλήρης προσχώρηση των χώρων που πληρούν τις προϋποθέσεις. Μετά, το μήνυμα που αποστέλουμε το να μην είναι κανείς πλήρες μέλος ε, της δεν δίνει την ε, εντύπωση στους πολίτες αυτών των δύο χωρών ότι είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας και ότι δεν χαίρουν των ίδιων δικαιωμάτων με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους πολίτες. Αν πιστεύουμε λοιπόν πραγματικά στην ευρωπαϊκή ηθαγένεια πρέπει να δώσουμε και σε αυτούς τους πολίτες το ίδιο καθεστώς. Τέλος, Πρόεδρε. Αν με ρωτήσατε τι μπορούμε να συναγάγουμε ως δίδαγμα από αυτή τη ε, διαδικασία, πρέπει, θεωρώ, να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι είναι λανθασμένη, κακή η ομοφωνία σε αυτούς τους τομείς πολιτικής, γιατί έτσι ε, οι εθνικές, τα εθνικά πολιτικά συμφέροντα κρατάνε όμοιρο τις πολιτικές αποφάσεις. Πρέπει λοιπόν να αγωνιστούμε για μια ευρωπαϊκή επίλυση αυτών των θεμάτων. Μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας, σε πολλά ζητήματα της αρμοδιότητας της Επιτροπής μας έχουμε να κάνουμε με τη συναπόφαση. Από πλευρά Συμβουλίου έχουμε ειδική πλειοψηφία και όχι ομοφωνία. Ξέρουμε ότι στο συγκεκριμένο θέμα, για το συγκεκριμένο φάκελο υπάρχει ε, προϋπόθεση ομοφωνίας, όμως βλέπουμε ότι αυτό δεν είναι η σωστή λύση και βλέπουμε και το αποτέλεσμα, ότι το συζητούμε ακόμα αυτό το θέμα μετά από 7 χρόνια. Ευχαριστούμε τον κύριο Κοέλιο. Η κυρία Βεχζιά. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και κύριε εισηγητά παράλληλα. Θα είμαι σύντομη γιατί συμμερίζομαι απολύτως τα όσα είπατε και τα όσα είπε ο κύριος Κοέλιο. Για την πολιτική μας ομάδα δεν υπάρχει κανένας λόγος η Βουλγαρία και η Ρουμανία να μην είναι πλήρη μέλη του χώρου Σέγγεν. Όπως είπατε, αυτές οι δύο χώρες τηρούν τις νομικές προϋποθέσεις εδώ και 7 χρόνια, οπότε το μπλοκάρισμα αυτό είναι καθαρά πολιτικό. Ε, η προσέγγιση που δεν έχει καμία νομική βάση, όπως επίσης υπόθηκε. Και μάλιστα αφορά τα χερσαία σύνορα, αυτά που είναι ε, πιο κοντά στους, Ευρωπαίου στους Ευρωπαίους πολίτες. Και αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο το αίσθημα αδικίας που νιώθουν ε, οι Βούλγαροι και Ρουμάνοι υπήκοοι αλλά και οι, ε, όσοι εργάζονται διασυνοριακά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι βούτυρο στο ψωμί του λαϊκισμού και του ευρωσκεπτικισμού και αντιευρωπαϊσμού. Σας ευχαριστώ που στείλατε ε, τόσο έγκαιρα της, ε, το προσχέδιο τροπολογιών και μάλιστα νομίζω ότι θα υποβάλουμε καν τροπολογίες γιατί δεν έχουμε και πολλά να πούμε σε αντίθεση ε, με όλα αυτά που πολύ σωστά μας ε, περιγράψατε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάμοφ. Αντάμοφ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σα συγχαίρω για την εκπόνηση αυτή τη έκθεση. Έχετε την αμέριστη στήριξή μου. Για άλλη μια φορά προσπαθούμε να ζητήσουμε από το Συμβούλιο να πάρει μια απόφαση για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Στην Ευρώπη γίνεται λόγος για αλληλεγγύη, για δικαιοσύνη, όμως με το να μην γίνεται δεκτή η Βουλγαρία και η Ρουμανία στη ζώνη Σέγγεν, αυτό αποτελεί απόδειξη ενός ελλείμματος ε, δικαιοσύνης. Οι δύο αυτές χώρες τηρούν ε, και πληρούν τα κριτήρια από το 2011. Όμως δεν ε, είναι πλήρη μέλη της ζώνης έγκυνη και αυτό είναι μια ταπείνωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλούμε για την ε, πρωτοκαθεδρία του δικαίου. Ορισμένα κράτη-μέλη, για ορισμένα κράτη-μέλη ακολουθείται δικαστική διαδικασία, όμως κράτη-μέλη υπάρχουν επίσης που δεν τηρούν το δίκαιό τους. Επομένως, για ποιο δίκαιο μιλάμε Τη κυριαρχία του νόμου. Τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την προσχώρηση στη ζώνη Σέγγεν πληρούνται από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, όμως δεν έχουν γίνει ακόμα πλήρη μέλη. Κάποια κρατημέλη ζητούν ε, διαδικασία σε δύο στάδια για την προσχώρηση των δύο χωρών. Πρώτο, μας λένε ότι πρέπει ε, να ανασταλούν οι έλεγχοι στα σύνορα, τα εναέρια και τα θαλάσσια και μετά στα χερσαία. Αυτό θα ενοποιήσει όμως την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ νομίζω ότι είναι μια κακή πρακτική που ε, τροφοδοτεί και ενισχύει τον ευρωσκεπτικισμό ε, και τον εθνικισμό. Γι' αυτό η Βουλγαρία και η Ρουμανία θα πρέπει να γίνουν πλήρη μέλη της ζώνης Σιάνγκεν. Ελπίζω η Κροατία να μην έχει τα ίδια προβλήματα. Ευχαριστώ κύριε Πίτσουλα. Και μετά κύριε Μάκοβεϊ. Ευχαριστώ. Σας συγχαίρω που κάνετε μια θαυμάσια, που κάνετε μια θαυμάσια έκθεση. Σήμερα ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελεύθερη κυκλοφορία είναι μία από τις πιο σημαντικές ελευθερίες, αλλά θυσιάζεται για την ενίσχυση, στο βωμό της ενίσχυσης των συνόρων. Αυτό γίνεται για να αντισταθμίσουμε τις ελλείψεις άλλων πολιτικών όσο διαφορά το κοινό σύστημα ασύλου και τη μεταρρύθμιση του Δουβλίνου. Ο μόνος τρόπος που μπορούμε να προστατεύσουμε το επίτευγμα μας είναι αυτό, ε, είναι να ενισχύσουμε το στοιχείο αυτό. Σας, βάζω που βάλατε, σας ευχαριστώ που βάλετε και την Κροατία στην έκθεσή σας. Ε, όταν εφαρμόζουμε ε, επιτυχώς το, χρησιμοποιούμε το ΣΥΣ επιτυχώς και το κάνουμε ε, από πέρυσι, ε, μας βοηθάει πάρα πολύ. Και μάλιστα σε, σε λίγες εβδομάδες τα εναπομείναντα κριτήρια θα πληρούνται. Επίσης, μερικές λύσεις δεν είναι αποδεκτές μόνο πλήρης προσχώρηση με βάση αξιολογικά κριτήρια είναι ο μόνος τρόπος για να ενισχύσουμε το Σέγγεν και επομένως να ενισχύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Οικοδόμημα. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέη είναι η επόμενη ομιλήτρια. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω ρουμάνικα, την μητρική μου γλώσσα δηλαδή η αξιολόγηση έχει ολοκληρωθεί για τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία και για την προσχώρησή τους στο Σέγγεν. Και αυτό επιβεβαιώθηκε και από το Συμβούλιο του 2018. Η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο επιβεβαίωσαν το 2017 και το 2018 ε, ότι τεχνικά είναι έτοιμη και η Βουλγαρία και η Ρουμανία για να ενταχθεί στο Σέγγεν. Και επίσης στις 2 Ιουλίου του 2018 το πολιτικό ε, ε, δημοσίευσε μία απόφαση για να αρθούν τα τελευταία ε, εμπόδια στο κεκτημένο Σέγγεν από την Βουλγαρία και Ρουμανία. Η επίσημη εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηλαδή. Εγώ ήμουν εισηγήτρια για αυτή την έκθεση για την άρση των τελευταίων εμποδίων σε ό,τι αφορά την ε, εφαρμογή του κοινοτικού κεκτημένου τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Φυσικά και θέλω να ενταχθεί η χώρα μου στο Σέγγεν, αλλά θέλω να κάνω το εξή σχόλιο. Η Κομισιόν δεν, ε, συνέδεσε την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας με, την, με το Μηχανισμό Συνεργασίας και Επαλήθευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτές τις δύο χώρες. Επομένως, Αντίστοιχα, δεν θα πρέπει να συνδέσουμε το μηχανισμό αυτό ε, με τις προϋποθέσεις της έκθεσης αυτής. Γιατί ο μηχανισμός θα πρέπει να εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την υλοποίηση όλων των κριτηρίων που αναφέρονται εκεί. Και το λέω αυτό γιατί στη Ρουμανία υπάρχει μια φοβερή μάχη που μένεται κάθε μέρα εναντίον της ε, διαφθοράς. Και αυτό είναι ε, η κακή επίπτωση μιας ε, επιτυχούς προσπάθειας ε, καταπολέμησης διαφθοράς. Ε, σήμερα το πρωί έχασε το αξιωμά, έχασε το της ε, η υπεύθυνη για την καταπολέμηση της διαφθοράς, του, του φορέα δηλαδή για την καταπολέμηση της διαφθοράς, γιατί έδωσε μια συνέντευξη στο Euronews. Ε, οι πολιτικοί και η κυβέρνηση δεν θέλουν να επαληθεύονται, δεν θέλουν να ελέγχονται. Ε, όχι, χρειαζόμαστε το μηχανισμό συνεργασίας και επαλήθευσης και περιμένουμε την ε, επόμενη έκθεση. Ευχαριστώ κυρία Μέλοβα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για τη δουλειά που κάνετε στην έκθεση αυτή. Όπως είπε και ο κύριος Κοέγιο, από το 2011 η Βουλγαρία και η Ρουμανία πληρούν τα κριτήρια για την ε, προσχώρηση στο, Σέγγεν, στο χώρο Σέγγεν. Η άδικη στάση ε, απέντη στη χώρα μας εδώ και χρόνια με με θλίβει και χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους θα μπει ένα τέλος σε αυτήν την κατάσταση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε πάντα στεναριστάσει ότι οι κανόνες δηλαδή θα πρέπει να εφαρμόζονται με ισότιμο τρόπο και δίκαιο τρόπο για όλους. Και ευχαριστώ τον συνάδελφο ή τους συναδέλφους για την υποστήριξή τους. Τα εμπόδια για την ένταξή μας στο Σέγγεν είναι καθαρά πολιτικά. Δεδομένων της ε, μεταναστευτικής κρίσης, θα ήθελα να σας πω ότι η Βουλγαρία συνεισφέρει κατά προτεραιότητα στον έλεγχο και στην ε, ανάσχεση των μεταναστευτικών ροών. Ε, επενδύουμε πάρα πολύ, μπορούμε να συνεισφέρουμε στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Μας υποστηρίζει η Ευρωπαϊκή Ακτοφυλακή και Συνοριαφυλακή επίσης. Εάν η έλεγχη στα εσωτερικά σύνορα Βουλγαρίας και Ρουμανίας καταργηθούν, τότε τα μέσα τα οποία δαπανώνται για τους εσωτερικούς ελέγχους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στα εξωτερικά σύνορα. Εκεί όπου έχουμε και περισσότερο ανάγκη από αυτούς τους πόρους. σορισμενα κρατη κράτη-μέλη, οι Βούλγαροι και οι Ρουμάνοι ελέγχονται επιπλέον Μερικέ φορέ ελέγχονται επιπλέον και οι αποσκευέ του. Και αυτό είναι άδικο απέναντι στου Βούλγαρου και στου Ρουμάνου. Ε, ε Επίση, πρέπει να προσθέσουμε και τι οικονομικέ συνέπειε όλα αυτά. Μία έρευνα του 2016 αξιολόγησε το κόστος ε, επανεισαγωγή των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα ε, σε επίπεδο 20 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και Μιλάμε για 2 μέχρι 4 ε, δισεκατομμύρια για τα λειτουργικά έξοδα. Γι' αυτό θα πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε το Συμβούλιο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πάβελ. Καταρχά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την έκθεσή σας και να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την στεναρή τους και συστηματική τους υποστήριξη στην προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν. Είναι πολύ σημαντικό να ασκηθεί πίεση στο Συμβούλιο προκειμένου να αρθεί αυτή η αδικία απέναντι στους πολίτες μας. Ορθώς είπατε ότι όλα τα τεχνικά κριτήρια ε, πληρούνται εδώ και πολλά χρόνια. Έχουμε δημοσιεύσει, ε, επενδύσει ε, χρήματα των Βουλγάρων και Ρουμάνων φορολογουμένων για να εξασφαλίσουμε και να προστατεύσουμε τα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης. Η απόφαση της Συνόδου ΔΕΗ, του Συμβουλίου ΔΕΗ ε, ε, είναι πραγματικά ε, απαράδεκτη. Πρόκειται περί ζητήματος που αφορά την υλοποίηση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια σε αυτό που γίνεται στο Συμβούλιο πρέπει να επιδείξουμε στεναρή στάση ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας καλώ λοιπόν ε, ε, συνάδελφοι να μην υποβάλλετε τροπολογίες σε αυτή την έκθεση, να μην επιτρέψουμε ε, από την πλευρά μας την εισαγωγή δύο σταδίων για την προσχώρηση. Δεν είναι δυνατόν να προστίθενται όλο ένα και περισσότερα κριτήρια για την προσχώρηση αυτών των δύο ευρωπαϊκών χωρών στο χώρο Σέγγεν. Έρχεται σε αντίθεση με τις ευρωπαϊκές αξίες. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα για την ανάκληση ε, του ε, διευθυντή ε, της Αρχής για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς. Μιας όμως και αναφέρθηκε το θέμα, πρέπει να σας πω ότι έχει συνταχθεί έκθεση 35 σελίδων συγκεκριμένα, ε, όπου αιτιολογείται η απόφαση αυτή. Υπάρχουν και κάποια απόρριτα έγγραφα, τα οποία δεν είναι δημοσιεύσιμα, και τα οποία ε, επίσης ε, αιτιολογούν την ε, ανάκληση αυτή. Μην ακούτε τώρα τι λέει το Euronews. Υπήρξαν παρατυπίες σοβαρότατες και προβλήματα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του και γι' αυτό έγινε η ανάκληση του συγκεκριμένου ανθρώπου. Σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ όλους για την υποστήριξη ως προς την ουσία αυτής της έκθεσης. Όπως είπε και ο κύριος Κοέλιο και έχει πει συστηματικά στην θητεία του, το Σέγγεν είναι λύση, όχι πρόβλημα. Γι' αυτό και σας ευχαριστώ που με βοηθάτε για να στείλουμε ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο άλλο ένα ισχυρό μήνυμα. Και όπως είπε και η κυρία Μακοβέη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ποτέ δεν συνέδεσε ε, το CVM με την, με την προσχώρηση στο Σέγγεν. Όμως στην πράξη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Εγώ, ε, μάλλον εμείς πρόσφατα ακούσαμε πρωθυπουργό στην Ολομέλεια να λέει κάτι ψευδές για να το θέσω ήπια. Είπε ότι η συμφωνία είναι συμφωνία και πρέπει οι δύο αυτές χώρες να ε, εκπληρώσουν το CVM. Κάτι το οποίο δεν ισχύει. Θέλω λοιπόν να πω το εξή. Αν θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διατηρήσει την αξιοπιστία τη, τότε πραγματικά θα πρέπει η ίδια πρώτα και κύρια να ακολουθεί του κανόνε που η ίδια έχει θέσει. Και αυτό αφορά ε, το Συμβούλιο και την Κομισιόν, βεβαίω, γιατί εμεί ω Κοινοβούλιο έχουμε πολύ συγκεκριμένη και πολύ ξεκάθαρη στάση εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Κυρία Μακοβέη. Πολύ σύντομα κύριε Πρόεδρε. Θέλω να δηλώσω τη στήριξή μου στην έκθεση και θέλω οι δύο αυτές χώρες, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, να προχωρήσουν στο χώρο Σέγγεν. Αυτό το λέμε εδώ και πολλά χρόνια, αλλά πρέπει πραγματικά να απεμπλακεί η διαδικασία από την εφαρμογή του CVM. Αν υπάρχουν προβλήματα διαφθοράς στις δύο αυτές χώρες, ε, τότε αυτά πρέπει να αντιμετωπιστούν. Αλλά δεν μπορεί αυτά τα δύο να συνδέονται με, με κριτήρια καταπολέμησης διαφθοράς. Ναι, το ξέρω, συμφωνούμε, λέει ο πρόεδρο. Απλά είπα ότι ακόμη και πρωθυπουργού έχουμε ακούσει να ισχυρίζονται κάτι τέτοιο. Κύριε Κοέλιο, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να συνδέσουμε την αξιολόγηση περί διαφθοράς με τα κριτήρια Σέγγεν, αν κάτι τέτοιο ίσχυε για όλα τα κράτη-μέλη. Αυτό όμως που δεν γίνεται με τίποτε είναι να εφαρμόζεται μια τέτοια διαδικασία για κάποια κράτη-μέλη και να μην εφαρμόζεται για όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Έχετε πολύ δίκιο, λέει ο Πρόεδρος. Το συντομότερο δυνατό και πριν το Σεπτέμβριο σε κάθε περίπτωση θα ξανασυνεδριάσουμε ισχυριώδης ε, για να ξαναδούμε το θέμα. Σας είπα, ε, προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι 20 Ιουλίου. Λοιπόν, και μπορούμε να περάσουμε στο έκτο θέμα, σημερινή σα διάταξη Έχουμε και προσκεκλημένου, τους οποίους καλωσορίζουμε. Συνάδελφοι, μπορούμε να ξεκινήσουμε νομίζω. Βλέπω ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τους δύο υπουργούς της Αυστριακής Προεδρίας που έχουμε μαζί μας. Να καλωσορίσω τον κύριο Χέρμπερτ Κίκλ, ο οποίος είναι καθοδόν. Βρίσκεται όμως στο κτίριο που είναι Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών τη Αυστρία, καθώ και τον κύριο Γιώζεφ Μόζερ, Ομοσπονδιακό Υπουργό Συνταγματικών Υποθέσεων, Μετακτήσεων, Απορρίθμιση και Δικαιοσύνη τη Αυστρία. Με πολύ μεγάλη μα χαρά σα υποδεχόμαστε εδώ στι Βρυξέλλε, κύριε Υπουργή, για να μα παρουσιάσετε τι προτεραιότητε τη Αυστριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Η Αυστριακή Προεδρία έρχεται σε ένα πολύ κρίσιμο στραβοδρόμι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς βρισκόμαστε στο τελευταίο πλήρες έτος της ε, θητείας της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι είναι ε, ασφαλές να πει κανείς ότι πρόκειται για προεδρία τελευταίας ελπίδας για να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις. Η ΛΥΜΠΕ έχει σημαντική ευθύνη να εξασφαλίσει ότι οι καλές προθέσεις σε κάποια πολύ πιεστικά ζητήματα για τους Ευρωπαίους πολίτες δεν θα παραμείνουν κενό γράμμα. Οι ε, προσδοκίες ε, του Κοινοβουλίου είναι πολύ υψηλές και τώρα η Αυστριακή Προεδρία έχει πλέον την ευκαιρία να ε, αποφέρει τους καρπούς που ε, ε, έχουν, που, έχουν, που αντιστοιχούν στο σκληρό έργο των τελευταίων τεσσάρων ετών. Σε πάρα πολλά ζητήματα, λοιπόν, η Αυστριακή Προεδρία έχει αναλάβει πρωτοβουλίες σε θέματα που μας απασχολούν και μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερως. Αυτό που θέλω όμως να τονίσω είναι ότι μας ενδιαφέρουν πολύ οι ευρωπαϊκές λύσεις και όχι τις κάθε χώρας ξεχωριστά που είναι της μόδας τον τελευταίο καιρό. Αυτό ελπίζουμε να είναι και η γραμμή που θα ακολουθήσει η Προεδρία. Όπως γνωρίζουν οι Υπουργοί, τους τελευταίους μήνες έχει σημειωθεί συμμονητική προόδος όσον αφορά ζητήματα που σχετίζονται με την μετανάστευση, το άσυλο, τις θεωρήσεις, την διαλειτουργικότητα των μηχανογραφικών συστημάτων. Γεια σας κύριε Πρόεδρε, σας καλωσορίζω. Uh, και σε άλλους τομείς βεβαίως που είναι απαραίτητο όπως ε, το ε, πακέτο για το άσυλο όπου ακόμα δεν έχουμε πετύχει από τα αποτελέσματα. Δυστυχώς πριν από δύο εβδομάδες μάλιστα φτάσαμε και σε ένα σημείο που οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έβγαλαν χαρτί και μολύβι και διαμόρφωσαν από κοινού μία διατύπωση ε, εξ ονόματος του Συμβουλίου. Η πλειονότητα των μελών αυτή τη Επιτροπή και αυτού του Κοινοβουλίου θεωρεί ότι υπάρχει διασύνδεση αυτών των ζητημάτων. Γι' αυτό θα ακούσουμε με ενδιαφέρον τη δική σα οπτική γωνία για τα όσα διαμήφθησαν στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στα επόμενα βήματα, αν θεωρείτε ότι πρέπει να διατηρήσουμε τα όσα έχουμε πετύχει και αν είστε διατεθειμένοι να καταβάλλετε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διατηρήσετε αυτή την προσέγγιση της δέσμη του πακέτου. Κατανοώ, κατανοούν μάλλον σίγουρα οι συνάδελφοι από την Αυστριακή Προεδρία το μέγεθος και την κλίμακα της δυσκολίας της πρόκλησης. Θα δώσω πρώτα το λόγο στους, ε, προεδ, στους υπουργούς για την ε, παρουσίασή τους, 10 λεπτά έκαστος και μετά θα δώσουμε το λόγο στα μέλη για την ε, γενική συζήτηση. Πρώτα θα δώσουμε το λόγο στους συντονιστές και μετά στα λοιπά μέλη προτείνω να περιοριστούν τα, μέλη στα δύο λεπτά έκαστος. Παρακαλώ, κύριε Υπουργέ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, αξιότιμη κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη μου χαρά που έχω σήμερα την ευκαιρία να σας παρουσιάσω τις προτεραιότητες της Αυστριακής Προεδρίας στον τομέα της αυστρικής ασφάλειας και που στη συνέχεια θα έχουμε και τη δυνατότητα να συζητήσουμε τα θέματα αυτά. Θεωρώ ότι είμαστε εταίροι και η συνεργασία μα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένα θέμα πολύ σημαντικό για μένα. Και αυτό άλλωστε είναι και ο λόγο που και στο παρελθόν έχω ε, συνομιλήσει με ευρωβουλευτέ, ε, συστηματικέ επαφέ, και αυτό ε, ισχύει ακόμη περισσότερο για του εμπειρογνώμονε που έχω μαζί μου και που με υποστηρίζουν στο έργο μου. Γνωρίζετε ότι η Αυστρία αναλαμβάνει για τρίτη φορά στην ιστορία τη την Προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Κάποιοι ισχυρίζονται ότι έχουμε εμπειρία πλέον. Γνωρίζετε όμως και τον, ε, ε, ε τη ρίση του Ηράκλειτου ότι ένας ποταμός δεν είναι ποτέ ο ίδιος. Υπό αυτές λοιπόν τις συνθήκες Ε, θέλω λοιπόν να σας παρουσιάσω ε, τα προβλήματα που, και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε πολλοί πολίτες ε, έχουν χάσει ένα μεγάλο μέρο τη της ε, εμπιστοσύνη του στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω τη μεταναστευτική κρίση και τη κρίση του ευρώ. Έχουμε λοιπόν ε, μπροστά μα πολύ δύσκολε δημοσιονομικέ διαπραγματεύσει. Νομίζω όμως ότι όλοι έχουμε πλήρη επίγνωση της, μεγάλης, των μεγάλων ευθυνών που έχουμε αναλάβει στους ώμους μας. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να χαράξουν κοινή πορεία για τις ε, δύσκολες ε, προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο μέλλον. Μία είναι η πολύ σημαντική ε, πρόκληση που πρέπει να τύχει της αμέριστη προσοχή μας. Λόγω της ε, μεταναστευτική κρίση του 2015 δημιουργήθηκε ε, σε πολλούς Ευρωπαίους πολίτες η αίσθηση ότι έχει χαθεί ο έλεγχος από τις ελίτ, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από τις κυβερνήσεις. Και αυτό αποτελεί και ένα πλήγμα για την εμπιστοσύνη προς την ε, ικανότητα των κυβερνήσεων, των θεσμικών οργάνων να λάβουν ε, δράσεις, ιδίω όσον αφορά την καταπολέμηση ε, τον, του οργανωμένου εγκλήματος και της διαφθοράς. Γι' αυτό και πρέπει από κοινού να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη των λαών μας. Και γι' αυτό το λόγο θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να εστιαστούμε σε εκείνα τα θέματα στα οποία οι πολίτες μας περιμένουν δικαίως λύσεις από εμάς. Εκεί όπου πραγματικά ε, χτυπά η καρδιά των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι πολίτες μας. Και αυτό είναι και ο λόγος που το σύνθημα της Αυστριακής Προεδρίας ε, που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Προεδρία είναι Ευρώπη που προστατεύει, γιατί η προστασία είναι μια πολύ βασική ανάγκη των ανθρώπων και ε, γι' αυτό το σκοπό έχουμε ε, ορίσει και έξι πολύ συγκεκριμένες προτεραιότητες. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 29ης ε, Ιουνίου 2018 που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικά για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων μας. Εκεί περιλαμβάνονται ουσιώδη θέματα που η Αυστρία εδώ και πολλά χρόνια με άλλα κράτη-μέλη ε, από κοινού συζητά ε, στο πλαίσιο της ε, μελλοντικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρούμε ότι το Συμβούλιο κατάφερε να ξεκινήσει ε, μια μεταστροφή στα ζητήματα ασύλου και μετανάστευσης. Τι σημαίνει αυτό. Αντί να επικεντρωνόμαστε σε ποσοστώσεις και κατανομή προσφύγων, υπάρχει πλέον επικέντρωση στην προστασία και τη διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων, την καταπολέμηση των διακινητών και την ενισχυμένη συνεργασία με τρίτες χώρες. Και υπό αυτές τις προϋποθέσεις ελπίζω και πιστεύω ότι θα διευκολυνθούν, ε, θα διευκολυνθεί και ε, η προώθηση των εσωτερικών πτυχών που σχετίζονται με την μετανάστευση και το άσυλο. Αυτή η μεταστροφή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αποδεικνύεται και στον τομέα ε, των ε, περιφερειακών ε, κέντρων διαχείρισης μεταναστών. Σημαντικό στοιχείο είναι πλέον η προώθηση ε, και η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής Ακτοφυλακής και της Frontex. Αυτό θα βοηθήσει στην ε, ε, διαφύλαξη, τη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων και την επιστροφή παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Γι' αυτό χρειαζόμαστε όμως ενισχυμένη εντολή και ενισχυμένα κονδύλια. Ως Ευρωπαϊκή Προεδρία εμείς ε, είμαστε δεσμευμένοι στη διατήρηση του χώρου Σέγγεν. Όσο όμως υπάρχουν ανεξέλεκτες μεταναστευτικές ροές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέτουν σε κίνδυνο, σε κίνδυνο την ασφάλεια των πολιτών μας, η διενέργεια εσωτερικών ελέγχων θα εξακολουθήσει να είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να δεχόμαστε ως πραγματικότητα. Ως ε, Προεδρία όμως θέλουμε να συμβάλλουμε ε, ώστε κατά το δυνατόν να επιστρέψουμε ε, στο παλαιό καθεστώς του Σέγγεν. Χρειαζόμαστε λοιπόν ένα σύστημα ασύλου και μετανάστευσης το οποίο θα αντιμετωπίζει και θα είναι ε, ισχυρό ακόμα και σε περιπτώσεις κρίσεων. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Γι' αυτό και το έργο μας στον τομέα του Δουμβλίνου και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου αποτελούν πολύ σημαντικές μας προτεραιότητες στο πλαίσιο της συνολικής μας προσέγγισης. Για μια πιθανή λύση λοιπόν όμως ε, χρειάζεται να σημειωθεί πρόοδος στην ε, διαφύλαξη των εξωτερικών σανόρων, στην εξωτερική διάσταση καθώς και ένας νέος ορισμός των όρων ε, αλληλεγγύη και ευθύνη. Εμείς θα καταβάλουμε προσπάθειες τον Οκτώβριο να παρουσιάσουμε πρόοδο στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων. Αυτό βεβαίως θα εξαρτηθεί από όλους μας, τόσο από εσάς όσο και από εμάς, όσο και από την στενή συνεργασία μεταξύ μας ε, όσον αφορά τα σχετικά ε, νομοθετικά εργαλεία. Θέλουμε ο, εξτρεμι, ο εξτρεμισμός και η τρομοκρατία να μην έχουν πού να σταθούν στην Ευρώπη και γι' αυτόν τον σκοπό ε, πρέπει να προωθηθούν ε, οι κοινέ μας αξίες, οι θεμελιώδεις μας αξίες, η ενίσχυση των μέτρων κατά πολέμηση του αντισημιτισμού και η ενίσχυση των μέτρων για την προστασία εβραϊκών κοινοτήτων και ιδρυμάτων. Και στο πλαίσιο αυτό θέλω να σας παραπέμψω και στην υπουργική διάσκεψη που έγινε το Νοέμβριο στη Βιέννη με ε, θέμα ευρωπαϊκές αξίες στην οποία και θα, που, που θα γίνει το Νοέμβριο και στην οποία στη διάσκεψη θα σας ε, καλέσουμε και εσάς. Βεβαίως χρειαζόμαστε και ενισχυμένη αστυνομική συνεργασία καθώς και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των υφιστάμενων ε, εργαλείων μας. Και σε αυτόν τον τομέα ε, θα επικεντρωθούμε και ε, στην ενισχυμένη ε, αστυνομική συνεργασία για τα έτη 2018-2021. Θέλουμε να σπάσουμε την, τον, την διασύνδεση οργανωμένου αγκλήματος και τρομοκρατίας. Θεωρώ ότι είναι προϋπόθεση για μια ένωση ασφαλείας οι ποινικέ μας διαδικασίες καθώς και οι αξιωμετούχοι που, ασχολούνται που απασχολούνται στον τομέα της μετανάστευσης να έχουν στη διάθεσή τους τις απαραίτητες πληροφορίες και εδώ υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης πρόταση της Κομισιόν λοιπόν για την εναρμόνιση των βάσεων δεδομένων είναι υπερόρημη. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα κλείσουν διάφορα χάσματα όσον αφορά την πληροφόρηση και να ε, βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των βάσεων δεδομένων. Βεβαίως αυτό πάντοτε με ε, ταυτόχρονη τήρηση των εγγυήσεων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Και εδώ βεβαίω βασιζόμαστε στην στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ελπίζουμε έω το τέλο τη ε, φετινή χρονιά να καταφέρουμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία. Για την επίτευξη των στόχων μα, ε, ε, απαιτείται και στενή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, με τις χώρες προέλευσης και τις χώρες διέλευσης. Και θα ενισχύσουμε την συνεργασία μας και με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων και θα τους παράσχουμε συνδρομή προκειμένου να εναρμονίσουν τα πρότυπά τους με τα ευρωπαϊκά. Το ίδιο και για τη Βόρεια Αφρική. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο ζήτημα της ασφάλειας και της μετανάστευσης απαιτεί ε, συνεργασία και εναρμόνιση των ευρωπαϊκών προσεγγίσεων. Και αυτό θα συζητηθεί και στην υπουργική διάσκεψη 13 και 14 Σεπτεμβρίου. Θεωρούμε ότι και η επιστροφή ε, ε, και η απέλαση πρέπει να αποτελέσουν ε, εργαλείο στη φαρέτρα μας και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί ανοιχτά. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε ένα πολύ έντονο εξάμεινο μπροστά μας το οποίο θα κρίνει και το, τις, τις κατευθύνσεις που θα πάρει η ευρωπαϊκή πολιτική τα επόμενα χρόνια. Εκεί όπου υπάρχει ε, τρόπος, εκεί που υπάρχει βούληση υπάρχει και τρόπος. Από τη δική μας πλευρά μπορώ να σας εξασφαλίσω ότι βούληση υπάρχει. Αν και εξασφαλιστεί και η δική σας συνεργασία θα υπάρξει και τρόπος. Ευχαριστούμε κύριε Μόζελ, έχετε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ευρωβουλευτές, ακούστηκε ε, από πολλές πλευρές ότι η Αυστρία ε, θέλει να ανταποκριθεί ε, στις ευθύνες της ως Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ υψηλέ οι προσδοκίες από την Αυστρία ακριβώς γιατί επίκυνται και ευρωεκλογέ το Μάιο του 2019. Γι' αυτό και θέλω να τονίσω ότι η συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών ε, οργάνων θα εξασφαλίσει ε, την επιτυχή ολοκλήρωση των εργασιών που έχουν ε, αναλυφθεί εδώ και πολλά χρόνια. Προτού υπησέλθω στους επιμέρους ε, τομείς πολιτικής, θα ήθελα να κάνω κάποιες βασικές παρατηρήσεις. Η Ευρώπη, και το είπε και ο κύριος Κίκλ, αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις και χρειάζεται βεβαίως μια ουσιώδηση μεταστροφή. Πρέπει να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η ικανότητα δράσης του ευρωπαϊκού εγχειρήματο. Είμαστε υπόλογοι απέναντι στους πολίτες μας προκειμένου να εξασφαλίσουμε ταχύς και αποτελεσματικές λύσεις και μπορώ να σα διαβεβαιώσω ότι η Αυστριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για την επιτεύξη τέτοιων λύσεων. Είμαι πεπισμένο ότι η Αυστριακή Προεδρία με την αναγνώριση και τη την προσήλωσή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα συμβάλλει ε, μαζί με όλες τις φιλοευρωπαϊκές δυνάμεις στην πρόοδο του κοινού μας εγχειρήματος. Ταυτόχρονα όμως πρέπει να τονίσω ότι... Ε, δεν πρέπει να είναι αυτό σκοπό η ανάληψη δράση στο επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντίθετα, ε, δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να αναλαμβάνεται μόνο εκεί όπου πράγματι και τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από ότι αν κάθε κράτο μέλο αναλάβει μόνο του δράση. Γι' αυτό και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται πλέον να στρέψει την προσοχή της και, του και τους σπόρους της σε πολύ συγκεκριμένου και λιγότερου από ό,τι μέχρι σήμερα τομεί. Εδώ σε αυτό συγκαταλέγεται βεβαίω η βελτίωση της αρχιτεκτονική ασφάλεια και τη δικαστική και αστυνομική συνεργασία, η ενίσχυση τη εσωτερική αγορά, αλλά και η ενίσχυση της σταθερότητα των γειτονικών μας κρατών. Επικορικότητα λοιπόν σημαίνει λιγότερα πράγματα, αλλά πιο αποτελεσματικά, χωρί ταυτόχρονα να σημαίνει μείωση της Ευρώπη. Αντίθετα, κάτι τέτοιο θα ενισχύσει την αποδοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωσης στου πολίτε μα και έτσι θα ενισχυθεί συνολικά και μακροπρόθεσμα και ε, το ευρωπαϊκό πνεύμα. Γι' αυτό το λόγο η, ευρωπαϊκή, η Αυστριακή Προεδρία έχει τρεις βασικές προτεραιότητες στη δικαιοσύνη και, στην εσωτερική, ε, και στις εσωτερικές υποθέσεις. Ενίσχυση της ασφάλειας. Σύνθημά μας είναι η μια Ευρώπη που θα προστατεύει. Είναι ακριβώ έτσι τα πράγματα. Η Ευρώπη πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να προστατεύσει του πολίτε τη και για τον σκοπό αυτό είναι αδύρυτη ανάγκη η βελτίωση τη συνεργασία προ όφελο των Ευρωπαίων πολιτών καθώ και η εναρμόνιση των νομικών μα προδιαγραφών. Αυτό αφορά ιδίω όσον αφορά την καταπολέμηση τη τρομοκρατία και του οργανωμένου εγκλήματο καθώ και η καταπολέμηση ε, του διασυνορικού εγκλήματο και η αντίστοιχη βελτίωση τη διασυνορική μα συνεργασία στι ποινικέ υποθέσει. Και γι' αυτό το σκοπό είναι πολύ σημαντικό σημαντικό, ιδίω οι ποινικοί φάκελοι που ε, τους οποίους επεξεργαζόμαστε να ολοκληρωθούν. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που επί Βουλγαρική Προεδρία καταφέραμε να καταλήξουμε σε πολιτική συμφωνία για την οδηγία για την καταπολέμηση τη ε, νομιμοποίηση παράνομων εσόδων καθώς και ε, την, τον, του οργανωμένου εγκλήματος και ακριβώς επειδή στο επίκεντρο της προσοχής μας είναι η ενίσχυση της ασφάλειας των πολιτών, είναι πολύ σημαντικό για εμάς να ε, καταφέρουμε να ε, καταλήξουμε ε, μαζί με εσά, με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε συγκεκριμένες λύσεις εμείς έχουμε κάνει τα απαραίτητα ε, βήματα συμβιβασμού. Σας καλώ να κάνετε και εσείς το ίδιο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρώ όμως ότι δεν είναι αγεφύρωτες οι διαφορές αυτές. Πρέπει ε, κοινό μας στόχος να είναι να δαθεί η δυνατότητα στις ε, αρχές επιβολής του νόμου να μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά να έχουν στη διάθεσή τους τις πληροφορίες προκειμένου να εκτελούν τα καθήκοντά τους και το έργο τους. Και σε αυτό το σκοπό ε, πρέπει να εξασφαλιστούν οι ε, απαραίτητες προϋποθέσεις για να μπορούν να κάνουν το έργο τους. Ο συμβασμός, λοιπόν πρέπει καλή την πίστη να εξευρεθεί προκειμένου να καταλήξουμε ενδεχομένως ακόμη και τον Οκτώβριο σε απόφαση στη Σύνοδο των Υπουργών Δικαιοσύνης. Και θέλουμε επίσης να προχωρήσουμε το έργο μας στις, ε, στον τομέα των μέσων πληρωμής. Στο Συμβούλιο ήδη έχουμε καταληξεί σε συμφωνία. Αυτή η νομική πράξη θα μας δώσει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε τις ε, ε, προκλήσεις καθώς και τεχνικά προβλήματα που έχουμε αντιμετωπίσει ε, όσον αφορά τα μέσα πληρωμών και στο βαθμό που αυτά συνδέονται με τη χρηματοδότηση τρομοκρατία και οργανωμένου εγκλήματο. Σε αυτά συγκαταλέγονται, για παράδειγμα, η καταπολέμηση απατών όσον αφορά την, την παραποίηση ε, στοιχείων πληρωτή και ε, μεταβιβάσεων χρηματικών ποσών μέσω τραπέζης. Γι' αυτό και θέλουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο στον τριμερή διάλογο. Όσον αφορά τα τεχνολογικά ε, εργαλεία που χρειαζόμαστε για την καταπολέμηση αυτού του είδους του εγκλήματος χρειάζεται να προχωρήσει το έργο όσον αφορά την οδηγία για τις ηλεκτρονικές ενδείξεις. 13 Ιουλίου στο Ίνσμπουργκ θα γίνει μια πρώτη άτυπη υπουργική διάσκεψη όπου θα συζητηθεί το θέμα αυτό και συγκεκριμένα των ε, αντικρώμενων συμφορώντων μεταξύ παρόχων υπηρεσιών πληρωμών. Εδώ ε, ε, μιλούμε για το ζήτημα της ε, της, ε, του, του, του, ότι κάποιο πάροχος ε, υπηρεσία πληρωμών μπορεί να έχει την έδρα του εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να παρέχει τι υπηρεσίε του στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το καθεστώς ε, που διέπει τι ενέργειες των αρχών επιβολή του νόμου και πώ μπορούν να αντιμετωπίζουν τέτοιες, τέτοια θέματα όταν ανακύπτουν ή υπάρχουν ενδείξει ή υποψίε για εγκληματικέ δραστηριότητε. Το Σεπτέμβριο θα ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Δεύτερη προτεραιότητα και κύριο στόχο τη Αυστριακή Προεδρία είναι η ενίσχυση της ψηφιοποίησης, ε, της διαδικασίας ψηφιοποίησης της Ευρωπαϊκής Ενιαίας Αγοράς. Θεωρώ ότι αυτό είναι μια προτεραιότητα ε, σε, ευρωπαϊκό επίπεδο που θα εξασφαλίσει και την καλύτερη πρόσβαση καταναλωτών σε υπηρεσίες και προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό θέλουμε να το καταλήξουμε, ε, να το καταφέρουμε μέσω αναθεώρησης και αναβάθμισης του νομοθετικού πλαισίου για τα πνευματικά δικαιώματα. Τέλος, ε, όπως είπε και ο Υπουργός Κίκλ, θέλουμε να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία μας με τις χώρες της γειτονία μας, ιδίως με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Και εδώ και σε αυτό το τομέα η Αυστριακή Προεδρία ε, διοργανώνει ε, υπουργή διάσκεψη στην Αλβανία. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ανεξαρτησία των ε, συστημάτων δικαιοσύνης σε, ε, ολόκληρο, σε ολόκληρα τα Δυτικά Βαλκάνια. Να ε, τονίσω κάτι τελευταίο. Η θεσμική συνεργασία μπορεί να βελτιωθεί μόνο αν υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη όσον αφορά τα πρότυπα κράτους δικαίου που διέπουν τη δικαιοσύνη μας. Και γι' αυτό χρειάζονται συγκεκριμένες συνθήκες πλαίσιο. Τα εργαλεία μας μπορούν να αποφέρουν τους επιθυμητούς καρπούς μόνο αν ε, ε, ακολουθούν αυστηρούς κανόνες κράτους δικαίου, κάτι που προϋποθέτει και επαρκείς χρηματοδοτικούς πόρους. Το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο, όμως αποτελεσματικό θα είναι αυτό το εργαλείο μόνο όταν κάθε κράτος μέλος θα έχει ένομη τάξη η οποία θα αντιστοιχεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα. Και από αυτό προκύπτει βεβαίως ότι υπάρχει πάρα πολύ έργο που πρέπει να κάνουν όλες οι πλευρές και αυτά τα θέματα θα συζητηθούν και στην υπουργική διάσκεψη που θα γίνει στο Ίνσπρουκ 13 και 14 Ιουλίου. Τα, ε, οι εκκρεμείς φάκελοι περιλαμβάνουν και θέματα όπου πραγματικά δεν γίνεται να βρούμε απλά έναν κοινό ελάχιστο παρονομαστή, αλλά λύσεις για το μέλλον. Και σε αυτό το πλαίσιο θα ήθελα να ευχαριστήσω το, το τρίο των Προεδριών, Βουλγαρία, Εστονία για το έργο τους και θέλω να καλέσω και εσάς αγαπητά μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να σας πω ότι όπως εσείς έχετε ε, προσδοκίε από εμά, έχουμε και εμεί προσδοκίε από εσά. Ιδίω στον τομέα τη οδηγία για τι ηλεκτρονικέ ενδείξει, ε, είμαστε ε, έτοιμοι να καταλήξουμε σε συμβιβασμό, σε συμφωνία γιατί κάθε άλλη λύση τελικά θα αποβεί ει βάρο των πολιτών. Γι' αυτό και θα σας καλό να καθίσετε μαζί μας στο τραπέζι των συζητήσεων των διαπραγματεύσεων ακριβώς για να προωθήσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, τις ευρωπαϊκές λύσεις που χρειάζονται οι πολίτες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τους δύο υπουργούς για τις παρουσιάσεις. Έχουμε έναν μακροσκελέστατο κατάλογο ομιλητών από τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Όπως είπα και προηγουμένως, θα ξεκινήσουμε από τους συντονιστές των πολιτικών ομάδων ή μέλη ε, του Κοινοβουλίου που εκπροσωπούν ε, τους συντονιστές. Πρώτος έχει το λόγο ο κύριο Μπέκερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τους δύο υπουργού για τις παρουσιάσεις τους, την παρουσίαση του προγράμματος της Προεδρία. Μπορώ να σας θέσω στον καθένα από δύο ερωτήσεις. Πρώτον, όσον αφορά αυτή την μεταστροφή την ε, οποία ανέφερε ο κύριος Κίκλ, θέλω να πω ότι την υποστηρίζω πλήρως. Άλλωστε φαίνεται και σε παρευρωπαϊκό επίπεδο ότι αυτή η μεταστροφή προσκρούει στην, ε, σε δίκο αότα στους Ευρωπαίους πολίτες. Και θέλω να πω ότι αυτή η απώλεια εμπιστοσύνης στους πολιτικούς τα τελευταία χρόνια δεν αφορά μόνο την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεσμικά όργανα της, αλλά και ε, την κάθε κυβέρνηση ξεχωριστά. Αυτό άλλωστε φάνηκε και από τις διαφωνίες που εμφανίστηκαν τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Γι' αυτό και αυτή η μεταστροφή πραγματικά αποτελεί μια νέα τάση που πραγματικά είναι πολύ ευπρόσδεκτη. Όσον αφορά τις ε, βασικές παρατηρήσεις που ακούστηκαν σε σχέση με τα κέντρα διαχείρισης μεταναστών και προσφύγων και το ε, ερώτημα πού θα πρέπει να υποβάλλονται οι αιτήσει ασύλου, ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Το ερώτημα είναι προφανές. Πώς θα καταφέρετε να καταλήξετε συμφωνία μεταξύ των κρατών μελών σε αυτά τα ακαθόδη ζητήματα. Δεύτερο ερώτημα. Συζητούμε εδώ στο Κοινοβούλιο την θέσπιση ανθρωπιστικής θεώρησης. Κάτι που θα προστατεύσει όπως αναφέρεται ε, από τους ε, υποστηρικτές αυτής της θεώρησης, τους ανθρώπους από τους διακινητές. Εσείς ποια, ποια στάση έχετε απέναντι σε αυτή την πρόταση. Ερώτημα προς τον κύριο Μόζελ. Καταρχάς να σας ευχαριστήσω που εκφράσατε την προσήλωσή σας στην αρχή της επικουρικότητας. Είναι κάτι που το χρειάζεται πραγματικά η Ευρώπη. Και στο πλαίσιο αυτό θα ήθελα να σας θέσω το εξή ερώτημα. Ποια είναι η πρόσβασή σας ε, ποια είναι η προσέγγιση σας όσον αφορά τους ε, τομείς ε, που αφορούν την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα. Εκεί όπου ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ήδη έχει τεθεί σε ισχύ και όπου πραγματικά έχουν εκφραστεί σημαντικότατη φόβη ότι μπορεί και να δημιουργηθεί ένα υπερβολική διοικητική επιβάρυνση για όλους τους εμπλεκόμενους. Τέλος, Υπάρχει επικείμενη ψηφοφορία για την ε, οδηγία για την καπιτολέμηση της, ε, ε, της νομιμοποίησης παράνομων μεσόδων. Θεωρείτε ότι είναι επαρκές αυτό το εργαλείο. Κύριε Βάιντεν Χόλσερ εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ αγαπητοί Υπουργοί Νομίζω ότι το θέμα της ε, σημερινής μας συζήτησης δεν είναι η αξιολόγηση της εσωτερικής πολιτικής στην Αυστρία, αλλά πώς η Αυστρία θα καταφέρει να συμβάλλει στην νομοθετική διαδικασία σε ε, επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποια προσέγγιση θα ακολουθήσει, πώς θα συμβάλλει σε αυτή τη διαδικασία η Αυστρία, διότι υπάρχει πάντοτε και ένα πριν και ένα μετά. Έτσι βρισκόμαστε σε ένα συνεχές. Γι' αυτό και θέλω να θέσω συγκεκριμένα θέματα προς τους υπουργού. Γιατί βεβαίως στο τέλος ε, ξυρίζει κανείς τον γαμπρό, ε, στο τέλος θα γίνει ο υπολογισμό της Αυστριακής Προεδρίας. Γι' αυτό και ως προς το πρόγραμμά σας. Κύριε Κίκλη, ποια είναι η στάση σας απέναντι στον χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων και τη Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεδομένου ότι και τα δικαστήρια προσανατολίζονται και βασίζονται σε αυτά τα δύο έγγραφα. Τι πιστεύετε ιδίω για τη διάσωση, διάσωση προσφύγων στη θάλασσα. Δεύτερον, μιλήσατε για ένα πακέτο προτάσεων για το άσυλο και τη μετανάστευση. Όπως είπατε ακριβώς, είναι πακέτο, θα πρέπει κανείς να τα δει όλα μαζί αυτά τα θέματα. Πώς θα εξασφαλίσετε εσεί την ε, απρόσκοπτη ε, και ομαλή εξέλιξη των συζητήσεων. Εδώ και μήνες έχουμε καταλήξει σε ένα πακέτο και το Συμβούλιο αποφεύγει να πάρει απόφαση. Σαν καυτή πατάτα το παίρνει η μία Προεδρία και το παραδίδει στην επόμενη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μα η Αυστρία επιτέλου να αναλάβει τι ευθύνε τη ω Προεδρία και να καταλήξουμε σε, αυτόν τον, ε, σε αυτό το θέμα. Επίσης, είμαι εισηγητής για, τον, για την πρόταση κανονισμού για το πρόγραμμα δικαιοσύνης που θα τρέξει την επόμενη δεκαετία. Θέλω λοιπόν να ε, σας ρωτήσω, ποιες δυνατότητες βλέπετε για την ενίσχυση της διασυνορικής συνεργασίας και θέλω να συμπεριστώ αυτό που είπε ο κύριος Μπέκερ. Για όλους μας είναι πάρα πολύ σημαντικό να ολοκληρωθούν οι συζητήσεις για την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα και να καταβάλει προσπάθειες μεγάλες η Αυστριακή Προεδρία γιατί είδαμε και ότι ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων έφερε πολύ σημαντικά αποτελέσματα όχι μόνο στην Ευρώπη, σε ολόκληρο τον κόσμο και θα θέλαμε κάτι αντίστοιχο να γίνει και με την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα. Η κυρία Γκρίσμπεκ για τους φιλελεύθερου. Ευχαριστώ τους δύο υπουργού. Πολλές φορές στις παρεμβάσεις σας αναφέρεται ότι η Αυστρία θέτει την Προεδρία της και βασικό μέλημα μάλλον της Προεδρίας της θέτει την Ευρώπη που προστατεύει. Αυτό το σλόγγαν έχει να κάνει και με την προστασία των αξιών. Με την συνάδελφο Αγγέλικα που θα πάρει το λόγο στη συνέχεια, θα ήθελα μόνο ε, να κάνω μια μικρή μνήα σε ένα ψήφισμα που υιοθέτησε το Κοινοβούλιο για τα δικαιώματα των παιδιών και πιο συγκεκριμένα σε διαδικασία μετανάστευση ή Ε, που υιοθετήθηκε από το, την ε, διακομματική ομάδα για τα δικαιώματα του παιδιού. Θα ήθελα σε αυτό το εξάμεινο, εφόσον έχετε και το σλόγγαν ε, «Την Ευρώπη που προστατεύει», να υπενθυμίσω ότι η υποδοχή των ε, παιδιών θα πρέπει να γίνεται ε, σε κοινοτικά κέντρα και όχι υποκράτηση. Θα πρέπει πάντα κατά προτεραιότητα να εξετάζονται τα παιδιά και να τα χειριζόμαστε ως ευάλωτα άτομα. Ε, και να λαμβάνουμε πάνω απ' όλα υπόψη το συμφέρον του παιδιού, ε, να έχουμε με, εντός πέντε ημερών την, τον διορισμό ενός ε, ε κηδεμόνα και να υπάρχουν οι απαραίτητες συνθήκες για την υποδοχή αυτών των ανηλίκων. Παράλληλα πρέπει να υπάρχει και ψυχολογική υποστήριξη των λύκων που ενδεχομένω να έχουν πέσει θύματα βία και να έχουν πρόσβαση σε παιδεία και περίθαλψη. Μια αντίστοιχη λοιπόν προστασία, αντίστοιχο επίπεδο με την ευρωπαϊκή προστασία. Επομένω, αυτό το τα επίπεδα προστασία πρέπει να είναι ίδια, είτε πρόκειται για ένα παιδί που προέρχεται από τη μετανάστευση, είτε για ένα ε, παιδί της Ευρώπης. Ελπίζω και η Αυστριακή Προεδρία να εργαστεί από κοινού μαζί μας για να πετύχουμε ακριβώς αυτή την Ευρώπη που προστατεύει. Thank you very much. Mr. Argentini, please. Η κυρία Σαρτζεντίνη. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα, κράτος δικαίου. Πρόσφατα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων έκαναμε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την Πολωνία κατόπιν ε, πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκκίνηση διαδικασίας ε, παραβάση υπό το άρθρο 7. Δεν ξέρω πότε θα λάβει η χώρα η επόμενη συζήτηση και τι έχετε βάλει εσείς ως στόχο για αυτήν την διαδικασία. Ξεκίνησε λοιπόν η διαδικασία το Δεκέμβριο του 2017 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επομένως, ε, έχει έρθει η ώρα να περάσουμε και στην πράξη. Φαντάζομαι ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τις ερευνές του μέχρι τώρα. Δεύτερον, μετανάστευση και άσυλο. Η Σύνοδος Κορυφής πριν από δύο εβδομάδες μίλησε για την ανάγκη ε, συνένεσης για το Δουβλίνο, ότι πρέπει να εξευρεθεί συνένεση μεταξύ των κρατών μελών για το Δουβλίνο. Ε, μπορείτε να μας εξηγήσετε ποιος θα είναι ο ρόλος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γιατί εάν η συνένεση πρέπει να εξευρεθεί μεταξύ των κρατών μελών, το πιο πιθανό είναι να παραγωνιστεί το ε, Κοινοβούλιο, ενώ εμείς είμαστε εδώ και χρόνια έτοιμοι να διαπραγματευτούμε μαζί σας. Επίσης, συμφωνήσαμε ε, επιορισμένων τεμερών διαλόγων με την Βουλγαρική Προεδρία και μια εβδομάδα αργότερα μάθαμε ότι δεν θα τα υιοθετήσει η Κορεπέρ για την ε, ε, για συγκεκριμένες διαδικασίες μετανάστευσης όπως είναι η επαναγκατάσταση. Θα υπάρξει επαναδιαπραγμάτευση με την Βουλγαρική Προεδρία γι' αυτό. Τώρα, εξέτασα ε, τα στοιχεία. 44 άτομα έχει μετακαταστήσει η ε, Ιταλία και κανέναν από την Ελλάδα. Ε, θα ακολουθήσετε τα στοιχεία για την ενδονοσιακή μετακατάσταση όπως έχουν τεθεί μέχρι τώρα. Πρέπει να μας δώσετε ένα παράδειγμα που να δείχνει ότι η αλληλεγγύη είναι ο μοναδικός δρόμος για μια ευρωπαϊκή λύση της κρίσης ασύλου και μετανάστευσης ή για να το πω καλύτερα της πολιτικής κρίσης με πολύ ε, χαμηλά στοιχεία. Τέλος, ε, αυτές, αυτά τα περιφερειακά κέντρα ε, τα disembarkation centers. πολλοί λένε ότι δεν θα έχουν τέτοιου είδους κέντρα. Ποια είναι τα σχέδια της ε, ε, Προεδρίας σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Ένστ, παρακαλώ. vielen herzlichen Dank. Ευχαριστώ πολύ. Για τον κύριο Κίκλ, θέλω να θέσω τις εξής ερωτήσεις. Εξήρατε τις αποφάσεις του τελευταίου συμβουλίου στον τομέα του ασύλου. Εκεί προτείνεται ότι τρίτες χώρες θα ενθαρρύνονται από εδώ και στο εξή και θα υποστηρίζονται ώστε να ε, εγκαταστήσουν καταβλισμούς για ετούντες άσυλο στην Αφρικανική Ήπειρο. Δεν υπάρχουν όμως καθόλου θετικά στοιχεία ή πληροφορίες από τις χώρες αυτές Πώς ακριβώς σκοπεύετε να ενθαρρύνετε, όπως λέτε, ε, τις χώρες ε, της Βόρειας Αφρικής να δημιουργήσουν καταβλισμούς. Επίσης, ε, στο Συμβούλιο αποφασίστηκε ότι προαιρετικά κράτη-μέλη θα μπορούν να υποδέχονται ετούντες άσυλο. Εσείς ποιος πιστεύετε ότι θα υλοποιήσει αυτό την, την προαιρετική δυνατότητα. Θεωρείτε ότι στην πράξη ρεαλιστικά θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο, θα υπάρξει κράτος μέλο το, οποίο θα υποδεχθεί εθελοντικά ετούντε άσυλο. Τρίτον, υπάρχουν ε, οι γνωστέ προτάσει του Horst Seehofer τα τελευταία χρόνια ε, να δημιουργηθούν ε, κέντρα διαχείρισης η κυβέρνηση συνασπισμού στη Γερμανία εξέφρασε προς το παρόν την ανοχή της σε μια τέτοια θέση. Εσάς ποια είναι η στάση σας. Η κυβέρνησή σας ε, έχει δηλώσει ότι δεν υπάρχει περίπτωση ε, οι λύσεις που θα βρεθούν σε ε, ευρωπαϊκό, επίπεδο να αποβούν σε, σε, σε βάρος της Αυστρίας. Ποια είναι η θέση σας λοιπόν και απέναντι σε στάσεις όπως εκείνη της Ιταλίας, όπως της κυβέρνησης της Ιταλίας. Επίσης, ο τριμερής διάλογος κατέληξε συγκεκριμένα αποτελέσματα σε ζητήματα της μετανάστευσης επί βουλγαρική προεδρία, τα οποία όμως φαίνεται ότι τώρα έχουν παγώσει, αφού αναλάβατε εσείς τα καθήκοντα της προεδρίας. Τέλος, ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε υποβάλει μια πρόταση για το Δουβλίνο 4 εσείς μπορείτε να δεσμευτείτε ως Αυστριακή Προεδρία ότι θα δώσετε την απαραίτητη προσοχή σε αυτή την πρόταση του Κοινοβουλίου ή δεν θα ασχοληθείτε καθόλου όπως αφορά την ε, επανένωση οικογενειών, την κοινωνική ένταξη των ετούντων άσυλων, των προσφύγων, τα κοινωνικά δικαιώματα των ε, προσφύγων καθώς και την κατάργηση ε, ε, αυτής της ε, ρήτρα ότι η πρώτη χώρα εισόδου θα πρέπει να είναι εκείνη που θα διαχειρίζεται τις αιτήσει ασύλου. Ποια είναι η στάση σας απέναντι στην πρόταση που έχει υποβάλει το Κοινοβούλιο για την αναθεώρηση του Δουβλίνου 4. Κύριε Μπόνη. Ευχαριστώ πολύ για τις παρουσιάσεις. Είναι θετικό που συνδυάζεται ορισμένα θέματα, τα οποία είναι σημαντικά για λόγους ασφαλείας, είναι σημαντικά για τους πολίτες και για το κράτος δικαίου. Δύο ερωτήματα. Πρώτον, πώς ε, σκοπεύετε ε, να κινηθείτε για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου σε ορισμένες χώρες. Ξέρουμε. Εγώ είμαι Πολωνός. Εξάλλου, ξέρουμε ότι η Πολωνία ε, περνάει τη διαδικασία του άρθρου 7 αλλά το σχόλιο μου δεν αφορά μόνο αυτές τις διαδικασίες, αλλά για το πώς θα γίνει πιο ευνόητο το κράτος δικαίου και πώς θα ασκήσουμε πιέσεις στις κυβερνήσεις. Γιατί έχουμε αφενός μετανάστες ε, προς την Ευρώπη, αλλά θέλουμε να τηρείται και το κράτος δικαίου. Και δεύτερον, η ιδιωτικότητα που αναφέρθηκε προηγουμένως είναι Πολύ σημαντικό αυτό το ζήτημα. Γιατί στην, κατά την Βουλγαρική Προεδρία δεν υπήρξε κανένα τριμερή διάλογο. Επομένω, σε αυτή την Προεδρία είναι η τελευταία ευκαιρία να τα συζητήσουμε. Χαιρετίζω και τη δήλωσή σας ότι πρέπει να προστατεύσουμε ε, και την ιδιωτικότητα, αλλά και να ε, δημιουργήσουμε το κατάλληλο περιβάλλον καινοτομία. Αυτά, ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζέλστρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τους υπουργούς ε, για τις παρεμβάσεις τους. Η νέα αυστριακή κυβέρνηση ήδη έχει πετύχει ε, στο στόχο της ε, ως προς την επιβολή απλών αλλά αποτελεσματικών εναλλακτικών. Και αυτό καταδεικνύει την έλλειψη εναλλακτικών ε, που προσφέρει η γερμανική κυβέρνηση. Σε αντίθεση λοιπόν με τη γερμανική κυβέρνηση, η αυστρική κυβέρνηση υιοθετεί νέα μέτρα που είναι απαραίτητα για το καλό της Ευρώπης. Και αυτό δείχνει ότι ο καγκελάριος ε, ήταν σε θέση να ε, εφαρμόσει μια σειρά μέτρα μεγάλη επιτυχία. Έχετε επιφέρει αλλαγές στην νομοθεσία σας πρόσφατα, για παράδειγμα πρόσβαση σε δεδομένα ή η δυνατότητα ε, δίμευσης ρευστού ή απώλεια της άδειας παραμονής. Μία σειρά μέτρα λοιπόν που έχετε υιοθετήσει πρόσφατα θα συνεχίσετε να προωθείτε αυτή την ε, πολιτική. Όσον αφορά την ε, δημιουργία καταβλησμών στην Αφρικανική Ήπειρο, κάτι που εκφράστηκε ως αίτημα ήδη από το 2014 από τον κύριο Φιλίμσκι, θεωρείτε κατά τη γνώμη σας λοιπόν κάτι τέτοιο θα επιφέρει θετικές αλλαγές όσον αφορά την ε, τροποποίηση του ε, Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Θα ενισχυθεί η αρχή, ότι, ε, η αρχή της, της προαιρετικότητας. Ο κύριος Μιούλε. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας εδώ. Κύριε Κίκλ, ξεκινήσατε λέγοντας ότι υπάρχει μια μεταναστευτική κρίση στην Ευρώπη. Εγώ όμως έχω την εντύπωση ότι δεν έχουμε μια κανονική μεταναστευτική κρίση, διότι οι αριθμοί των ε, μεταναστών μειώνονται διαρκώς. Έχουμε όμως πολιτική κρίση. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, στην Ευρώπη εμφανίζονται και ανακύπτουν διαρκώς νέα κόμματα τα οποία καταχρώνται αυτό, την ατζέντα της μετανάστευσης για ε, ίδιο πολιτικό όφελος. Ε, αναφερθήκατε και σε μια μεταστροφή. Θα το πω ξεκάθαρα. Αν αυτή η μεταστροφή αφορά τη δημιουργία καταβλισμών στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο ή τη δημιουργία ε, κέντρων διαχείρισης και διαμετακόμισης, τότε την δική μας ε, υποστήριξη ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θα την έχετε. Ε, δεν είναι αυτό που χρειαζόμαστε. πρέπει επιτέλους να δοθεί ένα τέλος σε σε αυτήν την αποστροφή που ε, εμφανίζεται απέναντι στους πρόσφυγες και πραγματικά μου έκανε αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ούτε μία λέξη δεν βρήκατε να πείτε για την προστασία των προσφύγων και την ευρωπαϊκή πολιτική που θα πρέπει να ακολουθεί στον τομέα αυτό. Εδώ και χρόνια έχετε ψηφίσματα και προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ως Συμβούλιο και δεν κάνετε τίποτα. Και αναρωτιέμαι πραγματικά πώς πώς θέλετε να καταλήξουμε σε συμφωνία όταν διαρκώς το μόνο για το οποίο ακούμε από εσάς είναι το κλείσιμο ε, συνόρων όταν δεν έχετε να πείτε ούτε μία κουβέντα για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και όταν το μόνο που ξέρετε να προτείνετε είναι η δημιουργία και η θέσπιση κέντρων ε, κράτησης για τους πρόσφυγες. Αυτή είναι η τομή στους οποίους θα κρυθεί το έργο σας. Εκεί είναι, ε, αυτή είναι η τομή στους οποίους πραγματικά χρειάζεται να, βρείτε και να βρούμε από κοινού λύσεις. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, μου δίνετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και τους ε, δύο υπουργού για τις παρεμβάσεις τους. Δεν θα θίξω ζητήματα που ήδη ανέφεραν άλλοι. Θα ήθελα να σταθώ μόνο σε ένα ζήτημα το οποίο ακόμα δεν έχει αναφερθεί. Και αυτό είναι το θέμα της διαδικασίας ασύλου εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος στις διαπραγματεύσεις σας ε, με χώρες όπως η Αλβανία ή χώρες της ε, Βορείου Αφρικής. Θεωρείτε ότι υπάρχει βούληση και προθυμία από πλευρά τους ε, να δημιουργηθούν ενδεχομένως προσωρινοί καταβλισμοί όπου θα λαμβάνουν χώρα αυτές οι διαδικασίες. Και δεύτερον, αυτές οι διαδικασίες δεν θα αυξήσουν την ε, έλξη που ασκεί η Ευρωπαϊκή Ένωση προς αυτούς τους ανθρώπους, που είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε να περιορίσουμε. Τρίτον, νομικός αντίκτυπος αυτών των ε, διαδικασιών. Έστω ότι υπάρχει μια τέτοια θετική απόφαση. Όλα τα κράτη-μέλη θα πρέπει να τις δεχθούν. Τι θα γίνει. Μάλιστα, θα διαβάσω τον ε, κατάλογο μελετών για να έχετε μια εικόνα. Miss Spinelli, Miss Mlinar, Mr. Koester, Miss Gomez, Miss Björk, Mr. Pavel, Miss Yaroka. Am I missing someone? Yes, and Wimberg. Ξέχασα κανένα, μάλιστα, και κυρία Βίμπερκ. Άλλος κανείς? Ναι, να προσθέσω και το δικό μου όνομα στο τέλος. Ο κύριος Λόπες Αγγιλάρη. Είναι θέμα τυπικό αλλά και καλή θέληση η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ να εκφράζει τι ευχέ τη. για κάθε επιτυχία στην καινούργια Προεδρία, την περιοδική εξαμηνία Προεδρία τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ίδιο θα κάνουμε και προ την Αυστριακή Προεδρία. Επίση από την άλλη, η Αυστριακή Προεδρία λαμβάνει χώρα σε μια αποτελεσματική συγκυρία, συγκυρία σε μια αποφασιστική συγγνώμη συγκυρία. <laughs> Πρέπει να σας πω ότι θα είναι η μόνη εναπομείνας πλήρης προεδρία πριν τις επερχόμενες ευρωεκλογές το 19. Και Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνουμε στον τομέα αρμοδιοτήτων της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ είναι πολύ πενιχρά και αυτό είναι πολύ ανησυχητικό και θα πρέπει να κάνετε κάνει για να βελτιώσετε τις επιδόσεις. Γιατί υπάρχουν διάφοροι φάκελοι που έχουν μπλοκαριστεί εδώ και καιρό στο Συμβούλιο δεν έχει την θέληση το Συμβούλιο να καταλάβει ότι μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης. Ε, είναι ισότιμο όργανο με το Συμβούλιο. Δεν παίζει μόνο αυτό το ρόλο του, του νομοθέτη το Συμβούλιο. Δεν, δεν παίζει μόνο του, δεν παίζει ενού παικτής. Είμαστε κι εμείς εδώ, το Κοινοβούλιο. Και ακούσαμε όλα όσα είπατε πολύ προσεκτικά. Να σας τονίσω ότι υπογραμμίζεται η έννοια της ασφάλειας. Ε, το Συμβούλιο μιλάει για διαλειτουργικότητα, ποιος μπαίνει μέσα από τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τονίζει συνέχεια την ασφάλεια. Αλλά και εμείς κάναμε μια εναλλακτική ανάλυση και εναλλακτική προσέγγιση που την ονομάζουμε ολιστική προσέγγιση και μιλάμε επίσης για αλληλεγγύη Μιλάμε επίσης για μικτές αρμοδιότητες. Μιλάμε επίσης για σεβασμό στην αξιοπρέπεια και στα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των ατόμων που ακολουθούν το μονοπάτι της μετανάστευσης και κυρίως των ετούν τον άσυλο, δίνουμε σημασία στους νομοθετικούς φακέλους που εκρεμούν και δεν έχουν αποφασιστεί στο Συμβούλιο. Σας επιστούμε, επιστούμε την προσοχή ότι πρέπει εσείς να κάνετε τη διαφορά και να προωθήσετε αυτούς τους φακέλους, αυτά τα θέματα που εκκρεμούν. Υπάρχει ένα θέμα, κωδικός θεωρήσεων. Ε, είμαι εισηγητής σε αυτό το θέμα. Ε, εδώ και δύο χρόνια έχει μπλοκαριστεί. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να, κάνετε ό,τι μπο... για... να συμφωνήσουμε το Συμβούλιο. Κάντε και εσείς ό,τι μπορείτε, ούτως ώστε αυτός ο φάκελος, επί του οποίου είμαι εισηγητής, να ολοκληρωθεί πριν από το τέλος αυτής της κοινοβουλευτικής θητείας. Και μία ερώτηση προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης, ο οποίος είπε το εξής. Μίλησα για τη σημασία της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και αναγνώρισης στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Δικαστικής Συνεργασίας. Αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαία αναγνώριση. Αυτές ε, μειώνονται, για να μην πω ότι καταραίουν τα τελευταία χρόνια. Το Ευρωπαϊκό Εντάγμα Σύλληψης, χάλια τα πάει. Δεν παίζει το ρόλο του θα πρέπει όχι μόνο να λέτε κουβέντε για αυτά, αλλά να δεσμευτείτε για να αποκαταστήσετε την αμοιβαία εμπιστοσύνη και αμοιβαία αναγνώριση των αποφάσεων στα πλαίσια τη ε, δικαστική συνεργασία. Επίσης, το άρθρο 7 και η συνθήκη της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έχουμε μια εκκρεμότητα εδώ για την Πολωνία και Ουγγαρία. Σας παρακαλώ. Συμφωνήσαμε για το χρόνο, συνάδελφοι. Προσοχή, σας το υπενθυμίζω, έτσι. Μην έχουμε υπερβάσεις. Η κυρία Σπινέλη είναι επόμενη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν με πείθει ο Υπουργός Κύκλου. Δεν με πείθει ότι έχει αλλάξει νοτροπία. Και αυτό που προτείνει δεν με πείθει και δεν νομίζω ότι πείθεται το Κοινοβούλιο. Είναι μια αλλαγή νοοτροπίας που βασίζεται στο ότι εγκαταλείπουμε την έννοια της αναδιανομής των ε, υποχρεώσεων, ε, εστιαζόμαστε απόλυτα στον έλεγχο των ε, συνόρων και εγκαταλείπουμε παντελώς την αρχή της αλληλεγγύης. Και η αλληλεγγύη αφορά μόνο τον έλεγχο των συνόρων. Λοιπόν, θα ήθελα να πω τρία πράγματα για αυτή την αλλαγή υποτιθέτης νοοτροπία. Σημεία που δεν, δεν είναι απλώ προβληματικά, αλλά δεν μπορούν να εφαρμοστούν. Καταρχά, οι πλατφόρμες αυτές, οι χώροι αυτοί αποβίβασης στις τρίτες χώρες. Ποιοι είναι οι εταίροι μα στην Αφρική, όταν οι περισσότερε βορειοαφρικανικέ χώρε έχουν πει όχι σε, αυτά, σε αυτού του χώρου. Δεν υπάρχει καμία δέσμευση για μετεγκατάσταση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είπα η αρμοστία για τους πρόσφυγες μας είπαν ότι δεν θα ασχοληθούν με, αυτούς, με αυτά τα κέντρα εάν δεν εγγυώνται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Τα κέντρα διέλευσης, δεύτερο σημείο. Θα, έλεγα, θα τα έλεγα καλύτερα κέντρα κράτησης, έτσι, όχι διέλευσης. Είναι εξεδαφικά κέντρα και θα ήθελα αυτούς που τους, στερούν, που τους η ελευθερία ε, γιατί τους κατηγορούμε, έτσι. Είναι χειρότερο από τον Κουαντάναμο. Επίσης, η απόρριψη της μεταρρύθμισης της, ε, του Δουβλίνου. Μια μεταρρύθμιση που την ήθελε το Κοινοβούλιο και που βασιζόταν στην αναδιανομή και στην αλληλεγγύη. Πώς θέλει να αλλάξει την οτροπία όταν τίποτα δεν γίνεται από αυτού. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να προασπίσετε τη μεταρρύθμιση που πρότεινε το Κοινοβούλιο, τα δύο τρίτα τουλάχιστον των Ευρωβουλευτών την υπερψήφισε αυτή την ε, πρόταση. Και πώς θα επιτύχετε την ε, συνένεση, γιατί συνένεση σημαίνει ομοφωνία και ομοφωνία σημαίνει εγκατάλειψη της πρότασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλετε να την εγκαταλείψετε. Αυτά ευχαριστώ. Thank you. Ευχαριστώ. Äh, Κυρία Μολίνα, ευχαριστώ για την παρουσία σας και τις παρουσιάσεις σας, κύριε Υπουργή. Είπατε και οι δύο δικαίως ότι επιδιώκετε και ελπίζετε τη συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι είναι σαφές σε όλους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε αυτό το θεμέλιο της προθυμίας για συνεργασία. Πρόκειται για θεμέλιο λίθο του εγχειρήματό μας. Γι' αυτό και ε, εγώ μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας αν βεβαίως γίνονται σεβαστές οι ευρωπαϊκές αξίες, ανθρώπινα δικαιώματα, θεμελιώδη δικαιώματα. Και νομίζω ότι σε αυτό το τομέα δεν αναφερθήκατε επαρκώς. Η Ευρώπη λοιπόν βασίζεται για εμένα ως φιλελεύθερη πολιτικό ακριβώς σε αυτές τις αξίες της συνεργασίας και της συνύπαρξης. Και όπως είπαν και οι συνάδελφοί μου, για μας είναι αποφασιστική σημασίας πώς θα χειριστείτε αυτά τα τρία, τις τρεις πράξεις ε, που αφορούν τη μετανάστευση και το άσυλο. Έχει γίνει πάρα πολύ δουλειά τα τελευταία χρόνια Φτάσαμε από μέσα από δύσκολε διαπραγματεύσει σε ένα αποτέλεσμα και βλέπουμε τώρα η διαδικασία να μπλοκάρει στο Συμβούλιο. Γι' αυτό και το ερώτημα προ εσά, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα ερώτημα και ένα θέμα που απασχολεί του Ευρωπαίου πολίτε και μόνο ευρωπαϊκή μπορεί να είναι η λύση. Τι θα κάνετε, κύριε Μόζη. Είπατε σωστά για το ζήτημα της ιδιωτικής ιδιωτικότητας και ε, ε, των ηλεκτρονικών ενδείξεων. Το μόνο πρόβλημα που ε, βλέπω εγώ είναι ότι, πρέπει να αποφευθεί ε, κάθε πιθανότητα ε, διακρίσεων εις βάρος ε, υπηκών ε, πολιτών διπλή, με διπλή υπηκότητα. Ποια είναι η στάση σας, κύριε Κιώστολ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σαφής. Ανησυχώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα καταφέρει να αποφύγει σοβαρά πλήγματα στην αλληλεγγύη και τη δημοκρατία το επόμενο εξάμεινο. Όποιο θεωρεί ότι μπορεί να παίζει με έννοιε όπως η επικουρικότητα, να τι αναιρέσει και να τι υπονομεύσει, ακόμα και έννοιε που είναι κατοχυρωμένε στη συνθήκη τη Λισαβόνα και στη Χάρτα των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων. Όποιο παίζει με την ιδέα ότι μπορούν άνθρωποι να επελάβνονται σε αφρικανικές χώρες όπου αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο βιασμών, βασανιστήριων αντίκειται στις βασικές αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, μου φαίνεται περίεργο πώς είναι δυνατόν να μιλάτε για μεταναστευτική κρίση. Έχουμε μια κρίση των πολιτικών απέναντι στους πρόσφυγες και στους μετανάστες. Αυτός είναι ο σωστός όρος. Και μιλώντας για τους μετανάστες και, τους, ε, και το άσυλο και, τη, και συνδέοντας αυτό το θέμα με την ασφάλεια και την τρομοκρατία, δημιουργείται την εντύπωση την ασφαλμένη ότι άνθρωποι που από ανάγκη κατέφυγαν και καταφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρομοκράτες και εγκληματίες. Θέτεται λοιπόν ανθρώπους εκτός της κοινότητάς μας τους εντάσσεται σε μια ιδιαίτερη κατηγορία ανθρώπων για τους οποίους δεν ισχύουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και υποδαβλίζεται ένα εχθρικό κλίμα των Ευρωπαίων πολιτών απέναντι σε αυτούς, υποδαβλίζεται τελικά τον ακροδεξιό εξτρεμισμό. Ποια είναι η στρατηγική σας για να αντιμετωπίσετε όμως τον ακροδεξιό εξτρεμισμό. Και δεν είπατε ούτε μία κουβέντε για την ανθρωπιστική κρίση στη Μεσόγεια. Από τα τελευταία χρόνια έχουν ε, πνιγεί 35.000 άνθρωποι. Άνδρες, γυναίκες, έφηβοι, παιδιά που έχουν πνιγεί στη θάλασσα. Ποια είναι η στρατηγική σας, τι σκοπεύετε να κάνετε για να δώσετε ένα τέλος επιτέλους σε αυτή την ανθρωπιστική κρίση. Και τέλος, έχουμε την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη βασίζονται ε, ε, και επικεντρώνονται μάλλον στην ε, ποινικοποίηση δραστηριοτήτων οργανώσεων που προσπαθούν να βοηθήσουν και να διασώσουν ανθρώπους από το να πνιγούν στη θάλασσα. Τι θα κάνετε θα φροντίσετε να τερματιστεί αυτή η κατάσταση στα κράτη-μέλη. Θα φροντίσετε οι οργανώσεις ε, διάσωσης στη θάλασσα να βοηθηθούν προκειμένου να μπορέσουν να επιτελέσουν το έργο τους και να φέρουν σε ασφάλεια τους πρόσφυγες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούροκ επίσης έχει ζητήσει το λόγο. κυρία Ρουίς. Κλείνει εδώ ο κατάλογος ομιλητών γιατί όλο είναι και αυξάνεται ο αριθμό των μελών που βρίσκεται στην αίθουσα και ζητάει το λόγο. Ωραία, κυρία Γκόμες, ευχαριστώ πολύ. Συμμερίζομαι ε, αυτή την ε, τοποθέτηση ότι δεν είναι μεταναστευτική κρίση, είναι πολιτική κρίση όπου δεν υπάρχει όχι αλληλεγγύη, ούτε καν σεβασμός ε, προς ε, το κράτος δικαίου και προς τις βασικές αξίε της ιστορίας μας. Με τη σκέψη αυτή να, να ανοίξουμε πλατφόρμες σαν κέντρα κράτηση μεταναστών και προσφύγων εκτό της Ευρώπης, να έχουμε κέντρα κράτηση για τους πρόσφυγες στην Ευρώπη και με την ποινικοποίηση των ΜΚΙΟ. Ακόμα και ο Πάπας πρόσφατα είπε πόσο απαράδεκτη και απάνθρωπη είναι αυτή η πρακτική. Το ερώτημά μου λοιπόν προς εσάς, ε, κύριε Κίκλ, είναι το εξή. Η Ευρώπη που προστατεύει, τι κάνει όταν δεν υπάρχει ασφαλής και νόμιμη δίωδος για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες προς την Ευρώπη. Δηλαδή, ουσιαστικά, συνεχίζεται ε, και δίνεται τα απαραίτητα καύσιμα σε αυτή την αγορά ε, των διακινητών. Δεύτερον, πού είναι η Ευρώπη που προστατεύει όταν οι κυβερνήσει των κρατών μελών δεν δίνουν προτεραιότητα. Ή μήπως θα το κάνει αυτό η δική σας Προεδρία. Θα δώσει προτεραιότητα στο να κλείσουν τα παραθυράκια στις, στη μεταρρύθμιση ΦΠΑ που δίνει ουσιαστικά δισεκατομμύρια ευρώ κέρδη σε εγκληματικές οργανώσεις συμπεριλαμβανομένου και του ISIS. Θα κλείσουν λοιπόν αυτά τα παραθυράκια και μέσω των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μην πηγαίνουν αυτά τα χρήματα στο οργανωμένο έγκλημα και στους τρομοκράτες θα ασκήσετε πιέσει στο Συμβούλιο για Ευρωπαϊκή Μονάδα ε, Χρηματοπιστωτικών Πληροφοριών, που είναι απαραίτητο εργαλείο για να καταπολεμήσουμε το ξέπνιμα βρωμικού χρήματο και την καταπολέμηση τη χρηματοδότηση τρομοκρατία. Εμεί, ε, από ό,τι φαίνεται, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με του πλούσιου ε, μετανάστε, γιατί λέτε ότι δίνεται ηθαγένεια αρκεί κάποιο να κάνει επενδύσει 2 εκατομμυρίων τουλάχιστον. Μπορείτε λοιπόν να μα δώσετε τα στοιχεία ποιοι είναι αυτοί που τους δόθηκε η ηθαγένεια ε, τα τελευταία χρόνια με αντάλλαγμα χρήματα. Και τα πρόσωπα αυτά και ε, οι συγγενείς τους ε, που ήρθαν μέσω της επανένωσης. Ποιον λοιπόν προστατεύει η Ευρώπη τελικά, τους πολίτες ή τους κλεπτοκράτες. Μπορώ να σας δώσω αν θέλετε και στοιχεία με ονόματα από Ουκρανία, από Κρεμλίνο, από τα Βαλκάνια, που ξέρετε ότι έχουν βρει ασφαλή λιμένα στην Αυστρία. Η κυρία Πιόρκα. Ευχαριστώ. Μιλάτε για αλλαγή νοοτροπία και ακούσαμε πολλέ ανησυχίε γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κοιτάξουμε το θέμα της αλληλεγγύης με τους πρόσφυγες, απέναντι στους πρόσφυγες. Θα πρέπει να έχουμε αξιοπρεπή υποδοχή, θα πρέπει να έχουμε διάσωση και ε, έρευνα και διάσωση. Αυτή την αλλαγή πρέπει να προωθήσουμε. Και πρέπει να υπάρχει κατάσταση επίσης. Ε, θα πρέπει να έχουμε ένα ανθρώπινο σύστημα όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση αναλαμβάνει την ευθύνη της απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον πλανήτη και βοηθάει και τις τρίτες χώρες ε, που έχουν προβλήματα προσφύγων. Δεν έχουμε φτάσει τόσο μακριά στις ε, διαπραγματεύσεις. Όταν μιλάμε για αυτές τις, ε, αυτούς τους χώρους ε, αποβίβασης, τους περιφερειακούς χώρους, η κέντρα, η Αυστριακή Προεδρία θα έχει θα προωθήσει την μετεγκατάσταση εκεί σε αυτού του χώρου αποβίβαση. Γιατί αν έχετε αυτό κατά νου, δεν πρόκειται να σα υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ κύριο Πάβελ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εδώ είμαι κύριε Υπουργέ. Θέλω να αναφερθώ σε δύο-τρία πράγματα που δυστυχώς δεν τα λάβατε υπόψη σας ούτε εσείς ούτε οι συνάδελφοί μου. Στην αρχή της ε, τοποθέτησής σας Είπατε ότι είναι πολύ σημαντικό να εξασφαλιστεί αυτή η εταιρική σχέση μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Μιλήσατε πολύ για τη φύλαξη των συνόρων και ε, πραγματικά η Ρουμανία και η Βουλγαρία έχουν τεράστια, τεράστιο μήκος εξωτερικών ε, συνόρων ε, που είναι και πολύ δύσκολο να διαφυλαχθούν από την Ουκρανία μέχρι την Τουρκία εκτείνονται τα σύνορα αυτά. Εμείς λοιπόν έχουμε διαπιστώσει ότι η Βουλγαρία και η Ρουμανία έχουν κάνει ε, τα μαθήματά τους, έχουν ε, εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους. Παρ' όλα αυτά δεν είναι μέλη του χώρου Σέγγεν. Θα μπορούσατε βεβαίως εσείς, αν αναλάβετε σχετικές πρωτοβουλίες, να ε, εντάξετε ή να διευκολύνετε την ένταξη των χωρών αυτών στο χώρο Σέγγεν. Τι θα κάνετε. Δεύτερον, οι δύο αυτές χώρες έχουν ξεχωριστό μηχανισμό για τη συνεργασία και την επαλήθευση. Εδώ και ένα χρόνο έχουμε καταλήξει, έχουμε θεσπίσει πλέον 12 νομοθετήματα, η Βουλγαρία δηλαδή, η Ρουμανία δεν ξέρω, ε, τα οποία και άπαξ και υλοποιηθούν. Μπορείτε εσείς να με, να με διαβεβαιώσετε δεν μπορείτε βεβαίως να δεσμεύσετε και τα 28 κράτη-μέλη, αλλά εσείς ως υπουργό μπορείτε να με διαβεβαιώσετε ότι θα καταλήξουμε πολύ σύντομα σε έναν ενιαίο μηχανισμό που θα αφορά και τις 28 χώρες ε, και όχι μόνο ε, τις 26 και κάποιες να εξαιρούνται. Πιστεύετε ότι θα το καταφέρουμε εντό τη Προεδρία σα. Επίση, είπατε ότι πρέπει να δοθεί νέο ορισμό στην αλληλεγγύη. Πραγματικά έχω πολύ μεγάλη αγωνία και δεν θα πω τίποτα παραπάνω για το πού θα καταλήξουμε. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γιαρόκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορη. Ευχαριστώ και τους δύο υπουργούς που μας μίλησαν για τα σχέδιά τους, πολύ φιλόδοξα. Ε, ακούσαμε και την προηγούμενη, την εβδομάδα τον κύριο στην Ολομέλεια. Αλλάζουν τα δεδομένα. Καλή τύχη λοιπόν. Η τρομοκρατία και η διαφθορά, όπως είπατε, είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει πολύ προσεκτικά. Ως Αντιπρόεδρος για τα Βαλκάνια εντός του Κοινοβουλίου θα ήθελα να σας επιστήσω την προσοχή στο εξή. Σε ένα από τα σημεία ε, από τα 10 που ετοίμασε η ΛΥΜΠΕ για το δίκτυο δράσης κατά της ε, ισοσπαστικοποίησης. Είναι μια εκστρατεία ενημερωτική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί δεν πρέπει να κάνετε τίποτα εάν δεν ε, καταλάβετε πόσο προωθείται η ριζοσπαστικοποίηση στους στοχούς της Ευρώπης. Έχουμε 100 εκατομμύρια φτωχού στην Ευρώπη. Ε, υποτίθεται ότι την προηγούμενη, με την προηγούμενη στρατηγική για τους Ρωμά ε, κάναμε κάτι για αυτούς τους ανθρώπους. Ε, τώρα είναι η δική σας Προεδρία και έχετε το, τη σκητάλη για να κάνετε κάτι παραπάνω. Όχι μόνο για τη ριζοσπαστικοποίηση ε, γεννάτε στη φτώχεια, αλλά υπάρχουν εκατομμύρια νέων ανθρώπων δεύτερης-τρίτης γενιάς, μερικοί από αυτούς γεννήθηκαν εδώ και είναι ανικανοποίητοι αυτό το project ε, θα ήταν τέλειο γιατί έχουμε ακόμα τρεις τρία χρόνια πόρους για να καταπολεμήσουμε τη ριοσπαστικοποίηση. Επίσης, έχετε και την ε, στήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα μειονότητας, γιατί από όλα τα λεφτά τα 7 εκατομμύρια είναι για τις μειονότητες. Στην ε, Ουγγαρία. Ας πούμε, η Ρουμανία και η Ουγγαρία έχουν τεράστια θέματα με τις μειονότητες ημέν των ΔΕ, ας πούμε. Δεν μπορείς να αγοράσεις σε πόλεις, ας πούμε, που ε, ρουμάνικες που ζουν κυρίως ε, Ούγγροι, δεν μπορείς να αγοράσεις, ας πούμε, να πας στο σιδηροδρομικό σταθμό και να αγοράσεις σιτήριο στα Ουγγρικά. Δεν μπορείς να μιλήσεις αυτή τη γλώσσα. Και αντίθετα, δεν μπορείς να βάλεις, ας πούμε, σημαίες ε, ρουμάνικες ε, στην Ουγγαρία. Σας ευχαριστώ, είναι τεράστιο το θέμα. Και σας ευχαριστώ για την ε, προσπάθεια που κάνετε για την κοινότητα του, των Ρωμά στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Χαίρομαι πολύ που... Είναι και οι δύο υπουργοί εδώ. Είναι μια τεράστια ικανοποίηση για μας. Ε, ακούσαμε στο Στρασβούργο και την παρέμβαση του καγκελάριου σας, ο οποίος μίλησε για εκείνη την Ευρώπη η οποία προστατεύει, αλλά και που σέβεται τις διαφορές. που είναι και η βάση του πολιτισμού μας. Μία από τις προκλήσεις που ε, μας ε, αντιμετωπίζουν που αντιμετωπίζουμε είναι να λάβουμε υπόψη μα αυτέ τι ε, διαφορέ. Θέλω να κάνω μια έκκληση στην Αυστριακή Προεδρία, ούτω ώστε να παίξει ένα θετικό ρόλο στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, κυρίω όταν βλέπουμε αυτού του ανταγωνισμού του εθνικού. Ε, Παραδείγματο χάρη σε αυτέ τι διαδικασίε εναντίον τη Πολωνία ή τη Ουγγαρία. Δεν θέλω να μιλήσω για την Πολωνία, τη χώρα μου, γιατί θα μου πείτε ότι δεν θα είμαι αντικειμενικό όταν μιλάω. Α μιλήσουμε όμω για του Ούγγρου. Για του Ούγγρου που του επιτίθενται. Γιατί προστατεύονται, προστατεύουν τα σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουγγαρία προστατεύει αυτά τα νότια σύνορα, τα εξωτερικά σύνορα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και γι' αυτό δέχεται επιθέσει. Θα ήθελα λοιπόν να πω στην Αυστριακή ε, Προεδρία να παίξει ένα θετικό ρόλο στο Συμβούλιο για να ηρεμήσουν λιγάκι αυτές οι εντάσεις που υπάρχουν. Ε, το Συμβούλιο δεν θα έπρεπε να γίνει ένα φόρουμ όπου υπάρχει απλώς ανταγωνισμός ανάμεσα στα έθνη. Και αυτό το λέω γιατί οι προσωπικέ μου πεπιθήσει, και τώρα α μιλήσω για την Πολωνία λιγάκι, είναι ότι για την Πολωνία ε, υπήρχε έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και περιμένουμε υπομονετικά ε, την ετοιμιγορία. Όταν λειτουργεί μια δημοκρατία, θα πρέπει να ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας, έτσι. Και ελπίζω να μην υπάρχει στο τέλος αυτής της πορείας α, κίνδυνος για τη δημοκρατία. Είναι ένας από τους α, μηχανισμούς που πρέπει να προωθήσουμε. Επίσης, ε, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην αρχή της μεταναστευτικής κρίσης πήρε μία απόφαση για να καταπολεμήσει την ε, λαθρομετανάστευση εν το γενάστε της, ε, εκεί όπου δημιουργείται. Και τώρα βλέπουμε ότι αυτή η λαθρομετανάστευση μπορεί να γίνει προπομπός της νόμιμης μετανάστευσης. Είναι παράλογο αυτό το πράγμα και ελπίζω επί Αυστριακής Προεδρίας το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να ξαναπαίξει το ρόλο που έχει για να προστατεύσει την Ένωση. Γιατί η Ένωση είναι ε, Ένωση κρατών και όχι Ένωση ιδεολογιών ή ποιονδήποτε τέλος πάντων, ένα συνοθήλευμα ιδεολογιών. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα θερμό ευχαριστώ προς τους Υπουργούς. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να σας ακούω, οι περιγραφές σας, οι φιλοδοξίες που έχετε για τους επόμενους έξι μήνες. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη σε εσά και περιμένω να δω με υπομονεσία πώ θα προωθήσετε αυτά τα θέματα. Μιλήσατε για την Ευρώπη που προστατεύει. Είμαι Σουηδέζα. Και νομίζω ότι είναι ανθρώπινο δικαίωμα να αισθάνεσαι ασφαλή στη χώρα σου. Και δεν ξέρω αν πραγματικά αισθάνομαι ασφαλή πια στην χώρα μου. Γιατί στη Σουηδία, α πούμε, είδαμε τι επιπτώσει σε περιοχές όπου υπάρχει αποκλισμός, υπάρχουν παράνομα όπλα τα οποία χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν ανθρώπους, ε, γυναίκες βιάζονται, άνθρωποι βιάζονται. Δεν αισθανόμαστε ασφαλείς στην ε, Σουηδία. Χαίρομαι λοιπόν που βάζετε το θέμα της ασφάλειας στην ατζέντα. Επίσης, διαρωτώ με, τι είδους φραγμούς βλέπετε να υπάρχουν στην προσπάθεια και εμπόδια που υπάρχουν στην προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε αυτά τα εξωτερικά σύνορα. Σκέφτομαι αυτά τα παράνομα όπλα που εισραίουν στην Ευρώπη. Συγγνώμη, αλλά κάντε, θορυβείτε πάρα πολύ. Μπορείτε να ησυχάσετε επιτέλους για να μιλήσω. Το σκεφτήκατε αυτό. Ε, τι εντολή θα λάβει η Frontex. Η Frontex ε, αυξάνει τον προπολογισμό της σύντο χρόνο. Ε, και ο περισσότερο προπολογισμό πηγαίνει για επιχειρήσει έρευνα και διάσωση. Θα πρέπει επιτέλου ε, να εξασφαλίσουμε ότι όλοι αυτοί που πνίγονται στη Μεσόγειο. ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η ιστορία, θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Κάτι πρέπει να γίνει επιτέλου. Το να έχουμε κέντρα ασύλου και άτομα τα οποία είναι θύματα βιασμού και βασανιστήριων ε, αν τα στήσουμε θα πρέπει να μας βοηθήσει και ο ΙΕ. Πώς θα τα επιλύσετε αυτά τα θέματα στην Αυστραλία. Εκεί θα επιλύθουν αυτά τα θέματα. Τελευταίος. Ο μιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ένα από τα πράγματα που είπατε με ενόχλησε. Ε, μιλάμε για την προστασία των ευρωπαϊκών αξιών, έτσι και το δικαιωμάτων των, ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι καθολικά δικαιώματα. Η αλλαγή νοοτροπίας τώρα, είναι η ερώτησή μου, τι σημαίνει. Ε, δηλαδή, ε, αυτά τα δικαιώματα έχουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και αυτοί που μπορούν να αγοράσουν τις χρυσές ε, θεωρήσεις μόνο. Εάν αυτή η αλλαγή της ε, νοοτροπίας είναι αυτή, θα χάσουμε αυτές τις αξίες στο μέλλον. Ε, θα σας ρωτήσω το εξή. Το μοντέλο της Λιβύης είναι το κατάλληλο μοντέλο για να πετύχετε αυτή την αλλαγή της νοοτροπίας, γιατί αν ναι, τότε μπορεί να διαπιστέσουμε ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και η ανθρώπινη αξιοπρέπεια είναι για κάποιους, όχι για όλους. Σας απασχολείτε ότι γίνεται στη Λιβύη, γιατί υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή. Διπλασιάζεται το, ο αριθμός των πνιγμένων σε κάποιες μεσογειακές οδού, οδούς και διπλασιάστηκε ε, ο αριθμός των ατόπων που επιστρέφονται στη Λιβύη όπου βιάζονται και βασανίζονται, το ξέρουμε αυτό. Τι θα κάνετε για το θέμα αυτό, για το θέμα της Λιβύης. Mm. Όπως ακούσατε, Υπουργοί, τα μέλη μας σας έθεσαν ε, πολλά ερωτήματα και είναι υψηλές οι προσδοκίες των μελών από την Αυστριακή Προεδρία, γιατί είναι η τελευταία ευκαιρία ε, επίτευξη αποτελεσμάτων πριν από τις ευρωεκλογέ. Ε, βλέπετε ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ε, και πολυμορφία και καταφέρνουμε παρόλα αυτά να προχωρήσουμε, να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε ένα σημαντικό πακέτο. Πολλά από τα ερωτήματα λοιπόν, που σας επέβαλαν τα μέλη αφορούν αυτό το πακέτο του ασύλου ε, για την προστασία και την αίσθηση ασφαλείας των Ευρωπαίων πολιτών, χωρίς βέβαια ε, να παραμελούμε και τις διεθνείς ε, υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ ένα ερώτημα το οποίο έθεσε ο κύριος Πάβελ προηγουμένως. Πριν έρθετε στην Επιτροπή μας, εξετάσαμε μία έκθεση που θα ψηφιστεί ε, στο Κοινοβούλιο για την ε, πλήρη προσχώρηση της ε, Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ζώνη Σένγκεν. Εφτά χρόνια έχουν περάσει από τότε που πλήρωσαν τα κριτήρια προσχώρηση τη ζώνη Σένγκεν αυτές οι δύο χώρες, αλλά ακόμα δεν έχουν μπει στην ζώνη Σένγκεν. τι ακριβώς θα κάνετε με αυτή τη διαδικασία. Έχετε το λόγο. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα να σα ευχαριστήσω θερμότατα για τι ερωτήσει που μου θέσατε και να πω εξ αρχή ότι αυτό που είπε η Ευρωβουλευτή Μλίνα όσον αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτο δικαίου αποτελούν βασική προτεραιότητα τη Αυστρική Προεδρία. Εγώ, ε, ξέρετε, είχα την δυνατότητα και την ευκαιρία στη ζωή μου να είμαι Γενικό Εισαγγελέα και πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 12 χρόνια στη χώρα μου και στόχο μου ήταν πάντοτε η ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη και η ασφάλεια ε, του δικαίου. Γι' αυτό και εγώ ε, είμαι μαχητής του κράτους δικαίου. Όμως για την υλοποίηση των αρχών του κράτους δικαίου απαιτείται αμοιβαία εμπιστοσύνη. Αυτό τι ακριβώς είναι η οδός που θα ακολουθήσει η Αυστριακή οδός. Η επόμενη άτυπη σύνοδος των Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων θα γίνει 13 και 14 Ιουλίου και εκεί στην ημερήσια διάταξη θα υπάρχει σχετικό θέμα, rule of law, κράτος δικαίου, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στα συστήματα δικαιοσύνης μας προκειμένου να εξασφαλιστεί η αμοιβαία εμπιστοσύνη, η αμοιβαία αναγνώριση αποφάσεων προκειμένου να καταλήξουμε σε μια κοινή πορεία, πορεία όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωση ε, στα ζητήματα που αφορούν για παράδειγμα την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, τα ευρωπαϊκά, το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης κτλ. Και γι' αυτά θα πρέπει να, δοθεί, ε, να σημειωθεί προόδος και στον τομέα των ηλεκτρονικών ενδείξεων. Αν όμω θέλουμε πραγματικά να επιτύχουμε όλου αυτό, αυτούς τους στόχους, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι ο διάλογος θα διενεργείται και θα διεξάγεται σε ένα περιβάλλον ε, που περιγράφεται και από τι αποφάσει του Ευρωπαϊκού ε, Δικαστηρίου. Πρέπει να εξασφαλίζονται κοινέ προσπάθειες και κοινή στόχοι. Σε αυτήν την διαδικασία λοιπόν εντάσσεται όλο το πρόγραμμα εργασιών της Αυστριακή Προεδρία, όχι μόνο αυτή η άτυπη σύνοδο των Υπουργών δικαιοσύνη. Τον φθινόπωρο, τον Οκτώβριο, με την Κομισιόν συνδιοργανώνουμε εκδήλωση πάλι με το συγκεκριμένο θέμα ως επίκεντρο της προσοχή μας, το κράτος δικαίου, ταυτόχρονα και στις επαφές μας με τα άλλα κράτη-μέλη αλλά και με τα κράτη των Δυτικών Βαλκανίων έχουμε παντού και πάντοτε το θέμα αυτό στο επίκεντρο της, προσοχή της προσοχής μας. Θέλουμε στο τέλος της Προεδρίας μας να καταλήξουμε σε συμπεράσματα του Συμβουλίου στα οποία θα δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα του κράτους δικαίου. Όσον αφορά την Πολωνία, θέλω να σας πω ότι στις 26 έκτου έγινε ακρόαση στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων για το θέμα αυτό και ο Επίτροπος Τίμερμανς σημείωσε ότι θεωρεί ότι εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνος σημαντικής παραβίασης των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ότι θα γίνει στις 18 Ενάτου έκτακτη σύνοδος με αυτό το θέμα και μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι παρακολουθούμε αυτό το θέμα στενά σε συνεργασία με την Κομισιόν και τις νομικές υπηρεσίες των θεσμικών μας οργάνων και ελπίζω ο διάλογος τον οποίο επιδιώκουμε θα καταφέρει να ε, εξασφαλίσει τις αρχές του κράτους δικαίου και σε αυτά τα κράτη-μέλη. Πρόκειται ε, άλλωστε υπάρχουν 11 κράτη-μέλη τα οποία έχουν δηλώσει την προθυμία τους να συνεχιστεί αυτός ο διάλογος. Και ξέρετε ο διάλογος αυτός δεν αφορά μόνο την Πολωνία, αφορά και άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και αφορά εν γέννη το ερώτημα πώς μπορεί να διευρυνθεί και να εμβαθυνθεί η εφαρμογή του κράτους δικαίου, πώς μπορούμε να βρούμε συγκεκριμένους μετρήσιμους δείκτες βάσει των οποίων θα μπορούμε να επαληθεύουμε την εφαρμογή του κράτους δικαίου. Είπε ο κύριος Αγγιλάρ, πρέπει κάτι να γίνει. Βεβαίως, αυτό αφορά όμως και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Και σα καλώ από αυτό το βήμα να στρέψουμε το βλέμμα μας προς το μέλλον της Ευρώπης και να εργαστούμε σκληρά πάνω στους φακέλους που έχουμε ήδη δουλέψει. Διότι αν έχουμε μια κοινή στάση η οποία θα εξασφαλίζει και την ασφάλεια της Ευρώπης αλλά και την αποτελεσματικότητά ξέρετε ότι μπορούμε να επιτύχουμε πολλά. Αυτό ε, το, αποδεικνύει, ε, το αποδεικνύει και η δουλειά μας ε, σε μια σειρά από που ήδη έχουν ολοκληρωθεί με επιτυχία. Το ίδιο τα ίδια αφορούν και την ηλεκτρονική ιδιωτικότητα. Όμω ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά εκκρεμή ερωτήματα, όπω είναι για παράδειγμα η χρησιμοποίηση των cookies, οι επιπτώσει σε, κανε... σε καινοτόμε υπηρεσίε, στι μικρομεσαίε επιχειρήσει τη Ευρώπη. Και ξέρετε ότι κάποια κράτη-μέλη θεωρούν ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις, στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά κράτη-μέλη θεωρούν ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη που θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή ε, το έγγραφο βάσει του οποίου συζητούμε δεν είναι επαρκής και πρέπει να διευρυνθεί και να υποβληθεί σε περαιτέρω επεξεργασία. Μπορώ εγώ να σας διαβεβαιώσω ότι θα γίνουν κάθε προσπάθεια από πλευρά Αυστριακή Προεδρία προκειμένου να ε, σημειωθεί πρόοδο. Έχουμε ήδη προγραμματίσει συνεδριάσει ε, των ε, σχετικών ομάδων εργασία μέσα στον, Ιούλιο. Είπατε και για, για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματο. Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε να μην υπάρχει ένα forum shopping, μια ε, μετακίνηση των, δια, ενδιαφερομένων από το ένα κράτος μέλος στο άλλο κράτος μέλος, προκειμένου να βρουν τις, ε, εκείνες τις χώρες που οι ρυθμίσεις τους τους βολεύουν κάθε φορά. Πρέπει να εναρμονιστεί το πλαίσιο και όσον αφορά τις κυρώσεις για την νομιμοποίηση παράνομων εσόδων. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ήδη πολλά επιτύχει, όμως πλέον αυτό που μένει να επιτύχουμε είναι και οι υπόλοιποι στόχοι που έχουμε δώσει όλοι μαζί από κοινού και σε αυτό το πλαίσιο θεωρώ ότι το Συμβούλιο του Οκτωβρίου θα στεφθεί με επιτυχία. Επίσης, έγινε αναφορά στο πρόγραμμα δικαιοσύνη. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί συζητήσει για μια σειρά αποζητήματα γύρω από τη δικαιοσύνη, όπω είναι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Έχει υπάρξει θέση σε εφαρμογή διαφόρων νομοθετημάτων που έχουν θεσπιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό που απομένει τώρα να γίνει είναι να εκαταρτιστούν και να εκπαιδευτούν οι δικαστές όλη η δικαστική λειτουργία στα κράτη-μέλη και όχι μόνο ε, οι δικαστές, όλοι όσοι εμπλέκονται στη διαδικασία της απονομής τη δικαιοσύνης να καταρτιστούν και να εκπαιδευτούν στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου ακριβώς για να ενισχυθεί η απονομή της δικαιοσύνης. Θέλουμε ενίσχυση της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ δικαστικών αρχών των κρατών μελών και ε, θέλουμε να ενισχύσουμε και να εμβαθύνουμε αυτό που είπατε και εσείς, το δίκτυο, το EJN, το, το δίκτυο για την κατάρτιση και τη μετεκπαίδευση δικαστικών λειτουργών. Γι' αυτό και προβλέπουμε και ε, κονδύλια, να προτείνουμε κονδύλια για την... Ε, για, την, για το δίκτυο αυτό. Διότι αν θέλουμε πραγματικά να ενισχύσουμε την έννοια του κράτου δικαίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προβλέπονται και τα αντίστοιχα κονδύλια. Και σα διαβεβαιώ ότι εμεί θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μα ε, προς αυτή την κατεύθυνση. Είπα λοιπόν ότι ο κράτο δικαίου είναι όχι απλά ένα, ε, ένα ε, παρεμπίπτον θέμα αλλά βασικό θέμα που μα απασχολεί. Και ακριβώ θέλουμε να θεσπίσουμε μέτρα προκειμένου και οι αρχέ επιβολή του νόμου να έχουν τι απαραίτητε σε εκείνε πληροφορίε προκειμένου να μπορούν να εκτελούν τα καθήκοντά του ξέρετε ότι οι εγκληματίες γίνονται όλο και πιο ικανοί. Ξέρετε ότι οι, οι, επικοινωνίες μεταξύ εγκληματιών γίνονται όλο και πιο ψηφιακές. ο χώρος και ο χρόνος έχει συμπυκνωθεί. Γι' αυτό και πρέπει οι αρχές επιβολής του νόμου, οι διοκτικές αρχές να έχουν τη δυνατότητα ταχύτατα να έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε ε, αναγκαίες πληροφορίες και μέσω υπηρεσιών ε, διαδικτυακού νέφους. Μάλιστα αυτή την κατεύθυνση βρισκόμαστε στις επαφές με τις ΗΠΑ. Το θέμα αυτό έχει ήδη θα συζητηθεί μάλλον και ατύπως στο, τον Ιούλιο στην ε, Υπουργική Διάσκεψη όπου και θέλουμε να γίνει μια γενική συζήτηση προς ανατολισμού, ώστε τον Οκτώβριο ε, να καταλήξουμε σε κάτι πιο συγκεκριμένο στην, ε, στο Συμβούλιο και το Δεκέμβριο σε συμπεράσματα του Συμβουλίου και ελπίζουμε να έχουμε την συμβολή σας σε αυτή τη διαδικασία. Ένα θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Ευρωβουλευτής Αγγιλάρ. Πραγματικά πρέπει... Ε, Ε, για, την, ε, για, την, ε, για τις ηλεκτρονικές ενδείξεις. Εδώ είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να γίνει μία συζήτηση και για δακτυλικά αποτυπώματα και για βιομετρικά δεδομένα και τις επόμενες μέρες 13 ε, Εβδόμου στην άτυπη ε, Σύνοδο Υπουργών θα γίνει αυτή η ε, σχετική συζήτηση και στις 18 Εβδόμου θα συζητηθεί το θέμα αυτό και ελπίζουμε το συντομότερο δυνατό να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, προκειμένου να δοθεί και μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου για τις διοκτικές αρχές. Πραγματικά σας διαβεβαιώ ότι στον τομέα της δικαιοσύνης κάνουμε πολύ μεγάλες προσπάθειε να εναρμονιστούν τα πρώτα πρότυπα στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί αυτή είναι η μόνη μα ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο αν καταφέρουμε να εξασφαλίσουμε εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και συνεργασία. Και γι' αυτό θέλω να σα καλέσω να συνεργαστούμε από κοινού και στους τομείς που άπτονται της δικαιοσύνης ε, και να ε, έρθουμε σε ειλικρινείς και ανοιχτές μεταξύ μας διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ε, Κύριο Κλίκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω καταρχάς για το ενδιαφέρον που επιδείξατε για το, για το πρόγραμμα εργασιών της μελλοντική μας Αυστριακής Προεδρίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω ακόμα και για τα ερωτήματα που εμπεριείχαν, αν θέλετε, μια κριτική. Είναι πάντοτε χρήσιμα και ωφέλιμα τέτοιου είδου ερωτήματα. ακριβώ γιατί δείχνουν ότι σε κάποια θέματα τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση οδηγήθηκε σε αδιέξοδο, κάτι που πρέπει να μα οδηγήσει βεβαίω και στην διαπίστωση ότι πρέπει να βγούμε από το αδιέξοδο αυτό. Ένα ερώτημα που μας απασχολεί όλους και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα να το πω εδώ σε αυτό το βήμα. Σε κανέναν δεν αρνούμε το δικαίωμα να επιθυμεί μια καλύτερη Ευρώπη όσο και αν διαφωνούμε, όσο και αν διαφωνώ. Βεβαίως σε κάθε οικογένεια χρειάζεται να γίνει συζήτηση και διάλογος για να καταλήξουμε σε συγκεκριμένη δράσεις. Πάντως, μπορώ να σας επιβεβαιώσω και να σας διαβεβαιώσω ότι η Αυστρία θα λειτουργήσει ως γεφυροποιός τους επόμενους ε, έξι μήνες. Αλλά το να προσπαθεί κανείς ε, να ε, γεφυρώσει ένα ποταμό σημαίνει ότι πρέπει πάντοτε τα έργα του να ξεκινήσουν από τη μία όχθη. Δεν μπορεί κανείς να ξεκινήσει από τη μέση του ποταμού. Θα απαντήσω τώρα με περισσότερη λεπτομέρεια ε, στα ερωτήματά σας. Ρωτήσατε για τις αξίες, την τήρηση των βασικών αρχών και αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την υπεράσπισή τους. Για μένα προσωπικά ε, είναι αυτονόητο αυτό. Κανείς δεν αμφισβητεί την Χάρτα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, κανείς δεν αμφισβητεί την Σύμβαση των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, διότι ε, εμείς είμαστε σε τελική ανάλυση αυτοί που είμαστε και εγγυητέ αυτών των ε, συμβάσεων και διακηρύξεων. Γι' αυτό και θα καταβάλουμε ε, σε, σε όλα τα φόρα, σε όλα τα βήματα προσπάθειες να τηρήσουμε, να συμβαστούμε, να διαφυλάξουμε τις αξίες αυτές. Το ερώτημα λοιπόν είναι ποιος ποια, ποιο είναι το μεγαλύτερο αμάρτημα ε, σε σχέση με τις αξίες μας. Γιατί ακούστηκε αυτός ο όρος. Θεωρώ ότι το μεγαλύτερο αμάρτημα σε σχέση ε, με τις αξίες μας είναι το να πνίγονται χιλιάδες άνθρωποι στη, Μεσά, ε, στη Μεσόγειο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων από τον θάνατο ενός ανθρώπου που θα μπορούσε να είχε ζήσει. Γι' αυτό και μίλησα για μεταστροφή, για αλλαγή νοοτροπίας. Διότι το ερώτημα που πρέπει να μας απασχολήσει είναι πώς τελικά θα προχωρήσουμε στη διαχείριση αυτής της μεταναστευτικής και προσφυγικής κρίσης. Και για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζεται να σπάσουμε, ε, για να, να εξαρθρώσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Εκεί είναι λοιπόν που χρειαζόμαστε συνεργασία. Όχι να πλήξουμε και να καταδιώξουμε αυτούς που έρχονται στην Ήπειρό μας, αλλά εκείνους που βγάζουν χρήματα από αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι το μεγάλο αμάρτημα που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να καταπολεμηθεί τώρα, τώρα και γι' αυτό ακριβώς απαιτείται αυτή η μεταστροφή στην οποία αναφέρθηκα. Ακούστηκε το ερώτημα τι θα γίνει με αυτές, με αυτές τις πλατφόρμες αποβίβασης στη Βόρεια Αφρική. Καταρχάς να σας πω ότι δεν πρόκειται για δική μας ε, καινοτομία, αλλά ε, για πρόταση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η εντολή ήταν πώς θα μορφοποιηθεί στην πράξη αυτή η ιδέα. Γνωρίζουμε και από το παρελθόν ότι τα μοντέλα που έχουν υλοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν μας οδήγησαν στο επιθυμητό επίπεδο. Γι' αυτό και σε κάποιους τομείς χρειάζεται να σκεφτούμε και με μια ορισμένη ε, ευελιξία και καινοτομία. Γι' αυτό και τον, το την Πέμπτη στο Ίνσπρουκ θα γίνει η πρώτη άτυπη σύνοδο Υπουργών δικαιοσύνη, όπου και θα συζητηθεί διεξοδικά το θέμα αυτών των πλατφορμών αποβίβαση. Αυτά από, από τα όσα θα ακουστούν και από τους υπόλοιπου υπουργού, θα εξαρτηθεί και η περαιτέρω δουλειά μα σε συνεργασία με ευρωπαϊκού οργανισμού, με την ύπατη αρμοστία του ΟΗΕ για του πρόσφυγε, αλλά και με τρίτε χώρε για το πώ ακριβώ, τι μορφή θα, μπορεί, ε, θα μπορούσε να πάρει αυτή η ιδέα για τι πλατφόρμε αποβίβαση. Δεν καταλαβαίνω γιατί είστε απεσιόδοξοι. Εγώ γενικά ω άνθρωπο είμαι φύση αισιόδοξο. Άκουσα ότι κάποιοι είπατε ότι οι αφρικανικέ χώρε είναι εκείνε που ήδη έχουν απορρίψει αυτό το μοντέλο. Μα δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο. Περιμένετε να δούμε ε, πώς, τι μορφή θα πάρει τελικά αυτή η πρόταση. Και από εκεί και πέρα θα μπορέσουμε να αρχίσουμε να μετράμε τα αποτελέσματα που θα αποφέρει η ιδέα αυτή και να γίνει ένας απολογισμός. Όσον αφορά την... το Δουβλίνο τώρα και το συνολικό πακέτο. Εγώ αναγνωρίζω πλήρως την ε, αξία αυτού του πακέτου του Δουβλίνου. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικό να καταλήξουμε σε ενιαίες προδιαγραφές, σε ενιαία πρότυπα, στην, ε, στον ορισμό ενιαίων και κοινών αρμοδιοτήτων ευθυνών προκειμένου να εξασφαλιστεί η σταθερότητα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου. Γι' αυτό άλλωστε είναι και δική μας θέση το πακέτο αυτό να το συζητήσουμε από κοινού με εσάς και εκεί όπου δεν υπάρχει ακόμα ενιαία στάση στο Συμβούλιο να εργαστούμε πάνω στη βάση του έργου που μας ε, άφησε ως παρακαταθήκη η Βουλγαρική Προεδρία, να προχωρήσουμε στις απαραίτητες αναλύσεις και να προχωρήσουμε στις ε, αναγκαίες κινήσεις ώστε να βγούμε από τα διέξοδα στα οποία έχουμε ε, οδηγηθεί. Όμως, μ' αρέσει και η ειλικρίνεια. Και πρέπει να είμαστε ειλικρινεί με τον εαυτό μα. Όταν μιλούμε για το Δουβλίνο, και εδώ πρόκειται για απόφαση και εντολή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να προχωρήσουμε σε κάτι απτό και συγκεκριμένο, έγκαιρα και γρήγορα, θα πρέπει να έχουμε ξεκάθαρο ότι πρόκειται για ένα θέμα που αφορά τον καταμερισμό των ευθυνών. Και αυτό είναι άλλωστε και ο λόγος που οι προσπάθειες αυτές δεν έχουν ακόμη στεφτεί με επιτυχία. Από αυτή λοιπόν την ειλικρινή αν θέλετε αξιολόγηση και ανάλυση της πραγματικότητας πρέπει να αρχίσουμε για να καταλήξουμε σε μια αναζωογόνηση αν θέλετε της έννοιας της αλληλεγγύης. Διότι η αλληλεγγύη δεν είναι ε, ε, δεν ε, ισούται μόνο με τον καταμερισμό και την κατανομή των προσφύγων. Μα δεν αφορά μόνο αυτό το ερώτημα, το ζήτημα της αλληλεγγύης. Μιλάμε για τη διάσωση στη θάλασσα, για τη φύλαξη των εξωτερικών συνόρων. Υπάρχουν πολλοί πολλά δομικά στοιχεία αν θέλετε τα οποία θα ε, συνδιαμορφώσουν την τελική εικόνα. Η τελική εικόνα η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι ικανοποιητική για κανέναν και φαντάζομαι ότι συμφωνείτε μαζί μου σε αυτό. Για την επανεγκατάσταση. Είπατε ότι η Αυστρία επανεγκατέστησε 44 ανθρώπους. Ναι, πράγματι, αυτό άλλωστε προέβλεπε σχεδόν η ποσόστοσή μας. Αυτό που ε, πράγματι ε, ισχύει είναι ότι δεν έχουμε πολύ μεγάλο ποσοστό αναγνωρίσεων. Αλλά δεν νομίζω ότι η Αυστρία είναι μια χώρα την οποία μπορεί κανείς να κατηγορήσει για έλλειψη αλληλεγγύης εν ώψη ε, και λαμβάνοντας υπόψη την ε, μεταναστευτική κρίση του 2015. Και μια τελευταία παρατήρηση για αυτές τις πλατφόρμες αποβίβασης. Προφανώς και θα απαιτηθεί ε, οι γειτονικέ μας χώρες να ε, αναλάβουν τις ευθύνες τους και να, τις, να, τους υπενθυμίσουμε τις ευθύνες τους. Εδώ θα πρέπει πραγματικά να αξιοποιηθούν διάφορα εργαλεία και οικονομικής πολιτικής αν θέλετε ή εξωτερικής πολιτικής προκειμένου να καταλήξουμε σε ένα σύστημα που θα είναι αμοιβαία εποφελές. Επίσης έγινε λόγος για τις θέσει Ζέχοφερ. Εξ όσων γνωρίζω εγώ και από όσα ξέρω από συζητήσει μου με τον ίδιο τον κύριο Ζέχοφερ, αυτή τη στιγμή υπάρχουν διαπραγματεύσεις μεταξύ Γερμανίας και χωρών που, ε, από τις οποίες προέρχονται οι πρόσφυγες. Μιλάμε δηλαδή για την Ιταλία και την Ελλάδα συγκεκριμένα. Θα δούμε τώρα τι θα προκύψει, αλλά αυτοί, εκείνοι είναι αρμόδιοι και θα δούμε πού θα οδηγηθούν οι διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά τις απελάσεις ε, ε, ανθρώπων που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν το σύστημα ασύλου, αυτό δεν αφορά απλώς την ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά την εσωτερική πολιτική των κρατών μελών. Υπάρχει όμως μια πρόταση ε, στην οδηγία η επιστροφή έστω και προσωρινή στη χώρα καταγωγής να μπορεί να αποτελέσει λόγο για την άρνηση παροχής ασύλου. εγώ συμφωνώ με την πρόταση αυτή. Είπατε ότι δεν έχουμε πια να κάνουμε μεταναστευτική κρίση. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο είναι πολύ πρόωρο για να το πείτε. Σας θυμίζω ότι το 2015 υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν κρούσει τον κόδωνα του κινδύνου και είχαν πει ότι μπορεί οι μηχανισμοί μας να μην καταφέρουν να ανταποκριθούν στη σοβαρότητα της κατάστασης. Και υπήρχαν άνθρωποι, και σε αυτούς συγκαταλέγομαι και εγώ, που κατηγορήθηκαν ως ε, κινδυνολόγοι. Εγώ πριν από 14, 14 ε, μέρες είχα συνάντηση με τον κύριο Αβραμόπουλο και τις, ε, τους εκπροσώπους των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων και πρέπει να σας πω ότι η εικόνα είναι πολύ διαφορετικά και, διαφορετική σε αυτούς τους ανθρώπους και, και μιλάω μόνο για έναν διάδρομο μετανάστευσης. Εκεί ακούσαμε ότι υπάρχουν υπάρχει ένταση του προβλήματος, όξυνση του προβλήματος και, και ότι υπάρχει ανάγκη να ληφθούν μέτρα άμεσα για να αποφευχθεί μια κατάσταση όπως αυτή που δημιουργήθηκε το 2015. Γι' αυτό και χρειάζεται προδραστικά να αναλάβουμε μέτρα και κινήσεις τώρα, προκειμένου να αποφύγουμε τα χειρότερα. Κέντρα ασύλου σε τρίτες χώρες. Αυτό που πρέπει να πετύχουμε είναι να, να καταπολεμήσουμε όλους εκείνους τους παράγοντες που δρούν ε, ως ε, ε, ελκυστικοί παράγοντες για την, για την προσέλκυση ανθρώπων εδώ στη, στην Ευρώπη. Για να μπορέσουμε πραγματικά να εξασφαλίσουμε ότι θα δοθεί βοήθεια και αρρωγή σε εκείνους που τη χρειάζονται. προβλέπετε πλέον ότι θα ε, ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μένουν έως τέσσερις εβδομάδες σε αυτές τις πλατφόρμες. Δεν νομίζω ότι μπορεί κάτι τέτοιο να το, να το ε, εξισώσει κανείς με κέντρα κράτησης όμως. Υπόθηκε, ε, μάλλον τέθηκε και ένα ερώτημα για την προσχώρηση Βουλγαρίας-Ρουμανίας στον χώρο Σέγγεν. Καταρχάς να ευχαριστήσω τις δύο χώρες αυτές για τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει για την εσωτερική ασφάλεια της Ένωσης. Γνωρίζετε όμως ότι οι θέσεις αυτές είναι αυτή τη στιγμή στο Συμβούλιο. Προβλέπετε ότι τον Οκτώβριο θα ξαναθέσουμε το θέμα αυτό ε, στην Μυρίσια Διάταξη, στο Συμβούλιο Κορυφής, στη Σύνοδο Κορυφής. Συγγνώμη, αλλά έχω ερωτήσει κάτι για το ξέπλυμα χρήματος, που είναι σημαντικό για την ασφάλεια των πολιτών και δεν άκουσα απάντηση. Α, ναι, συγγνώμη. Ερώτησε κάποιος τι θα κάνουμε ε, για την καταπολέμηση της ακροδεξιάς τρομοκρατίας. Εγώ καταρχά να πω ότι δεν, δεν διακρίνω, δεν θεωρώ ότι διακρίνεται η τρομοκρατία σε αριστερή και ακροδεξιά. Η τρομοκρατία είναι πλήγμα για όλο τον πληθυσμό μας και γι' αυτό όταν μιλάμε για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας μιλάμε για, για καταπολέμηση όλων των τρομοκρατικών απειλών. Όσον αφορά την νομοποίηση παράνομων εσόδων, πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα ιδιοκτικές αρχές θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα οι ιδιοκτικέ αρχές να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες ακόμη και ε, από τον τομέα ε, των χρηματοπιστωτικό. Γι' αυτό και θα κάνουμε κάθε προσπάθεια ε, και το, το, το εν λόγω έργο να το προχωρήσουμε και είμαι αισιοδόξη ότι θα καταφέρουμε να καταλήξουμε σε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. So many Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν πάρα πολλά τα ερωτήματα βεβαίως. Είναι δύσκολο κανείς να τα απαντήσει με τέτοια συντομία, αλλά ήταν μια καλή απόπειρα. Κοιτάξτε να δείτε, δεν ε, βρισκόμαστε εν έτη 2015 όπου ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι προετοιμασμένη για την εισρωή ε, και προσφύγων από τη Συρία αλλά και μεταναστών. Αυτό που πολλοί ανέφεραν με τον έναν τον άλλον τρόπο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να φέρει απτά αποτελέσματα προς τους πολίτες της. Ε, αποφάσεις που ε, θα είναι αποτελεσματικές, θα βασίζονται στις ε, αξίες μας και στις δεσμεύσεις που έχουμε κάνει και σε διεθνές επίπεδο. Και τώρα είναι η κατάλληλη χρονική στιγμή, γιατί σήμερα η εικόνα είναι πολύ διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν. Η εισρωή προς την Ιταλία περιορίστηκε χάρη σε μέτρα που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ιταλία κατά 80% σχεδόν. Το πρώτο εξάμεινο του 2018 μόνο 40.000 άτομα μπήκαν ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όχι 1,6 εκατομμύρια όπως το 2015. Και πράγματι πρέπει ε, να δουλέψουμε από κοινού. Βλέπετε ότι υπάρχουν ισχυρέ θέσεις ε, στο Κοινοβούλιο σε ορισμένα ζητήματα. Παρ' όλα αυτά θα συνεχιστεί ο διάλογος μεταξύ μας. Ελπίζουμε να έχει και καλά αποτελέσματα. Σα ευχαριστώ. Θα περάσουμε τώρα στο τελευταίο σημείο της ημέρης διάταξης, η θέσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας. The lead committee is uh, ample and... Καθήλυνα αρμόδια είναι η Επιτροπή Απασχόλησης ε, και η συγκητής ο κύριος Παύλ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ. Αρχικά θα ευχαριστήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πρόταση θέσπιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασία. Ησυχία παρακαλώ. Όσοι θέλουν να αποχωρήσουν, παρακαλώ ας αποχωρήσουν ησύχως για να ακούσουμε και τον εισηγητή. Συνέχιστε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είμαι μέλος της Επιτροπής ε, Απασχόλησης και έτσι είναι πολύ σημαντικό θεωρώ αυτό το ζήτημα και για τις δύο αυτές τις επιτροπές. Ε, η Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας θα πρέπει να συμβάλλει στην ε, ορθή εφαρμογή των συνθήκων εργασίας, εσφαλίζοντας την προστασία θεμελιδών δικαιωμάτων, όπως η ελεύθερη κυκλοφορία ατόμων και εργαζομένων και όσων έχουν ε, γαλάζια κάρτα, ε, των αποσπασμένων και όσων έχουν ε, άδεια παραμονής και των οικογενειών τους. Δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις, να δίνεται ίση πρόσβαση σε υπηρεσίες και δικαιώματα και να καταπολεμήσουμε τις ε, παράνομες δραστηριότητε. Για μένα ε, σημαντικό ζήτημα είναι η αδήλωτη εργασία, γι' αυτό έχω υποβάλει τροπολογία για την καταπολέμηση τη αδήλωτη εργασία, που συχνά έχει διασυνοριακή διάσταση και μπορεί να έχει σημαντικέ επιπτώσει για τους εργαζομένους. Κάποιε ευάλωτε ομάδε, όπω η υπήκοοι τρίτων χωρών, είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι στην αδηλωτή εργασία Ε, και συχνά πλήττονται τα δικαιώματά τους. Ε, θα πρέπει ο ΙΕΛΕ λοιπόν να ενισχύσει τη συνεργασία ε, για την καταπολέμηση της αδίλωτης εργασίας βάσει της απόφασης 344 του 2016 και να ενισχύσει περαιτέρω την συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για αυτό το τομέα. Για την προστασία προσωπικών δεδομένων και το σχετικό κανονισμό θα πρέπει φυσικά να τηρείται. Θέλω να διασφαλίσω ότι οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων θα περιορίζεται σε ό,τι είναι απαραίτητο και αναλογικό. Η συλλογή δεδομένων πρέπει να γίνεται για συγκεκριμένου και νόμιμου ε, σκοπού ε, και να μην υπάρχει διαφορετική επεξεργασία που δεν συνάδει με αυτού του σκοπού. Και προτείνω να διασαφίσουμε ότι η αρχή και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεωρηθούν κοινοί ε, κοινέ αρχέ ελέγχου για την επεξεργασία αυτών των δεδομένων. Τέλο, καταπολέμηση τη απάτη. Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το, τη θέσπιση του δημόσιου κατηγόρου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελία που συνδέεται με το έργο της Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας. Ευχαριστούμε τον κύριο Πάβελ. Ο Πρόεδρο ανακοινώνει ότι η διερμηνία θα σταματήσει στι 18.30. Οι σκιώδει ηγητέ θέλουν να πάρουν τον λόγο. Παρακαλώ, κύριε Ροκά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Εξ ονόματος του κυρίου Σούλκουρα από την ομάδα του ΕΛΚ, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το έργο σας, όχι μόνο για την κατάρτιση της έκθεσης, αλλά και για το πολύ θετικό κλίμα που υπήρχε. Και ο κύριος ε, Σόργορ ε, θα ακολουθήσει και, αυτό, και ο ίδιος αυτό το πνεύμα με τις ε, τροπολογίες του. Όμως ε, θα θέλαμε να ενισχύσουμε το κείμενο. Μία ομάδα τροπολογιών θα φορά την ελεύθερη ε, κυκλοφορία εργατικού δυναμικού. Είπα ότι θα πρέπει να τηρείται και να διευκολύνεται μέσω ευρωπαϊκών κανόνων που επιβάλλονται με απλό και αποτελεσματικό τρόπο. Η επιβολή των δίκαιων κανόνων αυτών αποτελούν εχέγγυο για την ύπαρξη λαϊκής υποστήριξης. Εάν δεν γίνουν σεβαστοί αυτοί οι κανόνες, ε, τότε απογοητεύουμε τους ευάλωτους πολίτες και επιχειρήσεις, αλλά υπάρχει κίνδυνος να χαθεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στην ενιαία αγορά και να δώσουμε έδαφος ε, στο λαϊκισμό ε, που θα ζητήσει περισσότερους περιορισμούς και τελικά θα απλήξει την ενιαία αγορά. Όπως αναγνωρίζει και η Επιτροπή, υπάρχουν προβληματισμοί σε ό,τι αφορά τους ε, εργαζόμενοι που αλλάζουν ε, χώρα, σε ό,τι αφορά τα δικαιώματά τους και για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αβέβαιο περιβάλλον με άνθρωπους όρους ανταγωνισμού. Επίσης, γίνεται μια ε, σε ορισμένα ζητήματα, γιατί υπάρχει μελέτη DPR που δείχνει τα εμπόδια ε, που έχουν να κάνουν με την ηλικία, ε, ε, ζητήματα επιδομάτων, ανεργίας, οικογενειακών επιδομάτων. Εμείς είμαστε κοντά και στην Αυστρία. Υπάρχουν πολλοί καταστηματάρχες που δουλεύουν εκεί και μπορώ και εγώ λοιπόν να μαρτυρήσω το ίδιο. Όπως αναφέρει επίσης ο κύριος Σουλγκόρ και εγώ ως Ρωμά μπορώ να σας πω ότι οι πήκοοι τρίτων χωρών και ιδιαίτερα η Ρωμά τυχάνουν χάνουν διακρίσεων όχι μόνο ε, για λόγους ε, υποβάθρου ή ηθαγένειας. Θα πρέπει να αξιοποιήσουμε όλα τα διαθέσιμα εργαλεία για την ε, εξάλληψη ανισοτήτων στην εφαρμογή του ευρωπαϊκού δικαίου, έμφαση να δοθεί και στην διακίνηση για εμπορία ανθρώπων Υπάρχει και έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που δείχνει και άλλες μορφές εκμετάλλευση σε οικονομικό επίπεδο, όχι μόνο στους εργαζόμενους, τους εργάτες στον τομέα της γεωργίας, αλλά και στην οικοδομή και σε άλλα επαγγέλματα χαμηλών δεξιοτήτων πολύ σημαντικό ως Όλγορ να ακολουθήσουμε ε, αυτή την ε, άγουσα που προτείνεται. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάτι άλλο. Κύριο κύριος Πάβελ, παρακαλώ. Και εγώ ζω στα σύνορα. 8 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουγγαρία και γνωρίζω και εγώ τα ζητήματα. Τέλεια. Τα γνωρίζετε λοιπόν και οι δύο. Προθεσμή υποβολή ε, τροπολογιών η 16 Ιουλίου, 4 το απόγευμα. Για ποιον θέλει να υποβάλει τροπολογίες, νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο τέλος της σα διάταξης για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.